Συνάδελφοι, πριν επαναλάβουμε τη σύνοδο, θα ήθελα να αποτίσουμε φορό τιμή στα θύματα των επιθέσεων της περασμένης Δευτέρα στην Ουτρέχτη, στην Ολλανδία. Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες ήταν ο απολογισμός. Έχω εξφράσει τα συλληπιτήριά μας στον Πρωθυπουργό της ε, Ολλανδία. τον κύριο Ρούτε, και σήμερα θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου σε όλους του συναδέλφου μου εδώ στην Ολομέλεια και κυρίως προς τον Ολλανδό, Ολλανδικό λαό και τα, θύματα των, τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων. Θλιβερό γεγονό. Δεν μπορούμε παρά να αφορά φορό τιμή και στα θύματα του Κρίστσετ στην ε, Νέα Ζηλανδία. Μια επίθεση που κόστησε τη ζωή 50 ανθρώπων. Δολοφονήθηκαν ε, φρικτά ενώ είχαν ε, προσέλθει για να προσευχηθούν σε δύο τζαμιά. Τα δύο αυτά περιστατικά μας υπενθυμίζουν ξανά ότι πρέπει να μην σταματήσουμε να προσπαθούμε να αμυνθούμε κατά του φιλετικού μίσους. Θα πρέπει όλες αυτές τις βάβαρε πράξεις, κάθε μορφή βία και φυλετική διάκριση να την καταπολεμήσουμε με πυγμή. Επίσης θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στα θύματα του τυφώνα που χτύπησε στο Μαλάουι, τη Μοζαμβίκη και τη Ζιμπάμπουε. Με πολλά θύματα και τρομερές καταστροφές. Επίσης, να θυμίσουμε και τις ε, ε μεταφορές ε, χιλιάδων ε, πολιτών από τις χώρες της Βαλτικής 21 Μαρτίου 1939 που ήταν η αρχή των επιθέσεων στις χώρες αυτές και που θεωρούνται κλίματα κατά της ανθρωπότητας όπως και τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να θυμηθούμε όλα τα αθώα θύματα και γι' αυτό το λόγο όπω ζητήθηκε και από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, να, τηρήσουμε ενό λεπτού σιγή για τα θύματα όλων αυτών των περιστατικών. Σας ευχαριστώ. Κυρίσω την επανάληψη των, της Συνόδου που διακόπηκε στις 14 Μαρτίου. Τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης έχουν διανεμηθεί. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρούμε ότι είναι εγκεκριμένα αυτά. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Πέζος του Amazon να διαγράψει τα στοιχεία της Amazon ε, του Billiot. Θα πρέπει ό,τι αναφέρεται στο Billiot να διαγραφεί από το Amazon. Θα πρέπει να θεωρηθεί ε, απολυταρχική και ναζιστική καταπίεση αυτή των Σοβιέτ. Ε, σας παρακαλώ, Πρόεδρε, ο ευρωπαϊκός λαός πρέπει να γνωρίζει την αλήθεια την αλήθεια της σοβιετικής καταπίεσης. Ρώτησαν αν υπήρχαν παρατηρήσεις για τα πρακτικά. Εάν δεν υπάρχουν, θεωρείται εγκεκριμένα, θεωρείται εγκεκριμένα τα πρακτικά. Συμφωνώ με τις καταγγελίες και τις ανησυχίες που εκφράζεται και αν χρειαστεί θα παρέμβουμε. Ο κύριος Μποργκέτσιο, ευρωβουλευτής, μου ζήτησε να καλύψουμε τα, την εντολή ε, και την ασυλία του στα πλαίσια μιας δικαστικής διαδικασίας τα, από την πλευρά της εισαγγελία της Ιμπέρια. Βάσει του κανονισμού, η αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου αναλαμβάνει το θέμα. Παρόμοια ε, σύσταση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την ε, Διαγωγή των Βουλευτών ε, έχει, έχει φτάσει στα χέρια μου και αποφασίζω να επιβάλλω κύρωση εις βάρος του κυρίου Μάρκος Πρετσέλ για έλλειψη σεβασμού στις ε, υποχρεώσεις του βάσει του κώδικα συμπεριφοράς. Η κύρωση είναι απλώς μια προειδοποίηση. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και από τον ενδιαφερόμενο στις 22 Μαρτίου. Βάσει του άρθρου 167 του κανονισμού, ο κύριος Πρετσέλ έχει δύο εβδομάδες διάθεσή του για, από την στιγμή της κοινοποίηση τη κύρωσης για να ε, προσφύγει εσωτερικά ε, κατά τη απόφαση του Προεδρείου. Επιτροπή ΕΝΒΗ έχει αποστείλει δύο διορθωτικά για κείμενα που έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 231.4. Τα διορθωτικά αυτά θα θεωρηθούν εγκεκριμένα εκτό και αν εντό 24 ωρών από τη στιγμή τη κοινοποίησή του, μια πολιτική ομάδα, ένα ικανό αριθμό ε, βουλευτών που είναι ε, ίσω με, με το ελάχιστο όριο, δεν ζητήσουν ψηφοφορία. Τα διορθωτικά διατίθενται στον ιστότοπο τη Ολομέλεια και οι τίτλοι του θα δημοσιευτούν στα πρακτικά τη τρέχουσα Ολομέλεια να ενημερώσω την Προεδρία του. Σήμερα, μαζί με τον Πρόεδρο του Συνοβουλίου, θα υπογράψουμε 13 νομοθετικέ πράξει βάσει τη ε, κλασική νομοθετική διαδικασία, βάσει του άρθρου 28 του ε, Κοινοβουλίου. Οι τίτλοι θα δημοσιευτούν στα πρακτικά τη τρέχουσα συνόδου. Τώρα περνάμε στην διάταξη των εργασιών ε, η ημερήσια διάταξη που έχει εγκριθεί στι 21 Μαρτίου από τη διάσκεψη των Προέδρων βάσει του άρθρου 49 έχει μοιραστεί. Σε ό,τι αφορά την Δευτέρα, η ομάδα Άλντε ζήτησε η, συζήτηση για την προφορική ερώτηση κατάσταση του κράτου δικαίου και καταπολέμηση τη διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω στη Μάλτα και τη Σλοβακία, να ολοκληρωθεί με ένα ψήφισμα τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που θα ψηφιστεί την Πέμπτη. Δίνω το λόγο στην κυρία Ιντβελτ για να παρουσιάσει το αίτημα αυτό τη ομάδα Άλντε. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι θα συζητήσουμε αργότερα την προφορική ερώτηση που αναφέρατε. Αρχικά η ψηφοφορία θα γινόταν την Πέμπτη. Ε, νομίζω ότι πρέπει να γίνει η συζήτηση και να ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία όμως, να μην είναι χωριστά. Ευχαριστώ. Η κυρία Σμόλκοβα για μια παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ να ρωτήσω τους συναδέλφους αν μπορεί η ψηφοφορία να ε, γίνει την επόμενη εβδομάδα. Γιατί στη Σλοβακία έχουμε γύρω εκλογών το Σάββατο και θα ήθελα να μην ε, έχουμε και αυτή την πρόταση στα πόδια μας ε, που μπορεί να επηρεάσει πριν από τις ευρωεκλογές. Φοβάμαι ότι θα επηρεαστεί η προεκλογική εκστρατεία. Δεν μπορεί λοιπόν να πάει για την επόμενη εβδομάδα. Κυρία Ίνφελτ. Ξέρω για τις εκλογές, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να σιωπούμε, οπότε υπάρχουν εκλογές. Όπως είπατε, σύντομα έχουμε και τις ευρωεκλογές. Δηλαδή τι, δεν θα μιλάμε σε καμία χώρα μέχρι τις ευρωεκλογέ πια. Ή το ψήφισμα είναι ισορροπημένο, αντικειμενικό και δεν καταλαβαίνω πώς θα επηρεάσει αρνητικά τις εκλογές. Δεν υπάρχει κανένα ρίσκο. Ε, είναι εν μέρει επικριτικό το ψήφισμα, αλλά λέει και ότι έχει επιτελεστεί πρόοδος στις δύο αναφερόμενες χώρες, οπότε δεν υπάρχει κανένα κίνδυνος. Το θέμα δεν είναι πολιτικό. Το ψήφισμα έχει ήδη ψηφιστεί στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών στην Σλοβακία, οπότε δεν νομίζω να υπάρχει κανένας φόβος, κίνδυνος και δεν πρέπει να πολιτικοποιούμε τα θέματα αυτά βγάζοντάς τα από την ημερήσια διάταξη. Να μείνει, να ψηφιστεί την Πέμπτη, το κράτος δικαίου δεν αφορά ένα κράτος μέλος ε, μόνο ή ορισμένα, αλλά είναι ένα καθολικό ζήτημα. Κυρία Σμόλκοβα, και μετά ψηφίζουμε. Δεν θέλω να ε, βγει από το πρόγραμμα, απλώς θέλω να πάει, να πάει την επόμενη εβδομάδα η ψηφοφορία. Δεν ζείτε εσείς στη Σλοβακία, συνάδελφοι. Εμείς θέλουμε να δράσουμε καλή την πίστη. Γι' αυτό σας απευθύνω αυτή την έκκληση να πάει την επόμενη εβδομάδα η ψηφοφορία. Μου φαίνεται ότι οι φιλελεύθεροι δεν θέλουν να γίνει αυτή η συζήτηση και να αναβληθεί η ψηφοφορία. Οπότε ας ψηφίσουμε το αίτημα και θα αποφασίσει η ίδια η Ολομέλεια. Θα ψηφίσουμε για το κατά πόσον, όπως προτείνουν οι φιλελεύθεροι, θα γίνει συζήτηση για την προφορική ερώτηση και θα υπάρξει και ψήφισμα την Πέμπτη ε, ποιοι είναι υπέρ της πρότασης των φιλελευθέρων της Άλντε. Κατά. Ας κάνουμε και έναν ηλεκτρονικό έλεγχο. Avete votato άπαντες. Η ψηφοφορία έληξε. Εγκρίνεται η πρόταση. Η συζήτηση για την προφορική ερώτηση σχετικά με την κατάσταση του κράτου δικαίου και την καταπολέμηση τη διαφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στην Μάλτα και τη Σλοβακία, θα ολοκληρωθεί με ε, ψήφισμα τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που θα ψηφιστεί την Πέμπτη. Για την Τρίτη, βάσει του άρθρου 113 παράγραφο 6. Α, για τη Δευτέρα πάλι. Για την τρίτη, βάσει του άρθρου 113.6, ε, οι ομάδε ENF και GUE ε έχουν υποβάλει αντίρρηση στην έκθεση τη συναδέλφου Βότμαν για την απόφαση ίδρυση ε, μια Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση για την Ειρήνη. Η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι την Τρίτη στην μία το μεσημέρι και η ψηφορία θα γίνει την Πέμπτη. Προτείνω η συζήτηση να γίνει την Τετάρτη το απόγευμα και να είναι το τελευταίο σημείο τη Συνόδου. Υπάρχουν αντιρρήσει. Ωραία, εγκρίνεται αυτή η αλλαγή. Και πάλι για την Τρίτη. Η ομάδα ΕΝΕΦ ζήτησε από το Συμβούλιο και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δηλώσει ω δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη για την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου που καταργεί ακυρώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, της 23 Δεκεμβρίου 2015 σε σχέση με τις κρατικές βοήθειες που δόθηκαν από την Ιταλία στην τράπεζα Τέρκας. Κατά συνέπεια, η Σύνοδο θα ξεκινήσει στι 8.30. Ο λόγος στον κύριο Τζάνι για να παρουσιάσει το αίτημα της ομάδας του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ε, εξηγήσατε, θα θέλαμε επί, του θέματος αυτού και τις αποφάσεις που ελήφθησαν υπήρχαν ολέθριες συνέπειες σε σχέση με τις αποταμιεύσεις οι οποίες κατέρευσαν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που αναμένουν μία απάντηση μετά από τέσσερα χρόνια αφού υπέστησαν τις ολέθριες συνέπειες της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία ε, ακύρωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λίγες μέρες πριν. Θέλουμε λοιπόν μία απάντηση και να γίνει μία αντιπαράθεση για να δούμε πού ε, βρίσκονται οι ευθύνε αυτής της ε, κατάρρευσης. Θα ήθελα να γίνει και ονομαστική ψηφοφορία. Θέλει κάποιος να προβάλλει αντίρρηση στην πρόταση της ομάδας ΕΝΕΦ. Περνάμε στην ψηφοφορία. Το αίτημα είναι να ε, προβλεφθεί συζήτηση που θα ξεκινήσει στις 8.30 την Τρίτη για την απόφαση του δικαστηρίου που ακυρώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2015 σε σχέση με την κρατική βοήθεια που δόθηκε από την Ιταλία υπέρ της τράπεζας Τέρκας. Η ψηφοφορία ξεκινάει τώρα. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται η πρόταση. Τετάρτη τώρα. Προηγουμένως ε, μια ενημέρωση. Κατάλαβα, κατάλαβα. Επειδή θα τάξουν τίποτα και για το πακέτο τη κινητικότητα πριν τα αιτήματα αυτά, θέλω να σα ενημερώσω ότι βάσει τη απόφαση τη διάσκεψη του Προέδρου να οριστεί προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στη μία το μεσημέρι τη περασμένη Παρασκευή, οι υπηρεσίε τη Ολομέλεια, οι νομικοί προγνώμονε και οι μετάφραστε ε, εργάστηκαν νυχθημερών όλο το Σαββατοκύριακο για να μπορέσουν να δημοσιευτούν περίπου χίλιε τροπολογίε και να ετοιμαστεί η ψηφοφορία. Σα ενημερώνω ότι όλε οι τροπολογίε έχουν διατεθεί στον ιστότοπο ή μάλλον θα διατεθούν μέχρι τις 17.30 σήμερα, τουλάχιστον στα αγγλικά. Οι υπόλοιπε γλώσσες θα είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του αυριανού απογεύματος. Η ε, κατάλογη ψηφοφοριών θα είναι διαθέσιμη ήδη απόψε. Παρακαλώ. Κύριε Εκχάουτ. Ευχαριστώ. Πρόκειται για την ψηφοφορία της Τρίτης, για την απαλλαγή, ιδιαίτερα για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν μερικές τροπολογίες που έχουν υποβάλει οι σοσιαλιστές για την θέση, για μια συγκεκριμένη θέση της Επιτροπής. Θεωρήσατε ότι μία πρόταση είναι παραδεκτή, μία άλλη όμως που αφορά τις συνέπειες της θέσης του κυρίου Σέλμαϊερ είναι απαράδεκτη. Αυτό είπατε. το άρθρο 170 αναφέρεται σε αυτό. Αν κάτι θεωρείται μη παραδεκτό, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Είναι πολιτική απόφαση που επαφίεται στο σώμα. Θα ήθελα να ανακαλέσετε την απόφασή σας να μην θεωρηθεί μη παραδεκτή η τροπολογία και να αφήσετε το σώμα να ψηφίσει αύριο. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα Σελμάγερ, ζήτησα από τι ερευνητέ τη Ολομέλεια να ελέγξουν το μη παραδεκτό ή όχι τη τοπολογία. Η απάντηση που δέχτηκα και την οποία συμμερίζομαι με οδήγησαν να θεωρήσω ότι δεν είναι παραδεκτή η τροπολογία που ζητά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής είναι έτοιμα πολιτικού χαρακτήρα. Από τους συντάκτες της τροπολογίας. Η κυρίαρχη ολομέλεια θα αποφασίσει τι πρέπει να γίνει. Η άλλη τροπολογία όμως συνέδε αυτομάτως την αυτοκτονία μιας καημένης υπαλλήλου σε αυτήν αναφέρεστε. Πείτε μου. Ναι, υπήρχε κι άλλη μια τροπολογία σε σχέση με την αυτοκτονία που θεωρήθηκε μη παραδεκτή. Δεν αναφέρομαι σε αυτή γιατί κατανοώ γιατί είναι μη παραδεκτή. Αναφέρομαι σε μια τροπολογία στην παράγραφο 258 Δέλτα, όπου η τροπολογία λέει, λαμβάνοντας υπόψη σοβαρότητα της κατάστασης σε σχέση με την απαλλαγή το 2016, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει τη στάση της σε σχέση με το συγκεκριμένο τμήμα. Δηλαδή αφορά το συγκεκριμένο τμήμα και πρόκειται για μια πολιτική απόφαση που θα πρέπει να αφήσουμε στην Ολομέλεια και νομίζω ότι απαντήσατε ήδη εσείς γιατί πρέπει να αφαιθεί στο σώμα και νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό. Η τροπολογία στην οποία αναφέρεστε συνδέεται άμεσα με την ε, επόμενη τροπολογία. Γι' αυτό όταν ζήτησα από τι υπηρεσίε να το ελέγξω, μου είπαν ότι κατά τη δική του άποψη είναι μη παραδεκτή, γι' αυτό το θεώρησα και εγώ μη παραδεκτή. Τώρα για την πολιτική ψηφοφορία, για το πολιτικό ζήτημα, την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα, θα τοποθετηθεί η ίδια η Ολομέλεια. Σε ό,τι αφορά την Τετάρτη, μια ομάδα βουλευτών που θα πρέπει να φτάνουν στο ελάχιστο όριο από του συντηρικού και μεταρρυθμιστέ και την EFTD ζήτησαν τη συζήτηση και την ψηφοφορία για το πακέτο τη κινητικότητα που περιλαμβάνει τρει εκθέσει, Ερτου, Κιλόνεν και Βάντεν Κάμπ να αφαιρεθούν από την ημερήσια διάταξη. Δίνω το λόγο στον κύριο Νόβακοφ για να παρουσιάσει το αίτημα εκ μέρους του ικανού αριθμού βουλευτών που φτάνουν στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο. Δεν είστε κύριε Νόβακοφ στην αίθουσα. Α, ωραία. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, στο τέλος της τρέχουσας θητείας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει ένα σοβαρό σφάλμα, δηλαδή θα αφήσει ένα πακέτο που απορρίφθηκε τρεις φορές να ψηφιστεί μια τέταρτη φορά χωρίς κανένα συμβιβασμό. Δηλαδή είναι σαν να ρίχτεται τα ζάρια. Υπάρχουν 1.600 τροπολογίες. Αυτό θα οδηγήσει σε πλήρη σύγχυση. Παρακαλώ ψηφίστε το αίτημά μας για να σώσετε τη ζωή πολλών Ευρωπαίων. Εκ μέρους των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, παρακαλώ. Komisja Transportu rozpatrywała e, pakiet mobilności. Αυτό που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σε σχέση με το πακέτο κινητικότητας είναι ότι η Επιτροπή Μεταφορών συμφώνησε, αλλά το Κοινοβούλιο απέρριψε τη συμφωνία. Σήμερα δύο από τις τρεις εκθέσεις, για δύο από τις τρεις εκθέσεις δεν υπάρχει συμφωνία. Και καμία τροπολογία δεν εγκρίθηκε από την Επιτροπή Μεταφορών. Θα πρέπει να αποφασίζουμε για τις 1.600 τροπολογίες εδώ με τα μέλη που γνωρίζουν γενικά για αυτό το θέμα. Υποστηρίζω λοιπόν οι εκθέσεις Βαντεκάμπ και Κιλόνεν, οι δύο δηλαδή εκθέσεις οι οποίες δεν εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Μεταφορών, να μην ε, εξεταστούν. Ο λόγος των εισηγητή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι είναι εντελώ λανθασμένο αυτό ο τρόπο. Διότι έχουμε εργαστεί εδώ και δύο χρόνια περίπου για το θέμα αυτό, για το πακέτο κινητικότητα 1. Έχουμε βρει τι κατάλληλε συμβαστικέ λύσει ε, και σε συνεννόηση με ολόκληρο το Κοινοβούλιο, προκειμένου να αποφύγουμε την θλιβερή κατάσταση που θα προκύψει στου αυτοκινητοδρόμου τη Ευρώπη. Ε, και δεν, ε, αν δεν έχουμε νομική βεβαιότητα, θα πρέπει να ψηφίσουμε στη διάρκεια αυτή τη θητεία και αυτή την εβδομάδα εδώ στο Στρασβούργο. Βρήκαμε την δέουσα λύση. Θέλω να επαναλάβω ότι δεν υπάρχει ανάγκη να ε, μην γίνει ψηφοφορία. Απλώ ε, είναι πολιτικέ οι σκοπιμότητε όσων θέλουν να μην γίνει ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Σα ε, παροτρύνω λοιπόν να ψηφίσουμε αυτήν την εβδομάδα για το πακέτο κινητικότητα παριθμών 1. Ωραία λοιπόν, α ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε για την πρόταση της ε, ομάδας βουλευτών που είναι ίση με το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο ECR και EFTD που ζητούν η συζήτηση και η ψηφοφορία για το πακέτο κινητικότητα να αφαιρεθούν από την ημερήσια διάταξη. Άρχε, θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία, με ονομαστική δηλαδή κλίση, άρχεται αυτή. Πέρας. Η πρόταση απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. Η ημερήσια διάταξη παραμένει ως έχει. Και πάλι για την Τετάρτη. Η ομάδα του ΕΛΚ έχει Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, αποφασίσατε να προβλέψετε στην εμείς διάταξη το πακέτο κινητικότητας. Να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής. Πάνω από χίλιες τροπολογίες δεν έχουν μεταφραστεί. Ναι, ναι, το ξέρω. Το ψηφίσατε και θα σεβαστούμε την επιλογή που κάνατε. Ωστόσο, Τώρα ο καθένας καλείται να αναλάβει τις ευθύνες του. Σήμερα οφείλουμε να δείξουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι. Και υπεύθυνοι τι θα πει θα πει ότι θα πρέπει να προσφέρουμε κοινωνική συνοχή σε όλους μας τους εργαζομένους, ιδίως αυτούς που εργάζονται στις οδικές μεταφορές. Εσείς λοιπόν να μην κάνετε αυτό που κάνατε και την περασμένη φορά, να προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε ως εργαλείο το κείμενο αυτό για πολιτικές σκοπιμότητες, διότι εν τέλει θα καταλήξουμε να μην έχουμε κείμενο. Ευχαριστώ. Κύριε Γκουόγκα. Η λιθουανική αντιπροσωπεία δεν είναι εδώ. Θα ψήφιζαν όλοι υπέρ τη αναβολή τη ψηφοφορία. Είναι εντελώ άδικο. Είναι άδικο. Έπρεπε να αναβληθεί η ψηφοφορία. Και να το γνωρίζετε. Η Λιθουανία, μια από τι μικρότερε χώρε τη Ευρώπη, θα πληγεί από όλα αυτά. Σα παρακαλώ, Πρόεδρε. Σα παρακαλώ, σκεφτείτε και τι μικρέ χώρε. Στηρίζουμε την ευρωπαϊκή πορεία. Αγωνιζόμαστε για τον ευρωπαϊκό σκοπό. Μας καταστρέφετε με αυτή την τροπολογία. Καταγράψτε το. Κύριε Γκόγκα, η Ολομέλεια αποφασίζει και είναι υπεύθυνη για τι αποφάσει τη. Έχω ενημερώσει και για το πρόβλημα τη μετάφραση. Έχω πει πω θα λυθεί. Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει ψήφισε μάλλον με ονομαστική κλίση και τελικά η Ολομέλεια αποφασίζει τι πρέπει να πραχθεί. Την Τετάρτη η ομάδα του ΕΛΚ έχει ζητήσει να προσθεθεί το απόγευμα δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις απειλές κατά της ασφαλείας που προκύπτουν από την ε, ταχεία διάδοση του τρομοκρατικού περιεχομένου επιγραμμικός στο διαδίκτυο. Θέλει κάποιος να παρουσιάσει το αίτημα, κυρία Μετσόλα. Το ΕΛΚ θα ήθελε να ζητήσει μια δήλωση επιτροπής για τις ε, απειλές ε, λόγω της διάδοσης ε, τρομοκρατικού περιεχομένου. Επιγραμμικά είδαμε τι έγινε στη Νέα Ζηλανδία και την Ουτρέχτη και ακριβώς επειδή μπορούσαν να τα παρακολουθήσουν όλοι, γνωρίζουμε ότι ο χώρος μας online χρησιμοποιείται από εξτρεμιστές για ρητορική μίσους, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να επιτρέψουμε. Ο επιγραμμικός χώρος θα πρέπει να καταστεί ασφαλής, γιατί θα πρέπει να αποσυρθεί αυτό το περιεχόμενο σε σχέση με τρομοκρατικές ομάδες ή με μονομένα άτομα. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Ξέρω ότι υπάρχει μια νομοθετική διαδικασία, θα πρέπει αυτή τη βδομάδα να αποστείλουμε ένα στεναρό πολιτικό μήνυμα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αμελήσουμε. Το λόγο ζήτησε ο κύριος Ντάλτον για να μιλήσει κατά της πρότασης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η επίθεση του Christ Church μας δείχνει ότι πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Το ζήτημα είναι πώς. Εγώ είμαι συντάκτης αυτού του θέματος. Η Επιτροπή έχει κάνει μια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου που διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε συνδυασμούς, έχουμε συνάντηση σκιωδών, και το ζήτημα θα συζητηθεί στη Λίμπε την επόμενη εβδομάδα και στην Ολομέλεια τον επόμενο μήνυμα μήνα. Άρα μπορείτε να το συζητήσετε τον επόμενο μήνα. Αυτή είναι η κοινοβουλευτική διαδικασία και πρέπει να την ακολουθήσουμε. Δεν έχει νόημα να κάνει ανακοίνωση η Επιτροπή όταν είμαστε εν μέσω διαπραγματεύσεων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Δέχομαι τη θεωρία αυτών που λέει το ΕΛΚ, αλλά νομίζω πρέπει να απορρίψουμε το αίτημα. Ωραία. Να ψηφίσουμε λοιπόν για αυτό το αίτημα τη ομάδα του ΕΛ και να προσθέσουμε την Τετάρτη το απόγευμα δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι απειλέ κατά τη ασφαλεία που προκύπτουν από ταχεία διάδοση του τρομοκρατικού περιεχομένου επιδομικώ. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Θέλετε να γίνει έλεγχο. Α ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται η πρόταση. Η ημερήσια διάταξη έχει πλέον εγκριθεί. Οπότε περνάμε στα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Πρώτο, έκθεση Κόφοντ και Νίντερμαϊερ σε σχέση με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Uh, uh, Συνεχίζουμε τώρα. Επόμενο και πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Έκθεση Κόφο και Νίτερ Μάγερ για το οικονομικό έγκλημα φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Συνάδελφοι, όσοι δεν θα συμμετάσχουν στη συζήτηση, παρακαλώ εγκαταλείψτε την αίθουσα ήρεμα για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Κόφον, τέσσερα λεπτά ως εισηγητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητέ επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τι έχουμε να αποφασίσουμε αύριο. Το πιο ολοκληρωμένο έργο του Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση φόρο διαφυγής, και οικονομικού εγκλήματος. Και Όλοι γνωρίζουμε ότι αν πάρουμε τη φοροαποφυγή για παράδειγμα και φοροδιαφυγή, συγγνώμη, είναι ασέβεια προς το πρόσωπό σας η φασαρία αυτή. Η συζήτηση επαναλαμβάνω να γίνει έξω ε, από την αίθουσα αυτή όταν δεν αφορά το θέμα. Παρακαλώ, ε, αποχωρήστε από την αίθουσα αν δεν θα συμμετάσχετε στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Συγγνώμη κύριε Κόφον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να τα ξαναπώ από την αρχή. Αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ολοκληρώθηκαν πολλά χρόνια δουλειά του Κοινοβουλίου ε, στο θέμα οικονομικών εγκλημάτων, φοροποφυγής, φοροδιαφυγής. Τώρα έχουμε το πιο ολοκληρωμένο έργο που έγινε από το Κοινοβούλιο αυτό στους τομείς καταπολέμησης ε, φοροδιαφυγής, φοροποφυγής, οικονομικού εγκλήματος. Πάρτε τη φοροδιαφυγή και τη φοροποφυγή. Στοιχίζει περίπου 1-3 ευρώ το χρόνο. 2.000 ευρώ ανά Ευρωπαίο πολίτη ανά χρόνο. Χρήματα που πρέπει να πάνε στα σχολεία, στα νοσοκομεία, να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν χρήματα για τους ευάλωτους και τους αδύναμους. Η κλοπή των φόρων γίνεται από, τους πιο ευάλωτους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά. Προσελκύουμε πολλές επιχειρήσεις και κεφάλαια. Ταυτόχρονα όμως δεν είμαστε αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση του ξεπλήματος ε, και της φοροδιαφυγής. Έρχονται πολλά χρήματα αλλά πολλές φορές δεν υπάρχει η σωστή επιβολή του νόμου, ούτε εφαρμόζονται κυρώσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες που δεν συνεργάζονται. Στην Danske Bank είναι ένα παράδειγμα. Έφευγαν χρήματα στην Εστονία περίπου 200 δις ευρώ που το τα ξέπλαιναν στην ενιαία αγορά μας οι Ρώσοι ολιγάρχες. Πρέπει να θωρακιστούμε. Και έχουμε πολλές καλές συστάσεις θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική, ελάχιστη εταιρική φορολόγηση, ε, να υπάρχει εναρμόνιση. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να σταματήσουν οι επιζήμιες ε, φορολογικές πρακτικές ε, διασυνοριακά για το ξέπλυμα χρήματος. Θέλουμε μια ε, συγκεντρωτική διαδικασία μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, γιατί σήμερα είναι πολύ εύκολο να έρχεται το βρώμικο χρήμα να ξεπλένεται και να διαχέεται σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι απειλή για την ε, χρηματοπιστωτική μας σταθερότητα, τη δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ε, μια αστυνομία για παράδειγμα χρηματοπιστωτική που θα μπορεί να παρακολουθεί ε, τις ε, συναλλαγές. Υπάρχει θέμα εφαρμογή όλων αυτών επίσης. Στις μεγάλες ε, επιχειρήσεις ε, οι γίγαντες κάνουν καλές δουλειές, χρησιμοποιούν, ε, δημιουργούν μεγάλη αξία, αλλά δεν πληρώνουν τους ανάλογους φόρους. Θα πρέπει να γίνει αυτό με την ανάλογη νομοθεσία. Χρειάζεται κοινή ενοποιημένη βάση επιχειρήσεων. Χρειάζονται οι εκθέσεις αναχώρα όταν πρόκειται για εταιρικούς φόρους για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι φέρονται υπεύθυνα και κοινωνικά ορθά. Θα πρέπει να εφαρμόζουν τα πρότυπα που υπάρχουν. Είναι μεγάλο βήμα μπροστά το ότι το Κοινοβούλιο, τα τρία και τα υπόλοιπα δύο θεσμικά όργανα έλαβαν για να υπάρχουν ε, ε, φορολογικές αρχές για τις επιχειρήσεις. Ε, πρέπει να σταματήσει επίσης και ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός που βλάπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες τις χώρες. Ε, ε, έχουμε μια καλή ολοκληρωμένη έκθεση, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά και στο μέλλον. Γι' αυτό ζητώ περισσότερο μόνιμες δομές ε, για να αντιμετωπιστούν τα θέματα φορολογίας και οικονομικού εγκλήματος. Θα συνεχίσουμε το έργο μας Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και τώρα ευχαριστώ κύριε Κοφόντο, δεύτερο συγκητής, ο κύριος Σνίντερ Μάγερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω έχω τέσσερα και δύο λεπτά αν δεν κάνω λάθος. Η έκθεση ολοκληρώνει το έργο της ειδική Επιτροπής και καλύπτει 300 τροπολογίες που κλείνουν παραθυράκια στην ομοθεσία που καλύπτει φοροδιαφυγή κλπ και προτείνει νέες λύσεις λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα σκάνδαλα και πορίσματα. Δεν συζητά μόνο το ξέπλυμα χρήματος ε, και τις φορολογικές απάτες αλλά και προβλήματα που αφορούν την ψηφιοποίηση φαίνεται ότι τα φορολογικά συστήματα δεν ε, ε, λύνουν τα προβλήματα και έχουμε μεγάλα προβλήματα στην ίσπραξη των φόρων. Επίσης εξετάζομαι τις ε, προηγούμενες αποκαλύψεις των Επιτροπών ΤΑΞ και ΤΑΞ 2. αυτό το καλύπτει η έκθεση σε σχέση με την αυξημένη διαφάνεια της εταιρική φορολογίας. Από την πρώτη πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πολλά άλλαξαν. Ε, ε, βελτιώθηκε η διαφάνεια, η δικαιοσύνη στη φορολόγηση, απλούστευση των φορολογικών καθεστώτων, ε, βελτιωμένη συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών δηλαδή μεταξύ κρατών μελών και άλλες, άλλους, άλλοι τομείς συνεργασίας. Ε, δεν μιλώ μόνο για τις πρωτοβουλίες που εισάγουν νέου παγκόσμια πρότυπα, αλλά υπάρχουν και βελτιώσεις στην ψηφιακή φορολόγηση. Έτσι βλέπουμε βελτίωση στην διαφάνεια της φορολογίας παντού στον κόσμο, αλλά θα πρέπει να πιέσουμε για να βρούμε καλούς τρόπους εξυγχρονισμού και ενίσχυσης των φορολογικών συστημάτων ώστε να διασφαλίσουμε τη σωστή εισπραξή των φόρων. Επίσης πρέπει να βεβαιωθούμε ότι εκείνοι που πληρώνουν σωστά αυτό που πρέπει δεν θα επιβαρύνονται υπερβολικά. Αναφέρομαι κυρίως στις ΜΜΕ, η ίσπραξη των φόρων καθ' αυτή ε, δεν είναι δαπανήρη και αναποτελεσματική. Μεγάλες αλλαγές συσχετίζονται και με τη βελτίωση ε, και το μεγαλύτερο ρόλο της ψηφιακής φορολόγησης. Πρέπει να βρούμε καινούριο τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τα νέα αυτά δεδομένα στην οικονομία. Είναι κρίμα διότι το Συμβούλιο δεν μπορεί να προχωρήσει με κέρυες πρωτοβουλίες εδώ, λαμβάνοντας υπόψη την κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για επιχείρησης την ψηφιακή ε, ε, φορολογία. Ελπίζω να παίξουμε ρόλο στην παγκόσμια οικονομία συμβάλλοντας στην εξέβρεση καλής λύσης ε, στα μεταβαλλόμενα δεδομένα. Επίσης, η TAX 3 και η σχετική έκθεση είναι καλός τρόπος για να βρεθεί συμφωνία ε, μεταξύ όλων των ε, χωρών. Είναι καλό που συμφωνούμε. Βεβαίως, δεν μπορεί να είμαστε σύμφωνοι σε όλα. Πρέπει να πω ότι εγώ πιστεύω σε κοινέ λύσεις όταν δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις σε επίπεδο μεμονωμένων κρατών μελών και κυβερνήσεων. Πιστεύω ότι μεγάλο κομμάτι της φορολογίας αποτελεί αρμοδιότητα αποκλειστική των κρατών μελών και πρέπει να την σεβόμεθα ιδιαίτερα όταν ε, μιλάμε για ε, τον ε, ελάχιστο αποτελεσματικό αποδοτικό φορολογικό συντελεστή. Είμαι υπέρ τη συνεργασία, αλλά δεν συμφωνώ με την πρόταση κάποιων μελών του να έχουμε 18% ε, ελάχιστο ε, συντελεστή. Νομίζω ότι ε, πρέπει να παραμείνουν πολλά θέματα στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όμως μπορούμε να βρούμε σε άλλα θέματα κοινό έδαφος. Μετά την συνεργασία που έγινε ε, υπάρχει ε, ε, ορισμός φορολογικών αρχών, έχουν αξιολογηθεί ε, νέες απειλές όπως επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός και νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Επίσης εκτιμώ ιδιαίτερα όλοι νομίζω την βελτιωμένη διαφάνεια στο έργο του Συμβουλίου, ιδιαίτερα στο φως των αλλαγών, στην συμπεριφορά, στην ομάδα δεοντολογίας και νομίζω ότι τα μέλη του Συμβουλίου θα κινηθούν προς τα μπρος σε σημαντικά θέματα που θα βελτιώσουν τη λειτουργικότητα της ε, ενιαίας αγοράς. Ε, επίσης, στην Επιτροπή ε, τάξη ε, ασχοληθήκαμε με πολλά θέματα ξεπλήματος χρήματος. Λυπούμε που η Κομισιόν έπρεπε να κινήσει διαδικασία επί παραβάση, επειδή κανένα κράτος μέλος δεν μετέφερε στην Εθνική Νομοθεσία ε, τη σχετική οδηγία για το ξέπλυμα. Αυτό χρειάζεται με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόζεται σωστά. Και εκεί δεν κινούμεθα αρκετά γρήγορα υπάρχει και το θέμα της χρυσή βίζας όπου η Επιτροπή πιστεύει ότι είναι πολύ λίγα τα ωφέλη ε, για τα κράτη-μέλη όταν προσφέρουν τη λύση της χρυσή βίζας. Γι' αυτό στην έκθεση ζητούμε να απαγορευτούν οι χρυσέ βίζες ή η παρομοια καθεστώτα και να αυξηθεί η διαφάνεια ή η ιδέουσα επιμέλεια. Ε, να τελειώσω ευχαριστώντας όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν στην έκθεση αυτή, ιδιαίτερα τον κύριο Κόφο, το συνεισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητέ και ιδιαίτερα εκτιμώ το έργο των συνεργατών μας ε, και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ναι, πράγματι είχατε τέσσερα λεπτά συν δύο, αλλά εξαντλήσατε και τα έξι λεπτά στις ε, εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Ο Επίτροπος, ο κύριος Μοσκοβισή, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε, που θα είναι μάλλον και η τελευταία κατά αυτή τη θητεία για να σας μιλήσω για την κοινή μας μάχη και αγώνα, για τη σωστή φορολόγηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την τεράστια εργασία τους τους εισηγητές και την ε, τάξτρια 3 η οποία συνεδρίασε 34 φορές, έκανε πληθώρα αποστολών και συνέταξε 6 εκθέσεις συνολικά. Και φυσικά ε, το, η εργασία αυτή είναι απότοκη της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Panama Papers. Πρόκειται για μια τεράστια εργασία τα τέσσερα τελευταία χρόνια μπορούμε να πούμε ότι τα δύο θεσμικά όργανα έγιναν σύμμαχοι για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Αυτό φάνηκε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να μιλήσω για τα πιο εμβληματικά σημεία της έκθεσης κατά της φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Είπα ότι το, το παγκόσμιο σύστημα φορολόγησης δεν έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες του 21ου αιώνα, διότι υπάρχουν άειλες αξίες και μία κινητικότητα, την οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Λυπάμαι γιατί δεν φτάσαμε σε μία συμφωνία σε σχέση με τις ψηφιακές ε, υπηρεσίες στο ΕΚΟΦΗΝ στις 12 Μαρτίου. Έχει επιτελεστεί πρόοδος και η φυσική βάση όπως έχει διαμορφωθεί αποτελεί μία καλή αρχή. Θα πρέπει όμως να επιταχύνουμε τις διεθνείς συζητήσεις και εργαζόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν δύο μεγάλοι πυλώνες ε, πέρα από την ε, ψηφιακή αγορά. Τα ε, δικαιώματα φορολόγησης και η ελάχιστη βάση φορολόγησης. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη ότι δεν είμαστε απλώς ένα σύνολο των 27-28. Αποτελούμε μία ενοποιημένη αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών και γι' αυτό το μήνυμα που θα πρέπει να αποστείλουμε είναι ότι θα πρέπει να συντονιστούμε και σε επίπεδο G20. Δεν θα πρέπει να έχουμε πληθώρα προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να μιλάμε με μία φωνή για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, να έχουμε μία απλή, ένα απλό σύστημα φορολόγησης και μία δίκαιη φορολόγηση. Χαίρομαι μετά την Επιτροπή Τάξη για την ψηφιακή αγορά, γιατί φτάσαμε σε μία κοινή βάση για τις 15 δικαιοδοσίες που δεν συνεργάζονται. Και λυπάμαι για την αποδυνάμωση της εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια αξιόπιστη εργασία που έχει μεγάλες επιπτώσεις στα, ε, στη διεθνή σκακέρα. Θα πρέπει λοιπόν να φτάσουμε στην μεταρρύθμιση των διαδικασιών και αυτό με τις ε, δικαιοδοσίες που δεν συνεργάζονται μαζί μας για να φύγουν από την κοινή λίστα τη στιγμή που δεν συνεργάζονται και εκεί που υπάρχει μηδενική βάση φορολόγησης των ε, εταιριών με βάση και τα προστάγματα του ΟΣΑ. Βεβαίως αναγνωρίζω ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν συμμετείχαν στη διαδικασία τάξη 3 όπως θα θέλαμε. Θεωρώ ότι με βάση τις ε, διεθνείς προδιαγραφές χρηστής διαχείρισης δεν υπάρχουν ε, φορολογικοί παράδεισοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγάλη διαφάνεια. Βεβαίως υπάρχουν ε, φορολογικές μαύρες τρύπες σε ορισμένες χώρες που προωθούν πρακτικές υπέρ της φορολογικής βελτιστοποίησης ή μιας επιθετικής φορολογικής πολιτικής. Όμως καταδικάζω αυτές τις πολιτικές και νομίζω ότι έχουμε άλλες βάσεις. Την, τον ενιαίο κατάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τον κώδικα συμπεριφοράς, καθώς και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Υπάρχει ευρεία συμφωνία επ' αυτών. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτά τα μέσα και να ε, τα, να για να υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη και φορολογική διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί που δεν συλλέγονται οι φόροι, ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ευάλωτες κοινωνικές δομές. Εάν οι πιο πλούσιοι δεν καταβάλουν φόρο, γιατί θα πρέπει να το κάνουν οι πιο φτωχοί. Νομίζω ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε ε, στα δεδομένα αυτά, έτσι ώστε οι μεγάλες πολυεθνικές και οι δικαστικές συμφωνίες να προωθηθούν ε, έτσι ώστε να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κρατών Euh, και μέσα στα πλαίσια των φορολογικών συμφωνιών θα δούμε πώς μπορούμε να ε, εξελίξουμε αυτό το σύστημα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει και αντιμετώπιση της φορολογικής επιθετικής πολιτικής για να ε, υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, όπως προβλέπεται από την 1η Ιουλίου 2020. Ε, έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση και από τη δημόσια διοίκηση των κρατών μελών σε όλα αυτά τα δεδομένα. Να μην ε, δεχτούμε δηλαδή την ε, νομιμοποίηση από παράνομα έσοδα και να προωθήσουμε την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με βάση το σχέδιο που προωθεί η συνάδελφος Γιούροβα. Επίσης, ως προς την καταπολέμηση της μη καταβολής ΦΠΑ, γίνονται έρευνες και έχουμε ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών και σε επίπεδο Eurofis και Europol έτσι ώστε να ε, μπορέσουμε να εχνηλατήσουμε αυτές τις δραστηριότητες. Δεν θα ήθελα να είμαι πιο διεξοδικός. Η έκθεσή σας μιλάει από μόνη της θα ήθελα όμως να μιλήσω για ένα άλλο εμβληματικό στοιχείο της έκθεσης που αποτελεί και ένα πολιτικό μήνυμα για τις ευρωεκλογέ και την επόμενη Επιτροπή και Κοινοβούλιο. Δηλαδή να περάσουμε στην ειδική πλειοψηφία. Δέχομαι αυτό το διάβημα και το υποστηρίζω για να περάσουμε στη ρήτρα της πασαρέλας για το μέλλον. Πρόκειται για στοιχεία ε, ζωτικής σημασίας. Θα πρέπει να περάσουμε από, την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία για να μπορεί να δράει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο αποδοτικά και πιο γρήγορα με βάση τις παγκόσμιες προκλήσεις γιατί η ομοφωνία αποτελεί τροχοπέδι. Επίσης, η απόφαση με ειδική πλειοψηφία θα αποτελέσει ε, μία δημοκρατική ενέργεια, γιατί γνωρίζω ότι θα μπορείτε να δράτε ως συνομοθέτης όπως ακριβώς πρέπει και όπως είστε. Επίσης, το πεδίο δράσης της φορολογικής ε, πολιτικής θα διευρυνθεί. Μιλάμε για την φορολόγηση της ενέργειας, της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών και ε, μία ενιαία φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία. Και εδώ μιλάω και για την προστασία του περιβάλλοντος και την διευθέτηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα πολιτικά του κόμματα θα πρέπει να ανοίξουν τη συζήτηση αυτής της μεταρρύθμισης έτσι ώστε να ενισχύσετε τις εξουσίες σας και να δώσετε φωνή στα κράτη-μέλη τα οποία μερικές φορές δεν κατανοούν το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Και εάν αύριο υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία για τέτοιες προτάσεις, τότε θα έχει επιτελεστεί μεγάλη πρόοδος για τη δημοκρατία και την αποτελεσματικότητα. Αυτοί θα είναι οι κανόνες του παιχνιδιού, αλλά και το ίδιο το παιχνίδι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τώρα το λόγο έχουν οι ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες για το ΕΛΚ για 1,5 λεπτό Λάγκεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την έκθεση. 410 επιμέρους σημεία και παρατηρήσεις περιέχει. Είναι το αποτέλεσμα μακρά συνεργασίας πολλών συναδέλφων και πρωτίστως των συνεισηγητών ε, περιλαμβάνεται η εργασία της ΤΑΞ, ΤΑΞ 1, ΤΑΞ 2 και η Επιτροπή Εξεταστική. Το θέμα είναι ο θεμητός, ε, ε, δίκαιη φορολογία. Αυτά πρέπει να μείνουν στην ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου. Δεν αρκεί να συζητούμε για ε, μια θητεία και μετά όλα να λιμνάζουν ξανά. Ε, είναι σωστό και κύριε Μοσκοβισή ε, υποβάλλατε πάρα πολλά αξιέπαινα νομοθετήματα και προτάσεις μέσα στην πενταετία. Αλλά η τελευταία πρόταση στο βαθμό που τα κράτη-μέλη ε, μπλοκάρουν την ε, πρόοδο ακόμα και ο δικός μου υπουργό που τάχθηκε κατά της ψηφιακής ε, φορολογίας στο βαθμό που τα κράτη-μέλη με την ομοφωνία μπλοκάρουν τη διαδικασία δεν θα έχουμε πρόοδο. Οι εκκλήσεις δεν αρκούν. Θα πρέπει να πιάσουμε και τους φορολογικούς παραδείσους μέσα στην Ένωση, να του κατονομάσουμε. θα ονομάσω δύο, το Λουξεμβούργο όπου ε, τα έσοδα προφόρων δεν φορολογούν μπορούν να μην να, να απαλλαγούν από τη φορολογία και η Ολλανδία επίσης. Η κυρία επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους εισηγητές για το, την καλή δουλειά. Τώρα ε, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε επαναστατικά βήματα. Ε, δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 820 μας διαφεύγουν. Ε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε τι, και τι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας για τους νέους που μπλοκάρουν όλα στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει η ομοφωνία στα φορολογικά θέματα να μην ισχύει. Ε, οι Υπουργοί Οικονομικών μπλοκάρουν τα θέματα. Ε, δεν προχωρεί η διαφάνεια σε φορολογικά θέματα. Ε, εμείς θέλουμε να ξέρουμε ε, ποιοι και πού μεγάλοι όμιλοι πληρώνουν τους φόρους τους και πού όχι. Πρέπει επίσης να θεσπίσουμε ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές. Ε, ψηφίστε το αυτό αύριο όταν θα τεθεί σε ψηφοφορία όλη η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριε Σίλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να αρχίσω ε, καταρχήν ευχαριστώντας τους δύο εισηγητές και όλους όσοι συμμετείχαν στην έκθεση αυτή γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεση, είχε πολλές τροποπολογίες, δεν ήταν εύκολο το θέμα. Το ξέπλυμα χρήματος ήταν και παραμένει μεγάλο θέματα στις ε, τρίτες χώρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις όπως αναφέρατε κι εσείς. Ε, οι βελτιώσεις συμπεριλαμβάνουν και την κατάργηση της χρυσής βίζας. Η έκθεση πολύ ε, σωστά ε, επισημαίνει κάποιες τράπεζες ε, ε, που ξεπλένουν χρήμα. Όμως το κείμενο που δυναμώθηκε στην Επιτροπή. Το θέμα δεν δημιουργείται σε μια συγκεκριμένη χώρα ή σε συγκεκριμένες τράπεζες. Υπάρχει ε, ένα ε, ε, σύστημα όπου γίνεται ένα προκαταρκτικό πλήσιμο και μετά το χρήμα ακολουθεί το δρόμο του αλλού. Η ειδική ομάδα έκανε πολλή δουλειά. Υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν είναι ακόμα μέλη της ΦΑΤΦΑ, αλλά Τώρα ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ε, πολλοί, πολλές λειτουργούν και ξεπλένουν χρήμα με διαφορετικό χώρο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γέζεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, μετά τα πρώτα σκάνδαλα περιφόρων, το LuxLeaks και έπειτα, το Κοινοβούλιο έχει αναλάβει γιατικό ρόλο στην καταπολέμηση του φορολογικού εγκλήματος τη φοροδιαφυγής και τη φοροαπάτη. Σε όλο τον κόσμο και με τη δράση μας στις Επιτροπές Τάξη 2 και επάνω έχουμε ε, ερευνήσει το θέμα ενδελεχώς και έχουμε συντάξει και τις αναλόγες συστάσεις για να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αυτά. Στην ε, Επιτροπή Τάξη 3 έχουμε ακόμα ένα παράδειγμα ε, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά και έχουμε ακόμη και ένα κείμενο. Και χάρη στη δουλειά των συνεισηγητών, σκιωδών, συνεργατών μας, της γραμματείας και όλων όσων εργάζονται εκεί και πάλι έχουμε ε, ετοιμάσει συντάξεις για δράσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δείξει την κατάλληλη ανταπόκριση σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και επίσης έχει προχωρήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες. Όμως τα κράτη-μέλη δεν κάνουν αρκετά. Το Συμβούλιο συστηματικά επεκδίεται των φορολογικών ευθυνών και και είναι σαφέ ότι τα, τα ε, μεταξύ των θεσμικών ευρωπαϊκών οργάνων το Συμβούλιο είναι αδύναμο κρίκο. Χωρί πολιτική βούληση δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδο. Είναι σαφέ ότι το Συμβούλιο ζητά τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να συζητήσει τα ζητήματα αυτά και να βρει κάποιε λύσει. Ιδάλω δεν προχωρούμε. Το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να αντιδρά όμω και να ερευνά τα φορολογικά εγκλήματα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτό, αλλά χωρί δράση από του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων θα παραμένουμε παγιδευμένοι σε αυτόν τον φαύλο κύκλο. Οι Ευρωπαίοι αξίζουν καλύτερη τύχη. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε, κύριε Γέζεκ. Και τώρα για του πράσινου. Για ένα λεπτό η κυρία Σκοτ Κέιτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η φοροδιαφυγή είναι τόσο σημαντική για τους συμπολίτε μας, διότι υπονομεύει τις δημόσιες υπηρεσίες, την άνοδο των ανισοτήτων και υπονομεύει και το κοινωνικό συμβόλαιο. Γιατί ε, δεν κάνουμε εδώ ε, δεν επιτελούμε πρόοδο. Σε φορολογικού παραδόσει όπω το Ηνωμένο Βασίλειο, η Μάλτα, το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία. Οι κυβερνήσει του έχουν τι ανάλογε φορολογικέ συμφωνίε, αλλά δεν έχουν ε, συνάψει τι σχετικέ ε, συμβάσει για να προχωρήσουμε σε αντιμετώπιση των φαινομένων. Καλώ έχουμε προχωρήσει στο Κοινοβούλιο σε έγκριση των νομοθετημάτων για να διώξουμε τι εικονικέ εταιρείε από την ήπειρό μα καθώς και την πώληση θεωρήσεων που είναι χρυσές και ψευδείς. Πρέπει όμως να κάνουμε και άλλα βήματα για να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή και τη φοροαπάτη και να μην μπορούν τα κράτη που έχουν δικαίωμα κυρίες να μπλοκάρουν την πρόοδο στη φορολογική μας συνεργασία. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να κάνουμε τις σχετικές έρευνες για το φόρο και να τις ολοκληρώσουμε. Όμως θα πρέπει τα επόμενα μέλη του Κοινοβουλίου στην επόμενη θητή να πιέζουν τα κράτη-μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας για την καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας. Ευχαριστούμε και τώρα για την ΚΟΕ για 1,5 λεπτό, κύριο Ούρμπαν Κρέσπο. Ευχαριστώ, πρόεδρα. Με την ψηφοφορία αυτή ολοκληρώνουμε την εργασία ολόκληρης ευθύτειας για να δούμε πού έγκυται το σφάλμα. Γιατί χάνουμε εκατομμύρια, ε, δισεκατομμύρια από την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Υποτίθεται ότι έχουμε προωθήσει μία πολιτική λιτότητας με το μάντρα ότι δεν υπάρχει χρήμα. Γι' αυτό οι πολίτες υφίστανται το τίμημα. Βλέπουμε ότι στο Λουξεμβούργο καταφεύγουν πολλές επιχειρήσεις για να φοραποφύγουν και γιατί έχουν μηδενική φορολογική βάση. Άρα το χρήμα διαφεύγει σε αστρονομικές ποσότητες. Και αυτό αφορά και την Ελβετία. Πότε θα περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις κατά της Ελβετίας. Πότε πόσο πρέπει να περιμένουμε ε, να ε, προβεί σε κυρώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Λουξεμβούργου και της Μάλτας, που στην ουσία είναι φορολογική παράδειση. Πότε θα καταπολεμήσουμε πραγματικά την ε, φοροαποφυγή. Τη στιγμή που το κεφάλαιο κινείται, αλλά δεν φορολογείται. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κόμπερν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της φοροδιαφυγής και της φοροαπα... φοροαποφυγής. Η φοροδιαφυγή είναι παράνομη και πρέπει να... Η φοροαπα... φοροαποφυγή, μάλλον, είναι παράνομη και πρέπει να σταματήσει. Ναι, φοροδιαφυγή. Ε, είναι κάτι το... Ε, απολύτως ε, ε, αποδεκτό οι εταιρείε στον Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλουν να εκθέτουν του μετόχου του στην υπερβολική φορολόγηση. Είναι πλεονέκτημα όσων έχουν επενδύσει στι εταιρείε δεν ε, γίνεται να ξεχνάμε τα χρήματα που πετιούνται για τους ε, υπέρογκους ευρωπαϊκούς μισθούς και τα δικά σας τα προγράμματα. Και οι εταιρείε εξασφαλίζουν μακροχρόνιες θέσεις εργασίας και δεν ε, πληρώνουν κακομαθημένους υπαλλήλους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δεχτούμε ότι οι εταιρείε φτιάχνουν την απασχόληση. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε μικρο, μικρομεσαίες εταιρείες. Όμω ε, βλέπετε ότι και οι Γάλλοι πολίτε δεν συμφωνούν με τον τρόπο που προχωρεί η Γαλλία, κύριε Μοσκοβεσί. Βεβαίω η λεύκανση ε, βρώμικου χρήματο ε, είναι παρανομή. Όμω υπάρχει τρόπο να χρησιμοποιήσουμε του φόρου και με τρόπο ένομο. Δεν σημαίνει ότι όλα είναι το χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Και δεν μπορείτε να χώνετε τη μύτη σα στι ιδιωτικέ υποθέσει των ανθρώπων. Γι' αυτό η Μεγάλη Βρετανία εγκαταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον έτσι ελπίζω, ε, γιατί με την Πρωθυπουργό που έχουμε δεν βλέπουμε να προχωράει το πράγμα, αλλά πρέπει να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου τη που δεν έχουμε φύγει ακόμα. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Σόσνιερτ, μη εγγεγραμμένο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην έκθεση αυτή βλέπουμε ότι δεν θέλετε να κλέβουμε ε, γιατί οι κυβερνήσεις δεν θέλουν ανταγωνισμό. Οι κυβερνήσεις κλέβουν με τους φόρους, οι κυβερνήσεις παίρνουν τα χρήματα από άλλους για να τα αναδιανύμουν σε άλλους παίρνουν ε, με ό,τι τρόπο μπορούν τι αποταμιεύσει μα. Παίρνουν από τι τράπεζε, μάλλον δίνουν στι τράπεζε το δικαίωμα να δανείζουν επανειλημμένω τα ίδια ποσά. Εάν αυτοί οι άνθρωποι δικάζονταν, θα βρίσκονταν στη φυλακή. Και οι κυβερνήσει δέχονται χειροκροτήματα. Δεν είναι λοιπόν η φοροδιαφυγή το πρόβλημα και η φοροαποφυγή. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι παίρνουν χρήματα κάποιων για να τα δώσουν σε άλλου. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξηγήσουμε και όχι τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. Η φοροαποφυγή χρειάζεται για να μην πάνε τα χρήματα στα χέρια ηλικίων πολιτικών που ούτω ή άλλω θα τα πετάξουν τα χρήματα για άχρηστου σκοπού. Γι' αυτό λοιπόν ε, να ε, σας επισημάνω ότι τα χρήματα για τις διακοπές του Κοινοβουλίου ε, ε, δεν είναι ε, κάτι που θέλουμε να πληρώνουμε. 20 εκατομμύρια μας κοστίζουν οι διακοπέ σα ενώ δεν έχουμε αρκετά για τον Εράσμο και του φοιτητέ. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό κύριο Κάρα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτρόπε, κυρίε και κύριοι, με την έκθεση αυτή φροντίζομαι για μεγαλύτερη δικαιοσύνη και αυτό είναι το μεγαλύτερο πακέτο ε, ετοιμάτων που είχαμε ποτέ. Ξέρουμε πόσο αναγκαία είναι όλα αυτά. Και μάλιστα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκεντρώθηκε ευρεία πλειοψηφία. Έχουμε στήριξη από την Κομισιόν. Υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης σε επίπεδο κρατών μελών. Δεν ε, αναλαμβάνουν να δώσουν τη μάχη και ε, το σύστημα ε, δίνει δυνατότητα σε τέτοιους αποκλεισμούς. Σταματήστε αυτό το μπλοκάρισμα δώστε τις προϋποθέσεις ώστε να έχουμε ψηφιακή φορολόγηση, να έχουμε ε, ενιαία φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις, να υπάρχει η ε, υποχρέωση υποβεβολής εκθέσεων. Συγγνώμη, διακόπτει ο πρόεδρος, πρέπει να... Δώσαμε το λόγο στον επόμενο μιλητή, στον κύριο Τάγκ. Έχουμε χρονικές πιέσεις να τηρείτε το περιθώριο. Ο κύριος Τάγκ, ευχαριστώ. Καταρχήν να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την έκθεση προς τους εισηγητές Νίτερ Μάγερ και Κόφοντα. Εξαιρετική έκθεση. Ε, ευχαριστώ και τον Επίτροπο Πιέρ Μοσκοβισή που επί τέσσερα χρόνια ε, ακούραστα αξιοποίησε κάθε ευκαιρία για να βάλει τους φόρους στην ημερήσια διάταξη. Με επιτυχία. Ε, σας εκτιμώ βαθύτατα γι' αυτό. Ε, τώρα, το θέμα που μας απασχολεί είναι η μεγαλύτερη αυξανόμενη ανισότητα που μεγενθύνεται από την φοροαποφυγή ε, που επιτρέπει ε, στους πλούσιους ε, να ε, αποκρύπτουν φόρους και να τους μεταβιβάζουν στο 99% των υπολείπων. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε διαρθρωτική μεταρρύθμιση σχετικά με τον, τη φορολογία των επιχειρήσεων. Προχωρήσαμε μετά από πρόταση κομισιών, θα γίνει και στην ΩΣΑ συζήτηση και πρέπει να έχει ενιαίο μέτωπο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η διανομή κερδών είναι ένας τρόπος για να ε, σταματήσει αυτή η μετατόπιση των κερδών. Δεύτερον, είναι σαφές ότι τουλάχιστον πέντε κράτη-μέλη της Ένωσης είναι φορολογική παράδειση. Ε, μόνο το όνομα δεν υπάρχει. Ε, έτσι μειώνονται οι ε, φόροι. Να μιλήσουμε για την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο. Ε, αυτή είναι φορολογική παράδειση. Υπάρχουν και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παίρνουμε μέτρα. Πρέπει όμως να μιλήσουμε και για τους φορολογικούς παραδείσους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας και ας ψηφίσουμε την έκθεση αύριο. Υπάρχει η γαλάζια κάρτα από τον κύριο Κόμπερν για σας. Την δέχεστε, έχετε μισό λεπτό κύριε Κόμπερν. Ευχαριστώ κύριε Τάγκ. Ε, προφανώς ε, υπάρχουν εταιρείε που δεν συμφωνούν με αυτά που λέτε και δεν είναι τόσο ότι ε, χρήματα αλλά πολλές φορές κατασπαταλούνται χρήματα για παράλογα ε, προγράμματα. Θα πρέπει να υπάρχει μια οικονομία όπως το Ηνωμένο Βασίλειο που θα δημιουργείται από τις επιχειρήσεις και, θα υπάρχει ανάπτυξη και απασχόληση που θα δημιουργείται όχι από το κράτος αλλά από τις επιχειρήσεις. Και ποια είναι η ερώτηση. Εγώ θέλω να απαντήσω όμως. Προσπάθησα να βρω την ποια ερώτηση ήταν, αλλά ο κύριος Τάνκ το κατάλαβε και θα απαντήσει. Ένα παράδειγμα θέλω να σας δώσω. Ε, στα Paradise Papers, η Nike που είναι στην Ολλανδία η έδρα της, πληρώνει 33% ε, φόρος επί των κερδών πλήρωσε το 2017 το, το 2017 ήταν 13% στην κρίση το φορολογικό βάρος μειώθηκε ποιος πληρώνει περισσότερους φόρους αυτοί που εργάζονται που έχουν, είναι μισθωτοί δηλαδή οπότε ναι τα ε, κίτρινα γυλαίκα νομίζω ότι θα ε, συμφωνούσαν με αυτή τη διαδικασία Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Λέρνεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, στην Επιτροπή Tax 3 λάβαμε νέες πληροφορίες ε, για την φοροδιαφυγή και το εύρος αυτού του φαινομένου. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ανέκυψαν στην Εσθονία... 200 δις νομιμοποιήθηκαν από παράνομα ε, έσοδα. Οι καταγγέλτες ε, ευτυχώς είχαν αναφερθεί σε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Πολύ συχνά οι τράπεζες δεν θέλουν να κοιτάξουν και πολύ μακριά τη στιγμή που διατίθενται πολλά χρήματα. Οι επιτροπή αυτή μας ε, ε, κατέδειξε και ένα από τα μεγάλα σκάνδαλα όπου ε, ρωσικοί κύκλοι χρησιμοποίησαν τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Ζολή, για ένα λεπτό. Σε μερικές εβδομάδες θα αποχωρήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από 10 χρόνια μαχών κατά της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής. Είμαι και ικανοποιημένη αλλά και δυσαρεστημένη. Χαίρομαι αφενός γιατί μετά από 10 χρόνια επειδή ακριβώς υπήρξαν καταγγέλτες και μετά από την ε, υπέροχη εργασία των εισηγητών υπάρχει μεγαλύτερη ε, διαφάνεια και συνεργασία. Είναι η δική μας βεβαίως νίκη, νίκη των πρασίνων. Λυπάμαι όμως γιατί οι ιδέες δεν ε, μετασχηματίστηκαν σε δράση. Χρειάζονται πολλές μεταρρυθμίσεις και θα πρέπει επίσης να γίνεται και κατάδοση όταν ε, υπάρχει ε, διαφθορά ή όταν ε, υπάρχει φοροδιαφύγη, έτσι ώστε η φορολογική δικαιοσύνη να είναι στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποτελέσει πραγματικότητα. Κάρθι, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να υπερασπιστούν τα εθνικά συστήματα φορολόγησης. Θα πρέπει να τύχουν προστασίες. Η φορολογική κυριαρχία δεν διαπραγματεύεται, αλλά θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στα εταιρικά συμβόλαια και φορολογική απόδοση ακούμε τους ε, πολίτες σε σχέση με τους εταιρικούς φόρους. Κατά το Tax 3 είδαμε ότι με τη βοήθεια της Ιρλανδίας η Apple έχει δημιουργήσει νέα διάρθρωση και δεν έχει αποδώσει, δεν 2,5 δις ε, σε φόρους από το 2015 και αυτό μέσω των άειλων περιουσιακών στοιχείων και φαίνεται ότι και η ίδια η Apple έχει διαφύγει του Ιρλανδικού δικαίου. Νομίζουμε ότι πρόκειται για επιλεκτική μεταχείριση και θα πρέπει να δούμε τις κρατικές ενισχύσεις. Αν δεν το αντιμετωπίσουμε τότε θα πλήξουμε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Φουντούλης για ένα λεπτό. Όλοι πλέον θα έπρεπε να μπορούν να αντιληφθούν τις εγγενείς παθογένειες της λεγόμενης ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως luxleaks panama papers paradise papers football leaks bahamas leaks cum ex και πόσα ακόμη οικονομικά σκάνδαλα δεν έχουν αποκαλυφθεί δείχνουν το μέγεθο του προβλήματο. δεν μπορεί να υπάρξει ενιαία αγορά όσο υπάρχουν διαφορετικά φορολογικά συστήματα στα κράτη μέλη. όσο ισχύει αυτό θα οδηγούμαστε σε νόμιμη φοροαποφυγή προ όφελο των μεγάλων εταιριών και γενικά όσων διαθέτουν τα χρήματα και τα μέσα για κάτι τέτοιο όμω η παράδοση φορολογική εξουσία στην ευρωπαϊκή ένωση θα συνιστούσε ουσιαστική κατάργηση των εθνικών κρατών και κάτι τέτοιο για εμά είναι ανεπίτρεπτο. επιπλέον ποτέ οι λαοί τη ευρώπη δεν έχουν ερωτηθεί αν το επιθυμούν αυτό. Τέλο, όσον αφορά τη δυνατότητα ελέγχου εκ μέρου του ευρωκοινοβουλίου είμαστε σύμφωνοι και υποστηρίζουμε την παραχώρηση τέτοιων δικαιωμάτων. το μόνο άμεσα εκλεγμένο όργανο τη ενώσεω είναι εκείνο το οποίο διαθέτει την νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο. με την ευκαιρία τη εθνική επετείου τη επαναστάσεω του 1821 να ευχηθώ σε όλους τους έλληνες χρόνια πολλά και ζήτω το έθνος. ευχαριστώ. Thank you for one minute. Για ένα λεπτό, κυρία Σαντέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, η δουλειά που έχει γίνει στα επίπεδα τη Επιτροπή Tax 3 είναι ένα σαφέ μήνυμα πριν τι ευρωπαϊκέ εκλογέ. Και αποδεικνύει ότι υπάρχει σαφή βούληση και φιλοδοξία από την πλευρά των Ευρωβουλευτών να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο, την φόρο αποφυγή και το σύνολο των οικονομικών σκανδάλων που μα πλήττουν. Τώρα όμω η μπάλα έχει περάσει στο γήπεδο των κρατών μελών. Είναι σημαντικό να δείξουν και εκείνοι ότι διαθέτουν πολιτική φιλοδοξία περισσότερη από ό,τι έχουν δείξει τώρα. Και αυτό με αφορμή την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου στι προτάσεις μας να χρησιμεύσουν, να χρησιμεύσουν ως αφορμή για τι επόμενε δράσει. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στην εναρμόνιση τη φορολογική βάση των εταιριών, την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή βάση του ΦΠΑ και την φορολόγηση των ψηφιακών εταιριών. Όμω τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν κυρίω τι ευθύνε του και είναι σημαντικό να μπορέσουμε να ψηφίσουμε με ενισχυμένη πλειοψηφία για θέματα που έχουν να κάνουν με την φορολόγηση. Είναι ο μόνος τρόπο για να υπάρξει περισσότερη φορολογική δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κυρία, ο κύριο Σάντ η καταπολέμηση των παραβιάσεων στα θέματα των αφορολογικών είναι σημαντικό προκειμένου να υπάρχουν κατάλληλε λύσει και τα ένδικα μέσα. Εδώ δυστυχώ η έκθεση είναι πολύ σύντομη. Απλώ βασίζεται σε εικασίε και κατηγορίε. Τα ε, στοιχεία των ε, φοροτεχνικών ε, πρακτικών πολλέ φορέ συνδέονται με σοβαρά εγκλήματα, πολλέ φορέ ει βάρο μικρών κρατών. Ε, και με σοβαρέ απώλειε. Γι' αυτό λοιπόν να δοθεί έμφαση και σε αυτή τη διάσταση. Η Deutsche Bank στη Γερμανία έχει δημιουργήσει τριγμού και σε άλλε χώρε. Ενώ οι χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε πολλέ φορέ βρίσκονται στα χέρια εγκληματικών δράσεων. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει φορολογική εναρμόνιση. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρχει και μια επίοικια ε, στα φορολογικά για μερικέ μικρέ χώρε που δυσκολεύονται στην εσωτερική αγορά. Θα πρέπει λοιπόν η έκθεση αυτή να λάβει υπόψη και πολιτικέ θεωρήσει. Δεν μπορεί να πιέζουν απλώ για κάποια πράγματα που θα μπορούσα να αποκαλέσω εγώ φορολογικό λαϊκισμό. Η έκθεση αυτή, το επαναλαμβάνω, είναι σαφώ σε λάθο κατεύθυνση. Ευχαριστούμε κύριε Σάντ. Ο κύριε. Ε, Γκόμε έχει ψώσει γαλάζια κάρτα. Τη δέχεστε την ερώτησή τη. Κύριε Σαν, ε, κυρία Γκόμε έχει να σα κάνει ερώτηση βάσει γαλάζια κάρτα. Δέχεστε, κυρία Γκόμε. Ναι, συμφωνώ απολύτω, κύριε Σαντ. Μάλλον διαφωνώ κάθετα, κύριε Σαντ. Και ήθελα να ρωτήσω τι κάνετε εσεί για να γίνει η χώρα σα ε, κάτι άλλο εκτό από φορολογικό παράδεισο. Αμφισβητείτε την καταπολέμηση του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματο και την χρηματοδότηση τη τρομοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνετε εσεί για να τα εμποδίσετε αυτά την, ε, τον τζόγο, την ε, κρυπτονομίσματα και όλα αυτά που συνέβαιναν με το Panama Papers. Ε, δύο μέλη της κυβέρνησής σας ακόμη δεν έχουν παρατηθεί, ενώ έχουν αποκαλυφθεί στοιχεία εναντίον τους βάσει του Panama Papers. Τι κάνετε για να τα εμποδίσετε, κύριε Σάντ. Πρόεδρε, θα επαναλάβω αυτά που μόλις διάβασα. Δυστυχώς η έκθεση και η κυρία έκθεση μαζί της απλώς κοιτάζει ε, εικασίες και κατηγορίες που είναι θεωρητικές. Ε, πολλές φορές οι πρακτικές αυτές των φροντεχνικών συσχετίζονται με ε, αβάσιμα στοιχεία που έχουν να κάνουν με εγκληματική δράση. Δεν είναι τρόπος αυτός μια σοβαρή ευρωβουλευτής να ε, προχωρεί σε αποφάσεις, λήψη αποφάσεων. Κύριε Γκίγκολτ, για ένα λεπτό. Τα τελευταία πέντε χρόνια σε τέσσερις επιτροπές και ερευνητικές επιτροπές εξετάσαμε το θέμα ξέπλυμα, φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή. Τα πέντε χρόνια αυτά κάναμε περισσότερες πρόοδους από ό,τι τα προηγούμενα 20 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντικές προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως έχουν μπλοκαριστεί τώρα στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών και με ενοχλεί πάρα πολύ ότι η μεγάλη πλειοψηφία, η μεγάλη, ο μεγάλος στη Γερμανία αντιτίθεται στην ε, διαφάνεια και την ψηφιακή φορολογία. Ήρθε η ώρα ο αποκλεισμό ενάντια στη φορολογική δικαιοσύνη να πάρει τέλος. Και αυτό πρέπει να γίνει θέμα και στην προεκλογική εκστρατεία. Δεν μπορεί να μιλάμε για φορολογική δικαιοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι χριστιανοδημοκράτες, οι σοσιαλδημοκράτες ε, στο Συμβούλιο Υπουργών να ε, μπλοκάρουν τις σχετικές ε, προτάσεις. Ο συνάδελφος Μαν ε, θέλει να σας κάνει ερώτηση, να έχει γαλάζια κάρτα. Δέχεστε, ναι. Και εγώ ήμουν στις τρεις επιτροπές τάξ και στα Panama Papers και στην Ερευνητική Επιτροπή και χαίρομαι για αυτά που είπαν οι καταγγέλτες, αυτοί οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Γιατί όμως τα κράτη-μέλη δεν κινήθηκαν αρκετά οι διαφορετικοί υπουργοί οικονομικών. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν είπαν ότι θα φροντίσουμε ώστε επιτέλους ε, να αλλάξει αυτό ότι όλα θα ρυθμίζονται σε επίπεδο κρατών μελών και κάποια θέματα θα αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριος Γκίγκολτ, λυπάμαι καταρχήν πολύ διότι... Ε, περιορίζεται η, η ευρωπαϊκή συνεργασία από μικρά κράτη που έχουν οικονομικό συμφέρον. Κέρδη που δημιουργούνται αλλού να φορολογούνται χαμηλότερα στα ίδια. Και αυτό είναι απαράδεκτο στην εσωτερική αγορά. Επίσης ε, όταν αρχίσαμε να εργαζόμεθα, ευχαριστώ τον διακόπτη ο πρόεδρος, τον κύριο Γκίγκολτ. Ο κύριος Σίρδεβαν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα φορολογικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών δείχνουν σαφώς την ε, φρενήρη ενέργεια των ε, ομίλων να προχωρούν σε ε, ε σε φοροδιαφυγή. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ χάνονται από την παιδεία, την υγεία, ε, την κοινωνική πρόνοια. Οι Ευρωπαίοι θέλουν φορολογική δικαιοσύνη και γι' αυτό χρειάζεται κατεπηγόντως ένα κοινοβούλιο που θα έχει δημοκρατικά εργαλεία στα χέρια του για να ε, βοηθήσει Χρειάζεται μόνιμη υποεπιτροπή που θα ασχολείται στο Κοινοβούλιο με το οργανωμένο το οικονομικό έγκλημα και τη φοροδιαφυγή. Επίσης χρειάζονται ελάχιστοι συντελεστές για την εταιρική φορολόγηση και ε, αναχώρα έκθεση ούτως ώστε να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η φοροδιαφυγή. Ευχαριστώ. Ε, Τελευταία γαλάζια κάρτα, μετά δεν έχουμε χρόνο για άλλες. Ε, ο κύριος ε, Σόσνιετ ε, θέλει να σας κάνει ερώτηση στα πλαίσια της γαλάζιας κάρτας. Δέχεστε? Αυτή είναι η τελευταία γαλάζια κάρτα που δεχόμαστε όμως, σας το ξαναλέω. Η φορολογική δικαιοσύνη τι είναι. Μία είναι η δικαιοσύνη. Ε, ε, γιατί έχουμε δικαίωμα να φορολογούμε κοιτάζοντας τις τσέπες του καθενός πόσα βγάζει και να τα φορολογούμε. Γιατί πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό το δικαίωμα. Ε, συνάδελφοι, η φορολογική δικαιοσύνη αξιολογείται από εσά διαφορετικά, από μένα διαφορετικά. Η επιχείρηση όμως μπορεί να μειώνει τους φόρους ανεξέλεγκτα σε βάρος της κοινωνίας. Κάποτε πρέπει να υπάρχουν ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές που δεν θα το επιτρέπουν αυτό. Δεν μπορεί να υπονομεύουμε συνέχεια την κοινωνική πρόνοια. Ε, γι' αυτό χρειάζεται φορολογική δικαιοσύνη που θα δίνει ίσες προοπτικές ανάπτυξης για όλους τους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ Κύριε Σάντσεθ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την εργασία τους. Άκουσα και τον κύριο Μοσκοβισή, ο οποίος παρακολουθεί αυτή την διαδικασία σήμερα και ο επιχειρηματικός κόσμος προσπαθεί να καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή και αυτό αυτό έτσι ώστε να υπάρχει μια ενιαία φορολογική βάση η οποία να είναι πιο ε, δίκαιη. Και αναφέρομαι και στην ψηφιακή ε, φορολογία και στην αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, η οποία δεν ήταν αποδοτική. Δυστυχώς αυτή η διαδικασία ήταν άκρος ε, δυσλειτουργική και αργή και τα στοιχεία είναι αστρονομικά ως προς την ε, διαφυγή, όπως μας είπε και ο Επίτροπος. Ευχαριστούμε πολύ η κυρία Γκόμες για ένα λεπτό. Η έκθεση αυτή προτείνει μια Ευρώπη που δεν θέλουμε να έχουμε όπως φορολογικές παραδείσους στην Κύπρο, την Μάλτα, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και ε, επίσης με ειδικέ ε, συμφωνίες στην Μαδέρα και στις Ασόρες. Εδώ θα πρέπει να μην στηρίζουν οι κυβερνήσεις ε, οργανώσει οργανώσεις ολόκληρου του κόσμου. Θα πρέπει να μην πληρώνουν το τίμημα οι πολίτες για να στηρίζονται οι τράπεζες διότι με τέτοια δημόσια ελλείμματα οι πολυεθνικές μαζεύουν απλώς ε, μεγάλα ποσά και συγκεντρώνουν περιουσίες. Όπως συνέβη στη χώρα μου με την παρέμβαση της Τρόικας όμως την πληρώνουν τα κράτη και πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε φορολογική δικαιοσύνη, διότι μεγάλε εταιρείε ε, τη τεχνολογία και του ψηφιακού χώρου ε, συνεχίζουν να μην πληρώνουν φόρου, ενώ ε, με την κυκλική απάτη και την απάτη του ΦΠΑ υποφελούνται οι τρομοκρατικέ οργανώσει που χρηματοδοτούνται από αυτά. Θα πρέπει λοιπόν στην εσωτερική αγορά να πάψει το φορολογικό dumping, να πάψουν οι φορολογικέ συμφωνίε σε διεθνή κλίμακα που απλώ βελτιώνει τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε τον ειδικό, την κοινή ενωπομημένη ευρωλογική βάση ε, για τις εταιρείε της ECBTB. Ευχαριστούμε συνάδελφο κύριο Κάζα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι καθήκον μας να προασπιστούμε τους πολίτες μας. Ε, γι' αυτό ε, ανέκαθεν ήμουν κατά της κατάχρησης εξουσίας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τη διαφορά, ούτε την κλοπή ει βάρο των συμπολιτών μα, ακόμη και αν είναι από μέρου κυβερνήσεων. Θα πρέπει οι πολίτε να είναι η πρώτη προτεραιότητα και η πρώτη μέρημνα πριν από κάθε άλλη μα μέρημνα. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι η έκθεση αυτή, τουλάχιστον από την Σκοπιά των Πολιτών, είναι μια καλή έκθεση. Όμω πρέπει να είμαστε συνεκτικοί. Οι προτάσει τη αριστερά για φορολογικού σκοπού δεν μπορούν να ισχύουν μόνο για ορισμένου πολίτε. Θα πρέπει λοιπόν τι προτάσει αυτέ να τις ε, δούμε ε, σοβαρά. Υπάρχουν αποφάσεις για να ενισχύσουμε τα φορολογικά μας συστήματα, να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, πράγμα που δεν έχει γίνει ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν θα καταπολεμήσω οποιαδήποτε πρόταση που μπορεί να πλήττουν τις θέσεις εργασίας σε κράτη-μέλη όπως η Μάλτα και τον Κόζο. Ήμουν υπέρ τη εθνικής κυριαρχίας για τον καθορισμό των φορολογικών συστημάτων από τα μελη Ευχαριστούμε, κύριο Σάιμον, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Μοσχοβησία, αγαπητοί συνάδελφοι, πέντε χρόνια η Σοσιαλδημοκρατική Ομάδα στην Ειδική Επιτροπή, Επιτροπή τάξε 1, 2 και στην Ερευνητική Επιτροπή συνέβαλε αποφασιστικά. Ήταν πολύ θετική η περίοδος αυτή, προχωρήσαμε σε επίπεδο ρυθμιστικό, κανονιστικό και από την Κομισιόν είχαμε έναν εξαιρετικό συνεργάτη εταίρο στο πρόσωπο του Επιτρόπου Μοσχοβησί ε, που έκανε πολλές προτάσεις για αποτελεσματική καταπολέμηση του ξεπλήματος και της φοροδιαφυγής. Για το μέλλον είναι σημαντικό τα αιτήματα για μόνιμες δομές που προήλθαν από τις επιτροπές να ενισχυθούν. Υπάρχει από την ομάδα μου σχετική τροπολογία. Πρέπει διαπαραταξιακά να συνεργαστούμε γιατί θα πρέπει να δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Ε, κάποιος που εργάζεται σε θέματα οικονομικά, νομισματικά θα δει τα πράγματα από ό,τι αναγκόμες από άλλη επιτροπή. Ε, δεν έχετε άλλο χρόνο. Ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Ο κύριος Χέι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, ήδη γνωρίζουμε ότι είμαστε μια κοινότητα δικαίου και οι συνθήκες είναι σαφές σε σχέση με την απέτηση ομοφωνίας για τα φορολογικά. Θα πρέπει λοιπόν τα μικρότερα κράτη-μέλη να μην είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τα μεγαλύτερα κράτα που έχουν περισσότερο, μεγαλύτερο πληθυσμό και ε, υψηλότερη, πιο διευρυμένη φορολογική βάση. Έχουμε κάνει πρόοδο σε επίπεδο ΣΑΜΠΕΠΣ και στον έλεγχο χώρα προς χώρα, καθώς και το, το, ως προς το EMLD 4. Αλλά δεν υπάρχει πλειοψηφία στο ε, Συμβουλίο για το ψηφιακό φόρο, CCCTB, και τον κοινό φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει μια άλλη τακτική έτσι ώστε να εγγράψει και να οριοθετήσει τις καλύτερες πρακτικές που να είναι μετρήσεις και να γίνεται μια ετήσια εποπτεία και να συντάσσεται μια ετήσια έκθεση. Ράντευ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Τα πρόσφατα σκάνδαλα όπως αυτά των εγγράφων του Παναμά, Λουξ, και τα δις που νομιμοποιούνται μέσω τραπεζών δείχνουν ότι πρέπει να διανύσουμε πολύ δρόμο για να γίνει πιο αποδοτικός ο δρόμος καταπολέμησης νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Η Επιτροπή Tax 3 κάνει πολλές συστάσεις και προτάσεις για την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας φοροοικονομικού εγκλήματος. Υπάρχουν κράτη που δεν δέχονται να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Δεν θα πρέπει να υπάρχει απόρριτο, θα πρέπει να γίνονται ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και αυτό ως προς τις ε, φορολογικές τους αρχές. Ελπίζω αυτή η αρχή να γίνει υποχρεωτική με συγκεκριμένες προθεσμίες. Δεν πρόκειται μόνο για την ε, ευρωπαϊκή ε, ροή, αλλά θα πρέπει να δούμε ποια είναι η διαδικασία ροής των παράνομων εσόδων. Λοιπόν, έχουμε ένα μακρύ κατάλογο Catch the Eye. Ε, θα ήθελα να τηρήσετε το χρόνο σας, Ντροϊεύσκη. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να ε, τονίσω το γεγονός ότι στην ίδια τη συζήτηση και ενώ εργαζόμαστε για τη σύνταξη αυτού του εγγράφου, υπάρχουν ακόμα περισσότερα ζητήματα παράθετικά. Και θα ήθελα να σας τα κατονομάσω. Οι χρυσές ε, βίζες και το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργούν. Οι διαδικασίες εφαρμογής ε, που είναι πολύ αργές. Τα χάσματα στον νόμο και η φορολογική παράδειση. Αυτά θα ήθελα να τα τονίσω γιατί δεν νομίζω ότι η νομοθεσία θα αλλάξει τα πάντα. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και να φτάσουμε σε συμφωνίες που να είναι αποτελεσματικές. Ο κύριος Καπούτο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η ειδική, η ειδική έκθεση για τη φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή και το ε, τα υπόλοιπα φορολογικά θέματα μας δίνει μια σαφή βάση για να καταπολεμήσουμε τις, ε, τα προβλήματα που έχουμε τα φορολογικά στην Ευρώπη. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν δείξει όμως απαραίτητη πολιτική βούληση για την καταπολέμηση των ε, χρηματοοικονομικών ε, και φορολογικών εγκλημάτων και της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Πρέπει να υπάρξει μια κοινή βάση, κυρίω για τι εταιρείε του χώρου των ψηφιακών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μια μεταρρυθμίση που να επιτρέπει να δοθεί ένα τέρμα στι ειδικέ φορολογικέ συμφωνίε και διακανονισμού ε, των κατομελών, όπου, ώστε κράτη όπω το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Κύπρο, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία και άλλοι να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται τι φορολογικέ του διευκολύνσει. Αυτό δεν μπορεί πλέον να, κρατάει, να συνεχιστεί. Θα πρέπει να συντονιστούν οι εθνικέ προσπάθειε ε, και όλοι να συμφωνήσουν να δημιουργήσουν μια φορολογική αστυνομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με δυνατότητε ερευνητικέ και εισαγγελικέ. Ευχαριστούμε. Τόντο, νομίζω ότι έχει γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια και θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε πανευρωπαϊκά την φοροδιαφυγή. Νομίζω ότι η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών ε, δεν αρκεί. Τα κράτη μεταξύ τους δεν μπορούν να βλάπτουν το ένα το άλλο. Είναι ε, όνειδος να υπάρχουν ε, φορολογική παράδειση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη στιγμή που υπάρχει μία ενιαία αγορά δεν πρέπει να επιτρέψει κάτι τέτοιο. Και επίσης ως προς τον κανόνα της ομοφωνίας, στην ουσία είναι δικαίωμα βέτο των ε, κρατών που δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Θα πρέπει να το δούμε με τις ρήτρε ε, τύπου πασαρέλας. Γι' αυτό θα πρέπει να εργαστούμε και στην αναθεώρηση των συνθήκων. Η κυρία Τόμασίτς για ένα λεπτό. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και την, πώς θα καταπλωμίσουμε τις κλιματικές αλλαγές καθώς και τις παράνομες δραστηριότητες. Αυτές οι εκθέσεις μιλάνε για τη δημιουργία νέων υπερεθνικών δομών, κάτι το οποίο δεν είναι απόλυτα αναγκαίο αυτές οι νέες αρχές δεν θα αποτελέσουν προστιθέμενη αξία, μάλλον θα αποτελέσουν άχθος. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και να καταβάλλεται συστηματικά ο ΦΠΑ. Να μην υπάρχει ε, παραεναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καταπολεμώντας τις απάτες για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Αντίθετα με τους περισσότερους από εμά, κάποιοι μεγάλοι επιχειρηματίες δεν θέλουν, δεν πιστεύουν ότι πρέπει να πληρώνουν φόρους. Η έκθεση δείχνει τη διεθνή διάσταση και το εύρος του προβλήματος. Η Τερίζα Μέη ε, τώρα ασχολείται με το Brexit ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Ε, οι συμπατριώτες μου βλέπουν ε, μεγάλα προβλήματα στις κοινωνικές υπηρεσίες, μέτρα λιτότητας και τα... Οι πιο φτωχοί και ευάλωτοι στην κοινωνία ζημιώνουν από το οικονομικό έγκλημα. Το συντηρητικό κόμμα όμως υπεράσπιζε τους τραπεζίτες που θέλουν πάντα περισσότερα. Εμείς θα πρέπει να έχουμε ένα ε, πρόγραμμα ε, που θα καταπολεμεί τους ε, offshore παραδείσους. Θα πρέπει να πάμε στο βάθος του προβλήματος. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής. Ε, καθίσταται σαφές ότι η έκθεση αντιμετωπίζει την φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή. Έχει κάνει μεγάλο πρόοδο, έχει κάνει μεγάλη πρόοδο, όμως το Συμβούλιο θα πρέπει να ξεκινήσει μια, μια νέα διαδικασία έτσι ώστε να προχωρήσει και η φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απαλληφθεί η αρχή της χρυσής βίζας και δεν μπορούμε να μειώνουμε τους συντελεστές εταιρικού φόρου σε ορισμένα κράτη. Ο κύριος Πάμπλο Κασάδο θα ήθελε να μειωθεί ο εταιρικός φόρος στην Ισπανία κάτω του 20% κάτω το 20% και ελπίζω αυτή η έκθεση να περάσει με μεγάλη πλειοψηφία αύριο. Πένιο λεπτό. Ευχαριστώ. πολύ κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή, η φορολογική παράδοση, παράδειση, όλα αυτά επηρεάζουν όχι μόνο οικονομικά, ε, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Ε, ε, ε, αν υπάρχουν λίγοι πλούσιοι που χρησιμοποιούν αυτά τα τρία εργαλεία και επιτυγχάνουν τεράστια κέρδη εκατομμυρίων και όταν αποδυναμώνεται συνεχώς η μεσαία τάξη, όταν αυξάνονται οι φτωχοί, ε, αυτό είναι απαράδεκτο. Ε, και έτσι αυξάνεται και ακροδεξιά. Νομίζω ότι μπορούμε να απαγορεύσουμε ε, όλες αυτές τις εικονικές επιχειρήσεις ε, και ομίλους που βρίσκονται στους λεγόμενου φορολογικού παραδείσους και πρέπει να έχουμε και μια ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική που δεν θα επιτρέπει να έχουν ε, πλεονεκτήματα στα κράτη-μέλη μεγάλες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς στην ομάδα των Πρασίνων θέλουμε φορολογική δικαιοσύνη, καταπολέμηση, φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και θεωρούμε ότι η έκθεση είναι ισορροπημένη. Η δέσμευση του Κοινοβουλίου ακόμα όμως ε, δεν έχει ε, πραγματοποιηθεί. Δικαιοσύνη στα φορολογικά, ε, καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, απαγόρευση των φορολογικών παραδείσων. Δεν θέλουμε να υπονομεύονται τα έσοδα και το δημόσιο συμφέρον πολλά κράτη-μέλη δεν επιδεικνύουν την απαραίτητη πολιτική βούληση για, ε, και δεν δέχονται θέματα ενιαίου ε, φορολογικού συντελεστή, ελάχιστου κλπ. Ή αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να παρακάμψουμε το κανόνα της ομοφωνίας ε, και να κινηθούμε προς ειδική πλειοψηφία, ούτως ώστε να είναι το Κοινοβούλιο συνομοθέτης και όχι απλώς να παρέχει συμβουλευτικές γνώμες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, το κείμενο που θα εγκρίνουμε είναι τελική πενελιά σε μια συνεκτική, ενδελεχή και συστηματική δουλειά του Κοινοβουλίου εδώ ε, και βάσει ετοιμάτων της κοινή γνώμης που όμως και πολλά σκάνδαλα, ε, για να το πω και στο σωστό γαλλικό πληθυντικό, ε, μας παρότριναν να ερευνήσουμε. Εδώ λοιπόν ανοίγει ο δρόμος για την επόμενη θητή του Κοινοβουλίου διότι περιέχονται πολλές χρήσιμες συστάσεις στο κείμενο αυτό μεταξύ των οποίων που ελπίζουμε να οδηγήσουν σε σύσταση Μόνη μόνιμη υποεπιτροπή. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τι φορολογικέ συμφωνίε, να σταματήσει η έκδοση χρυσών θεωρήσεων ή η υποστήριξη όσων ε, ουσιαστικά αποτελούν σύστημα ξεπλήματο βρώμικου χρήματο. Θα πρέπει να χτενίσουμε στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση όλου του κανόνε για να δούμε ποια δεν είναι νόμιμα και να δημιουργηθεί και μια χάρτα συνεργασία των ε, χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πρέπει να πάψουν να υπάρχουν φορολογικοί παράδεισοι. Αυτή την πραγματικότητα θα πρέπει να σταματήσουμε να την δεχόμαστε, όπω και να υπάρξει ένα ελάχιστο φορολογικό συντερνιστή για τι εταιρείε. Ευχαριστούμε. Τελευταίο στα πλαίσια τη διαδικασία αυτή, ο κ. Βιέγκα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η φοροαπάτη και φοροδιαφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα δις ευρώ. Στην Πορτογαλία είναι 10.000 εκατομμύρια. 10 δις αυτά που χάνουμε. 10 δις στην Πορτογαλία είναι αυτά που χάνουμε και ο φόρος ε, στον ΦΠΑ ε, που είναι ο μόνο ε, εναρμονισμένο φορό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο σημαντικότατο ε, με τι απάτε που γίνονται στι απώλειε. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη φορολογική εναρμόνιση. Στι χώρε μα ε, φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα διαφάνειας, ανταλλαγής πληροφοριών. Θα πρέπει αυτή η ιερία γελάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι απόλυτα ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, να πάψει. Θα πρέπει να σταματήσουμε να δεχόμαστε τέτοιου είδους πρακτικές, την επιθετική φορολογική, ε, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, διότι είναι έκφραση του καπιταλισμού και επίσης της πάλης των τάξεων υπέρ των κυρίαρχων Ευχαριστούμε κύριε που έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι για αυτή την ανταλλαγή απόψεων, τα πολλαπλά σας σχόλια που δείχνουν ότι σας απασχολεί αυτό το ζήτημα εκ του σύνεγγης. Ε, έχουμε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να προωθήσουμε την φορολογική δικαιοσύνη από το 2015% και τα 20 τελευταία χρόνια, σε σχέση με τα 20 τελευταία χρόνια, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει όμως να δώσουμε ένα μεγάλο αγώνα και να τονίσω ότι προασπίζεστε πληθώρα ε, ιδεών και χαίρομαι γι' αυτό να μην υπάρχει δυνατότητα μεταφορών μεταξύ επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μία ε, ρήτρα κατά των καταχρήσεων. Επίσης, μία ελάχιστη φορολογική βάση όπως ορίζει ο ΟΣΑ. Μεγαλύτερη διαφάνεια για τις ε, φορολογικές προδιαγραφές και σχήματα των κρατών μελών και η διαφάνεια θα πρέπει να ισχύει για όλους, δεν θα πρέπει να μείνει καμία μαύρη φορολογική τρύπα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία διαφανής φορολογική βάση και αυτό αφορά την ενιαία φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις. Ο κύριος Λαμασούρ εργάστηκε επί του θέματος αυτού. Επίσης, μεταρρύθμιση του ΦΠΑ για να σταματήσουν οι μαζικές απάτες. Αυτό το ζήτημα είναι ύψης της σημασίας. Μιλάμε για 50 δις ευρώ και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε 40 δις οικονομίες ετησίως ως προς τις ε, επιθετικές φορολογικές πολιτικές θα πρέπει να είμαστε πολύ φιλόδοξοι, πολύ μαχητικοί και θα πρέπει να αλλάξουν και οι κανόνες του παιχνιδιού. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε και τη διαδικασία ψήφου με ειδική πλειοψηφία. Αυτό θα επιτρέψει να αλλάξουμε άρδιν τα πράγματα και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε εύλογα τα φορολογικά ζητήματα έτσι ώστε να μην αποδυναμωθούμε. Κάτι το οποίο θα γίνει αν δεν υπάρχει αυτή η φορολογική κυριαρχία. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα κεντρικό θέμα των ευρωεκλογών και η κάθε ε, ομάδα θα πρέπει να προωθήσει αυτή την ε, λύση σε όλο το πολιτικό φάσμα. Είμαι ρεαλιστής, ξέρω ότι χρειάζεται πολύς χρόνος και θα πρέπει να περάσουμε οπωσδήποτε από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία. Αυτό θα το δούμε και σε επίπεδο εκοφήν. Ήδη έχει γίνει μία πρώτη συζήτηση και θα γίνει και τις επόμενες εβδομάδες υπό Ρουμανική Προεδρία. Και ε, γνωρίζω ότι υπάρχουν επιφυλάξεις και αντιστάσεις όμως το Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε θέση υπέρ των πολιτών και να πιέσουμε τα κράτη-μέλη για να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όπως και να έχει η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταβάλουν κοινή προσπάθεια μέσα στα πλαίσια μίας γενικότερης μάχης και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να ασχοληθούν με αυτό το ζήτημα, να είναι το κύριο τους μέλημα για μια φορολογική δικαιοσύνη, ιδιαίτερα για την επόμενη θητεία. Θα είναι και η τελευταία μου ε, παρέμβαση επί του θέματος αυτού και είμαι πεπισμένη μετά από πέντε χρόνια κοινή εργασίας ότι αυτό είναι ένα ε, θέμα το οποίο σφυριλατεί μία ενότητα του, της επαύριων. Υπάρχουν ε, διαφορετικές ευαισθησίες αλλά μεγάλη πλειοψηφία που υποστηρίζει την έκθεσή σας. Πρόκειται για κοινό συμφέρον της Ευρώπης που μας ενώνει όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξαιρετική αυτή εργασία υπέρ της ε, διαφάνειας και της καταπολέμησης της ε, φοροδιαφυγής. Είναι μια κοινή μάχη που θα συνεχίσουμε από κοινού. Κύριε έχετε το λόγο. Έχετε τα τελευταία δύο λεπτά για αυτή την Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και του συναδέλφου για αυτή την πολύ καλή και ουσιαστική συζήτηση, την έκθεση αυτή και τον κύριο Νίτερ Μάγερ, τον συνεισηγητή μου, καθώ και όλα τα μέλη τη Επιτροπή ΤΑΞΕ 3 που εργάστηκαν τόσο σκληρά για το θέμα αυτό, για τα θέματα ε, τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Ευχαριστώ πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Επίτροπο Μοσκοβισή και ε, τον Επίτροπο που βρίσκεται επίση εδώ. Σα ευχαριστούμε για τη συνεργασία μα για τα θέματα τη καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή και τη φοροαπάτη τη ε, και στα πλαίσια τη Επιτροπή Τάξε. Για την φορολόγηση πρέπει να πω ότι καταφέραμε να περάσουμε 14 νέα νομοθετήματα σε αυτή τη θητεία. Όμω νομίζω ότι απομένουν πολύ περισσότερα να γίνουν σε ό,τι αφορά την δίκαιη φορολόγηση. Κύριε Επίτροπε Μοσκοβισή, έχετε απόλυτο δίκιο. Η Ευρώπη θα πρέπει να ανοίξει το δρόμο για τον 21ο αιώνα και να υπάρξει ένα σύστημα για τι εταιρείε που φορολογικά να είναι δίκαιο και για του πολίτε και για τα κράτη-μέλη όλα. Και δικαίω και για τι επιχειρήσει. Άκουσα στη συζήτηση σήμερα ότι το θέμα των μεγάλων ομίλων και των μεγάλων πολυεθνικών είναι θέμα για τον κύριο Κόρμπιν. Όμω και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποκαλύψει ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, θα πρέπει ε, να ε, έχουν ένα εισόδημα που είναι ανάλογο με αυτό των πολυεθνικών εταιριών. Θέλουμε να υπάρχει δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών. Θέλουμε να αντιμετωπιστεί η φορολογική αδικία. Και επίση, κατά τη διάρκεια των εργασιών μα, νομίζω είδαμε ότι δεν είναι κανεί αρκετά πλούσιο ή αν είναι μια εταιρεία αρκετά πλούσια και αρκετά μεγάλη ώστε να ε, ε, ε, ξεπεράσει τα όρια του νόμου, το κάνει. Δεν θα πρέπει να δεχόμαστε τέτοιου είδου πρακτικέ. Ω Κοινοβούλιο που εκπροσωπούμε το λόγο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αναλάβουμε δράση κατά των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Όπω είδαμε και με την αφορμή του σκανδάλου Panama Papers, δεν μπορεί κανεί να είναι υπεράνω του νόμου. Δεν μπορεί κανεί να υπερβαίνει το, δικαστικό σύστημα και τη δικαιοσύνη. Συνάδελφοι, λοιπόν, σα ευχαριστώ. Ε, ανυπομονώ για την ψηφοφορία αύριο, αλλά νομίζω ότι στο νέο Κοινοβούλιο θα πρέπει αμέσω να ξεκινήσει η σχετική δουλειά και να πιέσουμε όλε μα τι κυβερνήσει ώστε οι δραστηριότητέ μα να είναι όλε αντικείμενο λογοδοσία. Ευχαριστούμε κύριε Κόφοντ. Και τώρα η συζήτηση ολοκληρώνεται. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο και περνάμε στο επόμενο θέμα. Περνάμε στο επόμενο θέμα τη σημερινή ημερήσια διάταξη. Προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κατάσταση όσον αφορά το κράτο δικαίου και η καταπολέμηση τη διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω στη Μάλτα και στη Σλοβακία. Η κυρία Ιντβέλτ έχει πρώτο λόγο για πέντε λεπτά, καθότι είναι η συντάκτρια τη προφορική αυτή ερώτηση. Και θα έχουμε βέβαια μαζί μας και την Επίτροπο Γιούροβα, η οποία θα πάρει και αυτή το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ πολύ μην κάνετε θόρυβο. Ας ακούσουμε τους ομιλητές και κάντε οποιαδήποτε συζήτηση εκτός εθούσης. Κύριε Ενβέλτε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πραγματικά κρίμα που απουσιάζει σήμερα το Συμβούλιο. Προφανώ θα πρέπει να ήταν παρόν για να συμμετάσχει στη σημερινή συζήτηση. Προτού επισέλθω στι λεπτομέρειε του ψηφίσματο και τη προφορική ερώτηση, θα ήθελα καταρχά να σε επενθυμίσω για μία ακόμη φορά τι έδωσε όφηση έναυσμα στην όλη αυτή διαδικασία. Αναφέρομαι στην δολοφονία της Δάφνης Καρουάνα Γκαλίσια, καθώς επίσης και τον Γιάν Κούτσια και τη μνηστής του Μαρτίνα Κουσνίροβα. Θα πρέπει πάντα να λέμε τα ονόματά τους, δεν θα πρέπει ποτέ να τους ξεχάσουμε. Συζητάμε σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, την προφορική ερώτηση, καθώ επίσης και το σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο θα ψηφίσουμε λίγο αργότερα φέτος και το οποίο συντάχθηκε από κοινού με όλες τις πολιτικές ομάδες, με την συμμετοχή της ομάδας παρακολούθησης του κράτους δικαίου και αποτελεί το ψήφισμα αυτό απόρρια μιας δεκάμινης διαδικασίας επιτόπου επισκέψεων, συναντήσεων, ακροάσεων, τηλεδιασκέψεων με εκπροσώπους των κυβερνήσεων, της αστυνομίας, με γενικούς εισαγγελείς, με μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημοσιογράφους, με πολλούς άλλους συμμετέχοντες. Αν δούμε λοιπόν το κείμενο του ψηφίσματος ως έχει σήμερα, θα συνειδητοποιήσετε ότι εστιάζεται μένα στην Μάλτα και τη Σλοβακία, αλλά όχι αποκλειστικά στις χώρες αυτές. Τονίζει όντω από τη μία πλευρά ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές ανησυχίες για συγκεκριμένα κενά στην νομοθεσία, για συγκεκριμένα εμπόδια τα οποία έχουν παρουσιαστεί. Από την άλλη αναφέρεται και σε κάποιε θετικέ εξελίξει. Και νομίζω τα διδάγματα τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράξη λειτουργεί. Η επέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθά τελικά τα κράτη-μέλη να επανέλθουν στο σωστό δρόμο όταν κινδυνεύουν ουσιαστικά να βγουν από το σωστό δρόμο όσον αφορά το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα. Στο ψήφισμα γίνονται ορισμένες συστάσεις, οι οποίες συνοψίζονται άλλωστε και στην προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις προς την Μάλτα και τη Σλοβακία η μία από τι συστάσει αυτέ απευθύνεται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ουσιαστικά καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει έναν διάλογο για το κράτος δικαίου με τη Μάλτα. Κρίνουμε ότι ε, είναι δικαιολογημένο κάτι τέτοιο και παράλληλα βέβαια θα πρέπει να υποβληθούν και κάποιες τροπολογίες όπου θα λέγεται ότι αναγνωρίζουμε ως Ευρωβουλευτές ότι ε, η Μάλτα έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι θα πρέπει να διεξαχθεί και ένας διάλογος με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λέμε ακόμα ότι ε, θα πρέπει να συλληφθεί όχι μόνο ο υπέτειος ή η υπέτειοι, αυτοί δηλαδή που διέπραξαν τη δολοφονία της Δάφνης Καρό Αναγκαλίσια, αλλά και ο ηθικός αυτοργός, αυτός ο οποίος ζήτησε τη δολοφονία της. Λέμε επίση ότι θα πρέπει να ελεγχθούν καλύτερα και να σταματήσουν οι χρυσέ θεωρήσεις στη Μάλτα, τη Σλοβεκία αλλά και στις υπόλοιπες εμπλεκόμενες χώρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να διελευκανθεί περισσότερο η περίπτωση της δολοφονίας του Γιάν Κούτσιακ και της Μαρτίνα Κουσνίροβα και επίσης να έχουμε επίσημη καταδίκη του επίσημου υπετίου. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες ανησυχίες αυτή τη στιγμή ακόμα όσον αφορά το σύστημα αυτή, αυτό της μεταπίδησης από τη μία θέση στην άλλη, από θέσεις του ιδιωτικού τομέα στο δημόσιο τομέα και αντίστροφα. Άτομα τα οποία εξαφανίζονται κάποια στιγμή εμφανίζονται με άλλες ιδιότητες. Καλούμε επίσης την κυβέρνηση της Σλοβακίας να σταματήσει την παρεπόδηση της, του διορισμού των νέων δικαστών στο ανώτατο δικαστήριο και επίσης να ασχοληθεί περισσότερο με τον νόμο εκείνο που έχει να κάνει με την ελευθερία της έκφρασης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στα πλαίσια της ομάδας παρακολούθησης του κράτους δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνειδητοποίησαμε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο το ρόλο της Ευρωπόλη, η οποία αναλαμβάνει δράση μόνο όταν καλείται να κάνει κάτι τέτοιο από τα κράτη-μέλη, τα μα λένε ότι έτσι λειτουργεί η επικορικότητα. Ωραία αυτό, αλλά στην πράξη βλέπουμε ότι οι δημόσιε αρχέ πολλέ φορέ οι ίδιε ε, εμπλέκονται σε σφάλματα και παρατυπίε. Στην περίπτωση αυτή, τότε εμεί θα πρέπει σε Ευρωπαϊκή Ένωση να απευθυνθούμε στις αρχές αυτές και να δούμε πώς μπορούν να διορθωθούν τα κακό κείμενα. Διότι είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, μια πραγματική ένωση. Αν λοιπόν υπάρχει έστω και ένα κράτος μέλος το οποίο δεν εφαρμόζει τα, πρότυπα, τα πρότυπά μας και τις αρχές μας, τότε τροχο... Μπλοκάρεται όλο το σύστημα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν επίση ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει εκ νέου να δημοσιεύει την ετήσια έκθεσή τη όσον αφορά τη διαφθορά. Γιατί ε, η μέθοδο που χρησιμοποιεί τώρα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θεωρούμε ότι δεν είναι επαρκή. Ζητούμε επίση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίω από τον κύριο Τίμερμαν που απουσιάζει σήμερα να απαντήσει επιτέλου στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να έχουμε έναν συλλογικό μηχανισμό όσον αφορά το κράτο δικαίου, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα. Και βλέπω ότι ε, οι Spitzenkandidaten, ο κύριος Βέμπερ αλλά και ο κύριος Τίμερμαν δεν έχουν δεσμευτεί ακόμα προκειμένου να υπάρχει ένα συνολικός τέτοιο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να υπάρχει ένας μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σαφές, ε, τα, σαφή τα όσα είπατε. Κύριε Επιτροπέ, έχετε το λόγο. Ε, κυρία Γιουροβά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται πλήρω ε, την προσήλωση του Ευρωπαϊκού Βουλίου και τη Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι κοινέ ευρωπαϊκέ μα αρχέ θα την χάνουν σεβασμού. Η Κομισιόν έχει αναλάβει δράση, ξεκινώντα για πρώτη φορά την διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 τη συνθήκη σχετικά με τι ε, δράσει τη πολωνική κυβέρνηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκκίνησε την διαδικασία σε σχέση με τις δράσεις της Ουγγρικής κυβέρνησης. Η Κομισιόν χρησιμοποίησε τον ρόλο της ως θεματοφύλακα των συνθήκων, ε, ξεκινώντας μια σειρά διαδικασιών επί παραβάση που σχετίζονται με θέματα κράτους δικαίου. Όλα τα κράτη-μέλη παρακολουθούνται από την Κομισιόν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το 2019 ε, η έκθεση για την Σλοβακία υπογραμμίζει ιδιαίτερος ότι υφίστανται ε, εδώ και αρκετό καιρό ανησυχίες σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Δεν φαίνεται αυτά τα προβλήματα να έχουν αντιμετωπιστεί ως τώρα. Η έκθεση για τη Μάλτα του 2019 υπογραμμίζει ότι οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις δεν έχουν ακόμα εξασφαλίσει πλήρως την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, κάτι το οποίο ε, επιβεβαιώνει και η Επιτροπή της Βενετίας ε, του ΟΕΕ Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Το ευρωπαϊκό, ε, η, αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου επίσης έχει προβάλλει ως προτεραιότητα, την μάχη κατά της διαφθόρας. Αυτό είναι σημαντικό και για την οικονομία μας και για την κοινωνία μας. Από το 2015 η Σλοβενία έχει λάβει συστάσεις για αυτό ακριβώς το θέμα επανειλημμένως η Κομισιόν έχει ε, εκφράσει τις ανησυχίες της για ε, την λογοδεσία της ε, αστυνομίας καθώς επίσης και για τον μικρό αριθμό ποινικών διώξεων καθώς επίσης και για τη μη επαρκή προστασία των καταγγελόντων της λειτουργίας. Σε ό,τι αφορά την ε, Μάλτα. Ε, οι ενσυχίες μας αφορούν υψηλού επίπεδου υποθέσεις διαφθοράς ε, και στο επίπεδο της ανάξης και σε επίπεδο εκδίκασης. παρακολουθούμε την κατάσταση και με τις δύο αυτές χώρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου και την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, η Κομισιόν επιμένει να προστατεύεται η ελευθερία τη ε, έκφραση και η ελευθερία του τύπου. Οι δημοκρατίε μπορούν να επιβιώσουν μόνον αν οι δημοσιογράφοι μπορούν ε, να ασκούν τα καθήκοντά τους ελεύθερα, χωρίς να παρενοχλούνται, χωρίς να απειλούνται και χωρίς να δολοφονούνται επειδή κάνουν καλά τη δουλειά τους. Είναι σαφές ότι αυτοί που κρύβονται πίσω από τη δολοφονία της Δάφνης Καρόνα Γαρίσια, του Γιάνν Κούτσιακ και της ε, Μαρτίνα Κουσνίροβα πρέπει να ε, δικαστούν. Οι έρευνες το, της αστυνομίας ε, αποτελούν αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους αλλά τα κράτη-μέλη έχουν και υποχρεώσεις όταν διεξάγουν τέτοιου είδους έρευνες. Επίσης έχουν την υποχρέωση να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε η ελευθερία έκφρασης να μπορεί να ασκείται ε, χωρίς περιορισμούς. Πρόσφερα και στη Μάλτα και στη Σλοβακία την βοήθεια της Europol και της Eurojust και επαναλαμβάνω αυτή την προσφορά εδώ. Τώρα, Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα της ε, θεωρήσεων ε, για ε, ε, για το οποίο η, τον Ιανουάριο 2019 η Κομισιόν εξέδωσε μια σφαιρική έκθεση. Ως επόμενο βήμα προτείνουμε να δημιουργηθεί μια ομάδα εμπειρογνωμών από τα κράτη-μέλη για να διερευνήσει τους ενδεχόμενους κινδύνους που προκύπτουν από τα, ε, από το, από τα συστήματα χορήγησης χρυσών θεωρήσεων σε επενδυτές. Θα πρέπει να δούμε τι είδους έλεγχοι ασφαλείας θα πρέπει να γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις περίπτωση. Η Κομισιόν έχει στόχο τον Ιούνιο να υποβάλει μια πρωτοβουλία για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να προετοιμάσουμε αυτή μας την ανακοίνωση, σκοπεύουμε να υιοθετήσουμε ένα ανακοινωθέν για τη σημερινή κατάσταση και για τα ενδεχόμενα επόμενα βήματα για να ενισχυθεί το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να, να γίνει μια διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους και τα θεσμικά όργανα. Η απόψη και η εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι ιδιαίτερα σημαντική έτσι προκειμένου να τροφοδοτήσει αυτή τη μελλοντική πρωτοβουλία. Θα λάβουμε ε, γνώση και θα ε, λάβουμε υπόψη ε, το ψήφισμα του Κοινοβουλίου και υπ' αυτή την έννοια θα σκεφτούμε και προτάσεις που έχουν σχέση, θα εξετάσουμε προτάσεις που θα έχουν σχέση με ένα ενδεχόμενο μηχανισμό ε, αξιολόγηση από ομοτήμους σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Ευχαριστούμε. Περνάμε στους ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Πρώτα για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για 1,5 λεπτό η κυρία Μετσόλα. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι περήφανη για τη χώρα μου. Είμαι περήφανοι για το μαλτέζικο λαό και για το γεγονός ότι ανήκουμε σε αυτή την ένωση αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι περήφανη που προέρχομαι και κατάγομαι από μια πολύ μικρή χώρα που παρά το μικρό της μέγεθος έχει συμβάλει σημαντικά στην ιστορία της Ευρώπης. Αυτό μας καθιστά Μαλτέζους. Το μέγεθός μας δεν ήταν ποτέ εμπόδιο. Θεωρούμε ότι η γεωγραφία δεν μπορεί να μας εμποδίσει. Δουλέψαμε σκληρά και τα καταφέραμε και το κάναμε γιατί η αποφασιστικότητά μας προέρχεται από την ακαιρεότητά μας, από τον χαρακτήρα του μαλτέζικου λαού. Και πρέπει να αγωνιστούμε για να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας αυτή. Και μάλιστα ακόμη και ενάντια σε ανθρώπους που ε, επιβουλεύτηκαν την ταυτότητά μα. Ξέρουμε εμεί ότι είμαστε Μαλτέζοι, είμαστε Ευρωπαίοι. Οι Μαλτέζικε αξίε είναι ευρωπαϊκέ αξίε και πρέπει να είμαστε σαφεί. Η δολοφονία δημοσιογράφων δεν μπορεί να γίνει ποτέ ανεκτή. Η διαφθορά είναι φαινόμενο απαράδεκτο. Η ασυλία και η αδικία πρέπει να καταπολεμηθούν και να καταπολεμούνται πάντοτε. Αυτέ είναι οι αξίε που εγώ υπερασπίζομαι και προωθώ πάντοτε. Και αυτό είναι το πνεύμα του ψηφίσματος που συζητούμε σήμερα. Ακριβώς διότι περιγράφει τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Και αυτό θα κάνω και εγώ πάντοτε στην ε, διαδρομή μου. Εγώ συμμετέχω στην πολιτική γιατί έχω πεπιθήσεις και αρχές και θα συνεχίσω να το κάνω αυτό ε, μιλώντας εκ μέρους του μαλτέζικου λαού. Ο κύριος Βάιντεν έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με το ότι ε, για τη δημοκρατία προϋπόθεση είναι η ασφάλεια των πολιτών. Εμπιστοσύνη μπορεί να υπάρχει μόνο όταν τηρούνται οι κανόνες και ε, εμποδίζεται η διαφθορά και εξασφαλίζεται η ελευθερία της έκφρασης. Αυτό δεν ισχύει μόνο στο εσωτερικό κάθε χώρα, αλλά και στις εξωτερικές του σχέσεις μεταξύ των χώρων. Γι' αυτό και δεν μπορεί το ένα κράτος μέλος να παρεμβαίνει, να επεμβαίνει στην, ε, στις υποθέσεις άλλου κράτους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι ευρωπαϊκή υπόθεση. Είναι ευθύνη των κρατών μελών να κατανοήσουν σε βάθος αυτή την αρχή. ιδίω ε, στην περίπτωση της Πολωνίας ξεκίνησε η διαδικασία του άρθρου 7 ε, στη Μάλτα και στη Σλοβακία με τις ε, δολοφονίες των δύο δημοσιογράφων που διερευνούσαν υποθέσεις διαφθοράς έπληξαν την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στις δομές, τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές, αλλά και την δικαιοσύνη. Και εδώ το ερώτημα που αναδεικνύεται είναι αν πρόκειται για συστηματική παραβίαση του κράτους δικαίου ή όχι. Και στις δύο χώρες υπάρχουν πράγματι διαρθρωτικά προβλήματα. Στην περίπτωση της Μάλτας, μάλιστα, ε, πολλές φορές έχουν ε, ε, κατατεθεί και προτάσεις από την πλευρά της Επιτροπής, οι οποίες μάλιστα υλοποιούνται. Δυστυχώς όμως υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για το αν μπορούν να εξαχθούν ή αν έχουν εξαχθεί ε, βιώσιμα συμπεράσματα για την ελευθερία της έκφρασης, του τύπου και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Όμως δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να χάσουμε αυτή τη δυναμική. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή συνείδηση για το κράτος δικαίου. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική η θέσπιση ενός μηχανισμού για την εξασφάλιση των αρχών του κράτους δικαίου, όπως έχει ζητήσει επαναλημμένος το Κοινοβούλιο. Το ότι ε, για την Κομισιόν φαίνεται ότι αυτό δεν είναι τόσο σαφέ και το γεγονό ότι κάνει ένα μισό βήμα προ τα πίσω, θέλω εκ μέρου τη πολιτική μου ομάδα να δηλώσω ότι είναι πραγματικά αρνητικό φαινόμενο. Για το ECR, το λόγο έχει κύριε Ρόνονεν Λένερ Πύρκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σύμφωνα με την ε, διεθνή διαφάνεια, η Μάλτα και η Σλοβακία βρίσκονται σε πολύ χαμηλέ θέσει όσον αφορά την ε, διαφθορά. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η ερευνητική δημοσιογραφία στι χώρε αυτέ ακριβώ για να αναδεικνύονται τα προβλήματα. Σοκαρισμένοι όλοι μάθαμε τι δολοφονίε ε, δημοσιογράφων στη Μάλτα και στη Σλοβακία. Είναι σαφέ ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι δικαστικέ και αστυνομικέ έρευνε και να οδηγηθούν ε, οι υπεύθυνοι ηθικοί και φυσικοί αυτούργοι μπροστά στην, στην δικαιοσύνη. Υπάρχουν κέντρα και άτομα που θέλουν να μην ολοκληρωθούν οι έρευνες αυτές και στις δύο χώρες. Η Μάλτα, μάλιστα, προσπαθεί με τις ε, θεωρήσεις και τις άδειες ε, παραμονής, με το σύστημα των χρυσών θεωρήσεων, να ε, καταπολεμήσει αυτές τις έρευνες και αυτές τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει. Γι' αυτό και πρέπει να κατεργηθούν αυτά τα συστήματα. Ευχαριστούμε για τους πράσινους ο κύριος Γκίγκολτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η υποχώρηση όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου και την ε, τήρηση των, θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ορισμένα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά ανησυχητικό φαινόμενο. Είναι ένα χτύπημα στο, στην καρδιά τη Ευρώπη, διότι η Ευρώπη δεν αφορούσε ποτέ μόνο την μεγιστοποίηση των συμφερόντων των κρατών μελών, αλλά ήταν πάντοτε και μια κοινότητα αξιών. Το να εξασφαλίζεται λοιπόν η τήρηση των αρχών αυτών από όλα τα κράτη-μέλη είναι ύψη τη σημασία και γι' αυτό χρειάζεται να θεσπιστεί επιτέλου ένα μηχανισμό διεθνικό, ευρωπαϊκό, ο οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση σε όλε τι ε, χώρε μέλη μέσω μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων και να διαπιστώνει αν τηρούνται οι αρχέ δημοκρατία και του κράτου δικαίου. Αν τα κράτη-μέλη μάλιστα διαπιστώνεται ότι, αυτό, ε, ότι δεν τηρούν τι αρχέ αυτέ, θα πρέπει να υπάρχουν και αυτό θα πρέπει να ισχύει και στο πλαίσιο του επόμενου ε, δημοσιονομικού ε, πλαισίου. Όταν λοιπόν θα υπάρχουν σημαντικές σοβαρέ παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου, θα πρέπει οι αποφάσεις πλέον να μην μπορούν να λαμβάνονται αποκλειστικά από τις εθνικές αρχές, αλλά από τις αρχές Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ για την ΚΟΕ, η κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δική μας ε, κοινοβουλευτική θητεία κατέδειξε ότι η κατάσταση του κράτους ε, δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Ζούμε σε χώρες όπου δολοφονούνται δημοσιογράφοι οι οποίοι διεξάγουν έρευνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να συμβάλλουμε επικοδομητικά ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η παρακολούθηση όμως την οποία θέλουμε προϋποθέτει ότι ο ρόλος μας θα πρέπει να είναι εντελώς ουδέτερος. Ποτέ πολιτικός, ποτέ κομματικός θα πρέπει να έχει ως στόχο να τηρηθούν συγκεκριμένα πρότυπα, να επιβλωθούν κυρώσεις και ουσιαστικά να ενισχύσουμε όλες τις ε, διεργασίες εκείνες ε, οι οποίες μπορούν να στραφούν κατά οποιασδήποτε προσπάθεια καταστολή του κράτου δικαίου. Δυστυχώ δεν βλέπουμε τεχέγγυα αυτά στο ψηφίσμα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο δικό μα ο ρόλος να μπορεί να είναι πραγματικά αμετάκλητο, γιατί διαφορετικά ο κίνδυνο που διατρέχουμε είναι ότι τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσουν να λειτουργούν όλο και περισσότερο ω όργανα τα οποία προέρχονται από μυθιστορήματα του Orwell και ουσιαστικά θα καταφέρουμε ποτέ στην πράξη να επιβάλλουμε το κράτο δικαίου. Σα ευχαριστούμε εξ του FDD. Το λόγο κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα τα οποία στρέφονται κατά τη δημοκρατία, του κράτου δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ορισμένα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω τη Μάλτα και τη Σλοβακία. Και αυτό το έχει τονίσει επανειλημμένο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδωσαν την απαραίτητη συνέχεια στι δικέ μα ανησυχίε. Ζητάμε να δημιουργηθεί ένα μηχανισμό παρακολούθηση για τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, προκειμένου να μπορούμε να στρεφόμαστε κατάλογο αυτών των παραβιάσεων. Για άλλη μια φορά, ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επίτροπη να μα πει ποια μέτρα επιτέλου προτίθεται να υιοθετήσει προκειμένου να διασφαλιστεί η διάκριση των εξουσιών, η εξαρτησία του δικαστικού συστήματο, η καταπολέμηση διαφθορά, η ασφάλεια των δημοσιογράφων, η ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση ενημέρωσης Δυστυχώ ε, τα φαινόμενα αυτά τα αρνητικά δεν τα βλέπουμε μόνο στη Μάλτα. Και αναφέρομαι εδώ πέρα στι χρυσέ θεωρήσει όσον αφορά του επενδυτέ για την απόκτηση τη Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια ή τη άδεια διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι η Ιθαγένεια στην περίπτωση αυτή γίνεται ένα απλώ εμπορεύσιμο προϊόν προκειμένου να νομιμοποιηθεί, νομιμοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή ενα απλο παρουσία πολλέ στην ευρωπαικη εντελώ ε, παράνομων ε, στοιχείων και οντοτήτων. Νομίζω λοιπόν ότι η καταπολέμηση τη διαφθορά θα πρέπει να ενισχυθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω συγκεκριμένων νομοθεσιών. Θα πρέπει να παταχθεί το φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό το λόγο περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα μέτρα, Όπω τα μέτρα αυτά τα οποία πρόσφατα εγκρίναμε στην Ιταλία, προκειμένου να καταφέρουμε να πατάξουμε τη διαφθορά ακόμα και στα πλαίσια τη δημόσια διοίκηση και προκειμένου να υπάρχει μια απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να υποστηρίξω το ψήφισμα αυτό το οποίο δεν στρέφεται εναντίον των πολιτών της Μάλτας και της Σλοβακίας, το αντίθετο, ασκεί κριτική στις πρακτικές που ακολουθούν οι κυβερνήσεις στις δύο αυτές χώρες. Το ψήφισμα αυτό βασίζεται στις δημοκρατικές αξίες που θα πρέπει να τηρούν όλες οι κυβερνήσεις. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μου, τη Σλοβακία, πραγματικά σοκαριστήκαμε για το γεγονός ότι οδηγηθήκαμε σε δολοφονία ενός δημοσιογράφου και της ε, αραβωνιαστικιάς του. Πιο πολύ σοκαρισμένοι όμως ήμασταν όταν διαπιστώσαμε ότι η μαφία είχε επαφές με κυβερνητικούς αξιωματούχους και ότι ε, σχεδιάζονταν και προγραμματίζονταν δολοφονίες και άλλων σημενόντων ε, προσώπων της σλοβακικής κοινωνίας όπως για παράδειγμα εισαγγελέων ή και ε, του, υπουργού, του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης. Υπήρξαν λοιπόν σε όλη τη χώρα διαδηλώσεις Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους ενάντια στη διαφθορά και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακριβώς γιατί στέκεται στο πλευρό του λαού της Σλοβακίας. Θέλω να επισημάνω ένα στοιχείο ακόμη. Στην ε, Βουλή της Σλοβακίας, κατόπιν αιτήματος του, της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, το αίτημα μάλλον της Επιτροπής Αναφορών ε, αγνοείται ε, συστηματικά από την Βουλή της Σλοβακίας για το ζήτημα της συλλογικής ευθύνης. Μάλιστα, θέλω τη σχετική απόφαση που έλαβε η Βουλή της Σλοβακίας πρόσφατα να την ελέγξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σμόλκοβα. Ευχαριστώ πολύ. Αμέσως μετά τη τηλεφωνία Δυστυχώς χάσαμε ε, την βεβαιότητά μας ότι το δίκαιο πάντοτε ε, νικά. Αυτό ήταν και το ε, χειρότερο φαινόμενο. Όμως Υπάρχουν και κάποιες ε, χαραμάδες, κάποιες αχτίδες αισιοδοξία. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε πέντε άτομα σήμερα για τη δολοφονία του δημοσιογράφου. Ο πρόεδρος της χώρας μου πρόσφατα ε, μίλησε για το πόσο σημαντική ε, υπόθεση είναι η καταπολέμηση τη διαφθοράς. Η κυβέρνηση της Σλοβακία. Έχει υποβάλει μάλιστα και σχετική πρόταση για την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς η οποία βασίζεται στις συστάσεις και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Στόχος δεν είναι η διαφθορά, ε, η καταπολέμηση της διαφθοράς μόνο στη Σλοβακία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές είναι σαφή τα στατιστικά στοιχεία. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση χάνονται ένα δισεκατομμύριο ευρώ κατέτο από τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Πότε επιτέλου θα δοθεί ένα τέλο στου φορολογικού ε, παραδείσου, πότε επιτέλου θα δοθεί ένα τέλο σε αυτήν την κατάχρηση των χρηματοπιστωτικών κανόνων. Και έχω άλλα πέντε δευτερόλεπτα στη διάθεσή μου. Κυρία Επίτροπε, θέλω να σα ευχαριστήσω για την επίσκεψή σα στην ε, Σλοβακία. Κύριε Δεκόφσκι, κύριε Δεκόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επανειλημμένως έχω επισκεφθεί τη Μάλτα και τη Σλοβακία φέτος και πέρσι και με τρόμαξε ο, ο αριθμός των υποθέσεων στις οποίες αγνοείται η, εθνική νομο, η κοινωτική νομοθεσία. Οι πολίτες αυτών κρατών θέλουν να βοηθηθούν, να λυθούν τα προβλήματα για τα οποία έχασαν τη ζωή του αυτοί οι δημοσιογράφοι. Η διαφθορά, η μη λειτουργία του κράτους δικαίου συγκεκριμένα. Αυτά είναι τα προβλήματα και είναι γνωστά. Σε μην προσποιούμεθα πως δεν τα γνωρίζουμε. Εμείς θα πρέπει να είμαστε αυστηροί. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε. Δεν χρειάζεται απλώς να, να διερευνηθούν αυτά τα εγκλήματα, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να επικρατήσει το κράτος δικαίου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να στρέφει αλλού την κεφαλή όταν γίνονται τέτοιου είδους παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Ευχαριστώ. Σάντ, ένα μισή λεπτό. Το θέμα αυτό έχει χρησιμοποιηθεί για να προωθηθούν πολιτικά συμφέροντα Οι έρευνες αυτές έχουν ως ε, στόχο να μαυρώσουν τη φήμη του εις Μάλτας. Είναι αποτέλεσμα της δράσης της αντιπολίτευσης. Πώς είναι δυνατόν να προσποιούμεθα ότι μιλάμε το κράτος δικαίου. Πρόκειται για μια ομάδα μελών που δεν έχει καν εκλεγεί, έχει αυτοοριστεί εισαγγελέα και δεν έχει κανένα είδου δικαιοδοσία. Αυτή είναι που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή. Την ε, περασμένη Παρασκευή η κυβέρνηση της ε, Μάλτας δεσμεύτηκε να κάνει νομοθετικές αλλαγές σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας. Προσωπικά πιστεύω δεν χρειαζόταν καν να γίνει μια τέτοιου είδους γρήγορη ε, να λυθεί μια τέτοια είδηση, ίδια γρήγορη απόφαση. Θα έπρεπε το θέμα να συζητηθεί με τους Μαλτέζους και μετά να ληφθούν αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αυτή η απόφαση κυβέρνηση είναι σαφής ε, ένδειξη ότι ε, η Μάλτα σέβεται και θα σέβεται το κράτος δικαίου πλήρως. Ζητώ από όλους και όλες εσάς να αντιμετωπίσετε την πραγματικότητα με ειλικρίνη. Ευχαριστώ. Ο Καντέμοφ για ένα λεπτό господин госпожо Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Καταδικάζω απερίφραστα τα όσα συνέβησαν με τους δημοσιογράφους στις δύο αυτές χώρες, στη Σλοβακία και στη Μάλτα, είναι φαινόμενα απαράδεκτα, τα οποία στρέφονται ευθέως εναντίον των ευρωπαϊκών κανόνων και των ευρωπαϊκών αξιών. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά πρέπει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σταλεί ένα κατηγορηματικό μήνυμα καταδίκη, να ασκηθεί πίεση ώστε οι χώρε να ολοκληρώσουν τι έρευνε, να χυθεί άπλετο φω στι υποθέσει αυτέ, γιατί δεν μιλάμε μόνο για του φυσικού αυτούργου, αλλά και για του ηθικού αυτούργου, εκείνου που κρύβονται και που έδωσαν την εντολή για, την, ε, για τα εγκλήματα αυτά. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την ελευθερία των ε, δημοσιογράφων του τύπου και την τήρηση και την ε, προστασία των αρχών και των αξιών μας. Εγώ ε, δεν συμφωνώ με εκείνους που επιχείρησαν μάλιστα να εμπλέξουν στις, σε τέτοιου είδους υποθέσεις και τη Βουλγαρία, διότι στη Βουλγαρία δημοσιογράφοι δεν έχουν δολοφονηθεί. Και περνάμε στην ε, διαδικασία Κατσδιάη, ο κ. Φαρία για ένα λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση που βασίζεται στη δημοκρατία, στο κράτο δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δυστυχώ όμω, Αυτά είναι, αυτό είναι νεκρό γράμμα σε ορισμένα κράτη και κάποιοι ερευνητικοί δημοσιογράφοι πληρώνουν το τίμα με τη ζωή τους. Ε, πρόκειται για κράτη τα οποία χαρακτηρίζονται από καταχρήσεις και από διαφθορά και από διαφάνεια. Το ίδιο έγινε και με τον Γιάν Κούτσιακ, ο οποίος ερευνούσε τη διαφθορά σε υψηλόβαθμα στελέχη του κράτους. Το ίδιο και στην ε, Μάλτα με την κυρία Καρουάνα Γκαλίτσια για την οποία δεν ξέρουμε ποιοι ήταν η πραγματική ηθική ευτουργή ακόμα. Όλα αυτά αναγκα... φημώνουν τον τύπο. Ε, η αιτία είναι η αδυναμία καταπολέμησης της ε, διαφθοράς ε, και η, ανεξέλεγκτη, η ανεξέλεγκτη λειτουργία της αστυνομίας. Επίσης, το σύστημα χρυσών θεωρήσεων αποτελεί δυνατότητα ε, νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων. Ευχαριστώ. το Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να ψηφίσουμε για το ψήφισμα αυτό αυτή την εβδομάδα, λέγοντας βέβαια ότι η Μάλτα δεν ενδιαφέρεται για το κράτος δικαίου. Τραγική ηρωνία όμως ότι το δικό μας το Κοινοβούλιο επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα ζητήματα, γνώντα όμω αυτή τη στιγμή ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία νομοθετεί αυτή τη στιγμή ακολουθώντα τι συστάσει τη Επιτροπή τη Βενετία. Υπάρχουν συγκεκριμένε προτάσει αυτή τη στιγμή που εξετάζονται από το Κοινοβούλιο μα και δυστυχώ το ψήφισμα αυτό που θα εγκρίνουμε σε αυτή την εβδομάδα δεν αντικατοπτρίζει σωστά την κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή στην χώρα μου, τη Μάλτα. Πολλά πράγματα έχουν γίνει, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, έχουμε προχωρήσει σε συγκεκριμένε μεταρρυθμίσει, έχουμε κάνει σε ε, συνταγματικέ επίση τροποποιήσει για τι οποίε απαιτούνται τα δύο τρίτα τη πλειοψηφία στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Δυστυχώ όμω το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν αναγνώρισε όλε αυτέ τι προσπάθειε που κάνει η δικιά μου η χώρα. παρακολουθούμε από πολύ κοντά τα όσοι συμβαίνουν στη χώρα μου ε, με το θέμα των ε, καταγγελών των δυσλειτουργίες οι οποίοι δεν προστατεύονται αρκετά. Δεν είναι δυνατόν από την άλλη μεριά στη Μάρτα να μην έχουν συλληφθεί ακόμα οι ηθικοί αυτούργοι της δολοφονίας της κυρίας ε, Καρουάνα Γκαλίσια. Η έρευνα έχει μπλοκαριστεί από τον Πρωθυπουργό τον κύριο Μουσκάτ. Καθώ επίση και από το Γενικό Εισαγγελέα και την αστυνομία. Δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών στη Μάλκα και βλέπουμε τα προβλήματα. Ε, μακάρι να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσει. Θα πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε η αυτοργοί του, της δολοφονίας του Γιάννη, τη Μαρτίνα και της Δάφνη να έρθουν στο δικαστήριο. Είναι αδύνατον, είναι απαράδεκτο ο Πρωθυπουργό της Μάλτας να εξακολουθεί να προστατεύει τα ονόματα ε, που προέκυψαν από, τα, ε, από το σκάνδαλο του Παναμά και να, μη, και να μπλοκάρει τις έρευνες που γίνονται για να διαλευκανθεί η δολοφονία της κυρίας Καρουάνα Γκαλίσια. Ο πρόεδρος διακόπτει την κυρία Γκόμες. Your... Σας παρακαλώ πολύ κυρία Γκόμες, δείξτε λίγο σεβασμό στους υπόλοιπους συναδέλφους που θέλουν να λάβουν το λόγο. Η κυρία Ντάλι ε, έχει μια μπλε κάρτα, τη δέχεστε. Ναι, κυρία Ντάλι, έχει το λόγο. Μια και αναφέρθηκε σε μένα, Γκόμε, σε έναν τρόπο που δεν κατάλαβα πολύ καλά. Θα μπορούσε να μου πει, συνάδελφο, εσείς είστε εναντίον αυτών των μεταρρυθμίσεων. Για πέστε μα κυρία Γκόμε. θα ήθελα να γίνουν μεταρρυθμίσει που θα οδηγήσουν διάκριση των εξουσιών και στην ε, εμπέδωση του κράτους δικαίου. Επειδή δεν υπάρχει το κράτο δικαίου αυτή τη στιγμή, έχουν μπλοκαριστεί οι έρευνε για την δολοφονία τη κυρία Καρουάνα Γκαλίσια. Αυτό είναι τρομακτικό και δυστυχώ ο πρόεδρο διακόπτει την ομιλήτρια. Έχετε πολλά να πείτε μία στην άλλη, οπότε ενδεχομένω θα μπορούσατε να τα πείτε εκτό τη αιθούση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Είναι η δεύτερη έκθεση που συζητούμε σχετικά με την κατάσταση στην Σλοβακία. Όπως και στην προηγούμενη συζήτηση που είχε γίνει εδώ στο Κοινοβούλιο, θέλω να επαναλάβω την οδύνη μου για τους θανάτους των δύο δημοσιογράφων, της κυρίας Γκαλίτσια και του Ιωκούτσιακ. Όμως νομίζω ότι η έκθεση αυτή πραγματικά έχει συγκεκριμένο πολιτικό χαρακτήρα και στόχευση. Γιατί εγώ βρισκόμουν με την, σε συνεχή ε, επαφή με την συγγήτρια δίνοντας τις, τροφοδοτώντας τις με στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν στην έκθεση, δεν αναφέρονται πουθενά. Ε, στην Σλοβακία έχουν γίνει συγκεκριμένε κινήσει, έχουν αναλυφθεί συγκεκριμένε πρωτοβουλίε διαρθρωτικέ και έχουν αποδοθεί και ευθύνε και κατηγορίε. Πραγματικά ε, λυπάμαι για τις αποκλήσεις που υπάρχουν ε, και που διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ανάμεσα στην Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη. Κάθε μήνα έχουμε την ίδια ιστορία. Οι Δυτικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγορούν τις ανατολικές χώρες ότι δεν ακολουθούν τις αρχές του κράτους δικαίου. μπλε κάρτα από την κυρία Πολύ ωραία, Ινβέλτ. Κύριε Ινβέλτ, έχετε το λόγο. Λοιπόν, άκουσα τι επικρίσει σα. Τι έχω ακούσει και στο παρελθόν. Νομίζω ότι δεν είναι βάσιμε. Δεν επρόκειτο να αντιδράσω, αλλά πραγματικά θα ήθελα να διευκρινίσετε την τελευταία σα δήλωση. Είπατε ότι το ψήφισμα αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχει μια, ένα χάσμα μεταξύ Ανατολική και Δυτική Ευρώπη. Εγώ πάντα έλεγα ότι δεν υπάρχει Δυτική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, Βόρεια, Νότια Ευρώπη. Μία και μοναδική ενιαία Ευρώπη υπάρχει. Και γι' αυτό εργάζομαι τελευταία 15 χρόνια. Δεν δέχομαι δήλωσή σας. Κυρία Μπένοβα, έχετε μισό λεπτό για να απαντήσετε. Ναι, θα απαντήσω πολύ απλά. Εγώ τα όσα είπα τα είπα στο πλαίσιο του γεγονότος ότι κάθε μήνα ασκείται κριστική σε κάποια χώρα της ε, Ανατολικής Ευρώπης. Βουλγαρία, Ρουμανία, Τσεχία, Πολωνία, ε, σε κάθε σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τίθεται στο στόχαστρο μία χώρα από την Ανατολική Ευρώπη. Ε, αυτό δεν δείχνει συνεργασία. Μιλήσατε για την καπτολέμηση της ε, διαφθοράς. Πριν από σύντομο χρονικό διάστημα είχαμε μιλήσει για τις ε, κάτω χώρες όπου μια χώρα όπου υπάρχουν άλλωστε τα δεδομένα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η Σλοβακία και η Μάλτα είναι δύο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολίτες του εκπροσωπούνται εδώ, αξίζει να τις σεβόμαστε. Όμως κανένα κράτος μέλος από μόνο του δεν ε, μπορεί να ε, ισχυριστεί ότι μπορεί να αποφύγει τον αγώνα κατά της διαφθοράς που ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειάζεται λοιπόν ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Εδώ έγιναν δύο δολοφονίες δημοσιογράφων. Αυτό καταδεικνύει ότι αυτές οι δύο χώρες θα πρέπει να κάνουν το καθήκον τους προκειμένου να διελευκανθούν αυτές οι υποθέσεις για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δημοσιογράφων. Και η καταπολέμηση της διαφθοράς σημαίνει ότι θα πρέπει να, σταματήσουν, να σταματήσει η εφαρμογή των συστημάτων χρυσή ε, θεώρησης διότι ε, αποτελούν, αποτελεί αυτό το σύστημα παράθυρο στην ε, ε λεύκανση παράνομου χρήματο. και θα πρέπει να προστατεύσουμε τους καταγγέλτες, τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος όταν καταγγέλουν ε, περιπτώσεις διαφθοράς. Η Μάλτα και η Σλοβακία λοιπόν θα πρέπει να διαλευκάνουν αυτές τις υποθέσεις το συντομότερο. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Ήταν πολύ σημαντική συζήτηση αυτή γιατί πραγματικά κάλυψε διάφορα κρίσιμα ζητήματα. Αναφερόμαστε εδώ πέρα στο κράτο δικαίου. Μιλήσαμε για την ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση. Δεν μιλήσαμε όμω τόσο πολύ για το ότι θα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητο χώρος για την ενεργοποίηση τη κοινωνία των πολιτών, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ίδιου ζητήματο. Και κάθε φορά που βλέπουμε ότι επιδεινώνεται η κατάσταση σε ορισμένα κράτη-μέλη, βλέπουμε ότι πολύ συχνά επιδεινώνεται και στου τρει αυτού πυλώνες η κατάσταση. Δεν θα ήθελα Μάλλον θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο στο ζήτημα του κράτου δικαίου και στου μηχανισμού που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να παρακολουθήσει την κατάσταση του κράτου δικαίου στα κράτη-μέλη. Όπω είπα πριν από λίγο, χρησιμοποιούμε το σύνολο τη διαθέσιμη εργαλειοθήκη. Όλα τα διαθέσιμα δηλαδή μέσα τα οποία έχουμε. Για πρώτη φορά κινητοποίησαμε το άρθρο 7 καλύψαμε το σημαντικό αυτό ζήτημα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Χρησιμοποιούμε διαδικασία επί παραβάση όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Και επίση χρησιμοποιούμε και κάτι το οποίο δεν το είπα πριν από λίγο, το ότι έχουμε τον πίνακα αυτό αποτελεσμάτων όσον αφορά το δικαστικό σύστημα. Ξέρετε ότι σε αιτήσια βάση γίνεται μια συγκριτική αξιολόγηση. Έχουμε ένα πίνακα αποτελεσμάτων, βάσει του οποίου βλέπουμε πώ οι πολίτε αλλά και επιχειρήσει σε όλε τι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν ή εκτιμούν την εξαρτησία του δικαστικού του συστήματο. Και βέβαια, πέρα από αυτό, προσπαθούμε να προσθέσουμε και νέα κριτήρια για την καταπολέμηση της διαφθοράς, για το πώς αυτή λαμβάνει χώρα στα κράτη-μέλη. Χρησιμοποιούμε λοιπόν όλα τα μέσα που έχουμε στην εργαλειοθήκη μας. Να πω κάποια πράγματα όσον αφορά τις νέες πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω είπα και στην αρχική μου παρέμβαση, προβλέπουμε μια νέα ανακοίνωση για το κράτο δικαίου, προκειμένου να αποσαφηνίσουμε τι εννοούμε με το κράτο δικαίου, ότι ε, το κράτο δικαίου δεν είναι αποκλειστικό ζήτημα μόνο των κρατών μελών, αλλά ότι είναι και ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και ότι μάλιστα καλύπτεται και από την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νομολογία αυτή θα αντικατοπτρίζεται πλέον πλήρω στην νέα ανακοίνωση που θα κάνουμε για το κράτο δικαίου. Μια άλλη πρωτοβουλία μα τώρα έχει να κάνει με τη διασύνδεση του κράτου δικαίου με τον νέο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα πρέπει να το θίξουμε. Εγκρίναμε μια νέα πρωτοβουλία για την προστασία των καταγγελόντων και τέλος, αλλά σημαντικό, έχουμε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της από το 2020 και μετά. Και αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική συμβολή για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος ιδίως όσον αφορά για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλε αυτέ τι περιπτώσει πρέπει να ενισχύσουμε την ένωμη τάξη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ελοποιηθούν όλε αυτέ οι πρωτοβουλίε και θα πρέπει να εξηγήσουμε στου Ευρωπαίου πολίτε για ποιο λόγο αναλαμβάνουμε αυτή τη δράση, για ποιο λόγο οι πρωτοβουλίε αυτέ είναι τόσο σημαντικέ. Αναφέρθηκα πριν από λίγο στην ανάγκη να υπερασπίσουμε το κράτος δικαίου, και να υλοποιήσουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα όμως, ως πολίτης της τσεχικής δημοκρατίας θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι τις απόψεις σας και ότι θα πρέπει πραγματικά να εμπιστευόμαστε περισσότερο τους πολίτες που ζουν στις χώρες μας, οι οποίοι λειτουργούν δημοκρατικά, οι οποίοι έχουν να προτείνουν τρόπους επίλυσης των προβλημάτων. Θα πρέπει και προς αυτούς να εκφράσουμε την εμπιστοσύνη μας και γι' αυτό το λόγο είπα πριν από λίγο ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε και να εμπιστευτούμε όλο και περισσότερο τι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών. Ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε όλου εκείνου του πολίτε μα που είναι ακτιβιστέ, οι οποίοι ορθώνουν το ανάστημά του και οι οποίοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά του κάθε φορά που κάτι δεν πηγαίνει καλά στη χώρα τους. Δεν λέω ότι θα πρέπει οι άνθρωποι να κατεβούν στους δρόμους, δεν λέω ότι θα πρέπει να επαναστατήσουν, λέω ότι θα πρέπει να εμπιστευόμαστε λίγο περισσότερο τους πολίτες που ζουν στα κράτη-μέλη μας, γιατί είναι δημοκράτες και γνωρίζουν πώς θα πρέπει να κινούνται τα πράγματα. Και βέβαια θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν και στις εκλογές και να ψηφίζουν, να υποστηρίζουν συγκεκριμένε δημοκρατικές δυνάμεις. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Η ψηφοφορία θα γίνει την Πέμπτη. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση της κυρίας Μαρίτα Ουλφσκοκ σχετικά με τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών τη ώρας. Να ζητήσω λοιπόν από την κυρία εισηγήτρια να λάβει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ. Ε, ε Eh, eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε λίγες μέρες θα αλλάξουμε για άλλη μια φορά τα ρολόγια μας για να βάλουμε την ε, θερινή ώρα. Θα είναι η δεύτερη φορά το τελευταίο εξάμεινο που θα έχουμε αλλάξει την ώρα μας. Και αυτή η αλλαγή της ώρας και των ρολογιών μας που την κάνουμε κάθε εξάμεινο εδώ και αρκετές δεκαετίες, σκοπός αυτής της διαδικασίας όταν θεσπίστηκε ε, ήταν να εξοικονομείται ενέργεια. Αυτό όμως δεν ισχύει πια. Η νέα τεχνολογία σε διάφορους ε, τομείς της ζωής σημαίνει ότι τελικά δεν εξοικονομούμε τίποτα πια με τις αλλαγές της ε, ώρας. Εγώ ξέρετε ότι είμαι ευρωβουλευτής ε, εδώ και 10 χρόνια και τα χρόνια αυτά έχω λάβει μεγάλο αριθμό επιστολών, email και έχω κάνει πολλές συζητήσεις με πολλούς πολίτες για πάρα πάρα πολλά θέματα. Υπάρχει όμως ένα θέμα το οποίο επανέρχεται διαρκώς και αυτό είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν αισθάνονται καλά όταν αλλάζει η ώρα οι άνθρωποι επηρεάζονται με διάφορους τρόπους. Κάποιοι χαλάει ο ύπνος τους, κάποιοι αντιδρούν πολύ άσχημα και υπάρχουν και πολύ ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, τα, νέα, τα πολύ μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς, καθώς και εκείνοι που έχουν φυσικά ή ψυχολογικά προβλήματα και που επηρεάζονται από αυτές τις, από αυτές τις αλλαγές της ώρας. Στη βάση όλων αυτών λοιπόν είναι πέρα για πέρα βάσιμο να επανεξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους ε, κάνουμε αυτές τις αλλαγές της ώρας. Διότι φαίνεται ότι τελικά για πάρα πολλούς ανθρώπους οι επιδράσεις, οι επιπτώσεις αυτής της ε, πρακτικής είναι αρνητικές. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από πρωτοβουλίες πολιτών σε πολλές ε, χώρες μέλη αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ακούσει ε, πάρα πολλούς πολίτες για το ποιε είναι οι σκέψεις τους, ποια είναι τα συναισθήματά τους και πραγματικά δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα που να κινητοποιεί τόσο πολύ τους Ευρωπαίους πολίτες, τους απλούς Ευρωπαίους πολίτες που ακόμη και εκείνου που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με την πολιτική, όσο αυτό το θέμα τη αλλαγή τη ώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποστείλει επιστολέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν, κάνει, ε, που έχουν συμμετάσχει σε διαβουλεύσεις και έρευνε τι οποίε διεξήγαγε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκατομμύρια άνθρωποι λοιπόν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα τη Επιτροπής και έδωσαν τι δικέ του απαντήσει. Ε, αυτές τις απαντήσεις λοιπόν πρέπει να τι εκτιμήσουμε και να τι αξιολογήσουμε. Την τελευταία χρονιά λοιπόν ε, επεξεργάστηκα μια πρόταση σχετικά με την κατάργηση της εποχικής αλλαγής της ώρας. Η έκθεση αυτή ε, έχει εγκριθεί με ψηφοφορία σε 7 κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάτι που αποδεικνύει και πώς είναι οι τομείς που πραγματικά επηρεάζονται από αυτήν την αλλαγή της ώρας. Η πρότασή μας πλέον είναι να καταργηθεί η εποχική αλλαγή της ώρας το φθινόπωρο του 2021. Κάτι που θα δώσει ε, και την εμπιστοσύνη στους πολίτες ότι τους ακούμε και θα δώσει και ε, επαρκή χρόνο σε εκείνους που επηρεάζονται ώστε να κάνουν τις αναγκαίες προσαρμογές και η εσωτερική αγορά βεβαίω χρειάζεται χρόνο για να κάνει τι σχετικέ αλλαγέ για να μην υπάρξουν αρνητικέ επιδράσει από την ε, κατάργηση τη εποχική αλλαγή τη ώρα. Πρέπει όλα αυτά να γίνουν οργανωμένα για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τη εσωτερική αγορά και όλων των κλάδων που θα επηρεαστούν. Από την κατάργηση αυτή, με την κατάργηση αυτή, τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, πάρουν μια θέση για το ποια θα είναι η μόνιμη ώρα που θα επιλέξουν. Και αυτή η διαδικασία λοιπόν θα πρέπει να διακρίνεται από συντονισμό και συνεργασία. Δεν θα πρέπει να υπάρξει ένα μοσαϊκό στο τέλο τη όλη διαδικασία, να μην υπάρχουν διάφορε ε, ώρες, ε, ζώνες ώρας σε κάθε ε, κράτο μέλο. Εγώ θα έλεγα λοιπόν να υπάρξει μια συνεργασία, ένα συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και να ενημερώσουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη αλλά και την Επιτροπή έω το τέλο του 2020 για το τι θέλουν να κάνουν. Καλώς ήρθατε, Επίτροπε Μπούλτς. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέρη. Μέλη, συγγνώμη. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγητήρα, την κυρία Ολτσκοκ, τους κοιόδης εισηγητές και τα μέλη των έξι επιτροπών που εξέτασαν και υιοθέτησαν γνωμοδοτήσεις για την πρόταση της Κομισιόν. Όπως γνωρίζετε, η Κομισιόν αποφάσισε πέρσι να προτείνει την ε, διακοπή της, ε, των εποχιακών αλλαγών της ώρας, των εποχικών αλλαγών της ώρας ως ε, ανταπόκριση σε εκκλήσεις του Κοινοβουλίου, πολλών κρατών μελών και πολλών επίσης πολιτών που έστειλαν επιστολές σε εμένα και σε άλλους επιτρόπους κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Τα επιστημονικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι η αιτιολόγηση των εποχικών αλλαγών που ίσχυε παλιότερα δεν ισχύει πλέον. Είναι επίσης σαφές ότι η διακοπή, ο τερματισμός των εποχικών αλλαγών θα διευκόλυνε τη ζωή των ανθρώπων και θα αντιμετώπιζε και κάποια προβλήματα υγείας τα οποία σχετίζονται με το ισχύον σύστημα. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που διοργάνωσε η Κομισιόν είναι σαφή, ξεκάθαρα. 4,6 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ανταποκρίθηκαν, εκ των οποίων το 84% στηρίζει την πρόταση τερματισμού των εποχικών αλλαγών της ώρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την στήριξη της Επιτροπής ε, Τραν και του εισηγητή <clears throat> για να τερματιστεί η εποχική αλλαγή της ώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δύο φορές το χρόνο. Η Κομισιόν, όπως γνωρίζετε, σκοπίμως ήταν πάρα πολύ φιλόδοξη και <clears throat> είχε προτείνει να γίνει φέτος η τελευταία εποχική αλλαγή της ώρας. Όμως, δεδομένου ότι το Συμβούλιο δεν έχει λάβει ακόμα θέση, δεν είχε λάβει ακόμα θέση, καταλαβαίνουμε ότι είναι αδύνατο να τηρηθεί αυτή η προθεσμία. Γι' αυτό το λόγο σημειώνω την έκθεσή σας και τη θέση σας που είναι υπέρ του τερματισμού των εποχικών αλλαγών της ώρας το 2021. να σχολιάσω και μέσα από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και τις οποίες ε, βλέπουμε, ε, θεωρούμε ότι είναι λίγο πιο δύσκολο να δεχτούμε. Προτείνεται να δημιουργηθεί ένα καινούριο δίκτυο συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και της Κομισιόν ε, προκειμένου να συζητάτε από κοινού και να αξιολογείτε η απόφαση του κάθε κράτους μέλους ό,τι αφορά την ε, ε, ώρα του ε, και τις επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά. Και αν η Κομισιόν θεωρεί ότι η επιλογή ενός κράτους μέλους θα επηρεάσει υπερβολικά την εσωτερική αγορά, το κράτος μέλος θα έχει την υποχρέωση να υπερασπίσει τον εαυτό του και να εξηγήσει πώς θα αντιμετωπίσει αυτές τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες. Εμείς ε, ω Κομισιόν ε, πιστεύουμε ότι πράγματι χρειάζεται επαρκή συντονισμό μεταξύ των κρατών μέλων, όμω, η επιλογή της ε, ζώνης ώρας και της πραγματικής ώρας δεν, κάθε κράτος μέλους δεν είναι αρμοδιότητα της Κομισιόν. Αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Η Κομισιόν δεν μπορεί να στηρίξει ε, νομικές διατάξεις ε, προς αυτήν την κατεύθυνση, διότι αυτό θα σήμαινε ότι θα παρεμβαίνει σε αρμοδιότητα των κρατών μελών για τον καθορισμό της επίσημης ώρας τους. Δεν θα σεβόμασταν με αυτόν τον τρόπο την αρχή της επικορικότητας. του. λεχθέντος. Να σας βεβαιώσω ότι γνωρίζω πως από τις, από τις συζητήσεις μου με τα κράτη-μέλη ότι όλα αναγνωρίζουν την ανάγκη μιας συντονισμένης προσέγγισης και είμαι σίγουρη ότι θα επιλέξουν την επίσημη ώρα τους με τρόπο συντονισμένο και υπεύθυνο. Κανείς ε, δεν θέλει να δει μπαλώματα ε, διαφορετικής ώρας μέσα σε νησίδες διαφορετικής ώρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, επίσης, ζητάτε να μπορούμε να αναβάλουμε τον τερματισμό μέσω κατεξοδότηση πράξεων. Όμως ε, η θέση σε ισχύ ε, της απόφασης αυτής ε, είναι ουσιαστικό σημείο και δεν μπορεί να τροποποιηθεί με κατεξοδότηση πράξης. Αυτά ήθελα να πω. Περιμένω να, δω, να ακούσω τη συζήτηση και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει τη θέση του πριν την διακοπή των ρασιών του. Αυτό θα στείλει ισχυρό μήνυμα προς το Συμβούλιο ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο και πρόθυμο να προωθήσει αυτή την πρόταση με τρόπο που να οδηγήσει σε επιτυχία. Ευχαριστώ. Uh, Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Πιέκα για ένα λεπτό το νόματος Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλουμε αυτή τη στιγμή να καταργήσουμε μία οδηγία και στέλνουμε κατά αυτόν τον τρόπο ένα πολύ χειρό μήνυμα και ένα πολιτικό μάλιστα μήνυμα θα έλεγα γιατί η κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράστηκε ξεκάθαρα. Είπε ότι δεν θέλει πλέον να συνεχίζεται η εποχική αλλαγή της ώρας. Και τίθεται παράλληλα και ένα οικονομικό ζήτημα. Δεν θα ασχοληθώ όμω με αυτό, γιατί τα οικονομικά ζητήματα, ξέρετε, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα, ιδίω όσον αφορά την ενιαία αγορά και άλλου τομεί τη οικονομία. Θα ήθελα παρόλα αυτά να σταθώ περισσότερο στις ε, πτυχές που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, όλες οι έρευνες που έχουν γίνει για τον βιορυθμό, για την λεγόμενη χρονοβιολογία, αναφέρονται στις επιπτώσεις, στις πολύ σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εποχική αλλαγή της ώρας. Λέγεται ότι αυξάνεται επίσης κατά αυτόν τον τρόπο και ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων. Επομένω, ασχοληθήκαμε με το ζήτημα αυτό εμεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντο και είπαμε ότι θα πρέπει το στομότερο δυνατό να καταργηθεί η εποχική αλλαγή τη ώρα και ουσιαστικά να καταργηθεί η υφιστάμενη οδηγία η οποία προβλέπει την εποχική αλλαγή τη ώρα. Στηρίζουμε λοιπόν εμεί την πρωτοβουλία αυτή για την κατάργηση τη οδηγία και λέμε βέβαια ότι είναι τα κράτη-μέλη αυτά τα οποία θα πάρουν την τελική απόφαση, θα πρέπει να καταφέρουν να αποφασίζουν αυτά για την επίσημη ώρα τους, αλλά θα πρέπει βέβαια η ώρα αυτή έπειτα να είναι εναρμονισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστούμε πολύ για την Επιτροπή Βιομηχανίας τώρα έχει ο κύριος Σούλτς για ένα λεπτό παρακαλώ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Υπάρχουν σίγουρα πιο σημαντικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών. Παρ' όλα αυτά, σε ε, συλλογή υπογραφών που έγινε στο διαδίκτυο, πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ε, ε, συνυπέγραψαν υπέρ αυτής της κατάργησης της εποχικής αλλαγής. Και εμείς λοιπόν ως Επιτροπή, στην Επιτροπή Βιομηχανίας δηλαδή, υπερψηφίσαμε την πρόταση τερματισμού των εποχικών αλλαγών της ώρας. Το ότι αυτό δεν θα γίνει άμεσα, αλλά το 2021 μόλις, θεωρώ ότι είναι αρνητικό. Όμως από άποψη βιομηχανίας υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να γίνει κάτι τέτοια. Για παράδειγμα στην αεροπορία, όπου υπάρχουν τα time slots, οι χρονοθυρίδες που έχουν τεθεί σε διαπραγμάτευση πολλές φορές χρόνια πριν. Γι' αυτό και δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια βιαστική αλλαγή. Πλέον το θέμα δεν είναι στα χέρια ούτε της Κομισιόν ούτε του Κοινοβουλίου αλλά στα χέρια των κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει ένα μοσαϊκό διαφόρων ρυθμίσεων και κανόνων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνα θα πρέπει να εξασφαλίσουν αυτό το στόχο, γι' αυτό και τα καλό να ενεργήσουν γρήγορα με βάση τη βούληση που έχουν εκφράσει οι πολίτε μέσα από τι πρωτοβουλίε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίω η Κομισιόν. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστούμε εξ τώρα τη Επιτροπή Εσωτερική Αγορά. Το λόγο έχει ο κύριο Σόλτε. Για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κυρία Επίτροπε. Πολύ συχνά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συζητήσει το ζήτημα αυτό και προφανώς δεν είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στην Ευρώπη ή στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό για όλες αυτές τις πτυχές που έθιξαν οι συνάδελφοι. Δημόσια υγεία, οικονομική πτυχή και πολλές άλλες πτυχές τις οποίες ε, ακούσαμε πολύ συχνά στις συζητήσεις που γίνανε πρόσφατα. Η Επιτροπή τώρα Εσωτερική Αγορά γνωμοδότησε για το ζήτημα αυτό και στα πλαίσια τη γνωμοδότηση είπαμε ότι υποστηρίζουμε την κατάργηση τη εποχική αλλαγή τη ώρα, ωστόσο όμω λέμε ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε όλε τι επιπτώσει μια τέτοια κατάργηση, γιατί θα έχουμε πολλέ επιπτώσει σε πολλού τομεί. Στον τομέα των μεταφορών, για παράδειγμα, αλλά και σε άλλου συναφεί οικονομικού τομεί. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο χρειαζόμαστε ένα παρέτο χρονοδιάγραμμα, μια ευελιξία χρόνου, προκειμένου να καταφέρουμε όλοι να προσαρμοστούμε σε αυτή την αλλαγή. Και προφανώ θα πρέπει να κάνουμε κάθε τι το δυνατό, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση στα πλαίσια τη εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι νέες ρυθμίσεις για την ώρα να μπορούν να έχουν και τον απαραίτητο βαθμό προβλεψιμότητα. Σα ευχαριστούμε, κύριο Μιούλερ. Έχει το λόγο εξ Επιτροπή Γεωργία. Η κυρία Μιούλερ, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ω συγγήτρια τη Επιτροπή Γεωργία, θεωρώ ότι είναι ιδίω πολύ σημαντικά τα εξή σημεία. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχουν τρει ε, ζώνε ώρα και επιστημονικέ μελέτε αποδεικνύουν ότι η ετήσια αλλαγή τη ώρα έχει επιπτώσει στην υγεία, στο βιορυθμό τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων. Ιδίω οι οικογένειε με μικρά παιδιά, αλλά και οι κτηνοτρόφοι αγελάδων γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα που δημιουργούνται κάθε φορά, κάθε έξι μήνε που αλλάζει η ώρα. Στην Επιτροπή γεωργία λοιπόν ε, υπερψηφίσαμε την πρόταση αλλαγής, τερματισμού της ε, εποχικής αλλαγής της ώρας από το 2021. Πρέπει όμως να γίνουν σεβαστά τα εξή σημεία. Η εσωτερική αγορά πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί εύρυθμα. Γι' αυτό χρειάζεται συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτό που επίσης πρέπει να εμποδιστεί είναι να δημιουργηθεί ένα μοσαϊκό διαφόρων ζωνών ώρα μεταξύ των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη πρέπει από κοινού να αποφασίσουν. Θέλουμε μία ενιαία ώρα, στην, ε, τυπική ώρα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ή θέλουμε να θεσπίσουμε ως τυπική ώρα την θερινή ώρα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα λειτουργεί η ενιαία αγορά. Ευχαριστούμε εξ ονόματος Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Το λόγο κύριος Σβόμποντα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, η έκθεση για τον τερματισμό της εποχής αλλαγής της ώρας, την οποία θα ψηφίσουμε αύριο, αποτελεί συμβιβασμό τον οποίο υποστηρίζω 100%. Υιοθετώντα αυτή την έκθεση, θα σημειώσουμε μια επιτυχία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακούμε τις επιθυμίες των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό που επιζητούμε είναι να σταματήσουμε τις εποχικές αλλαγές της ώρας το 2021, ιδιαίτερα εξαιτίας των επιπτώσεων που έχουν αυτές στην ανθρώπινη υγεία. Πρέπει ταυτόχρονα να δώσουμε και ασφάλεια στην εσωτερική αγορά. Γι' αυτό το λόγο προβλέπουμε την δυνατότητα μέσω κατεξιότηση πράξης η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίσει τα κράτη-μέλη. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε ε, να ψηφίσουμε αυτή την έκθεση πριν το τέλος της θητείας μας και το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα δώσουν συνέχεια. Ευχαριστώ. Ακούσαμε την άποψη του συγητή και των γνωμοδοτικών επιτροπών. Τώρα έχουμε τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Από το ΕΛΚ πρώτα ο κύριο Βίμ Βαντενκάμπ για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ας μην υπάρχει καμία παρανόηση. Εγώ σαφώς είμαι υποστηρικτής τη θερινή ώρα. και νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, όσοι έχουν ε, ε, Μοτοσακό ουσιαστικά συμφωνούν περισσότερο και υποστηρίζουν περισσότερο την ε, θερινή ώρα. Τώρα, αν ένα 20% των Ευρωπαίων πολιτών αντιμετωπίζουν προβλήματα υγεία εξαιτία εποχική αλλαγή τη ώρα, ε, τότε μάλλον πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με το ζήτημα αυτό. Και προφανώ θα πρέπει να γίνουν και έρευνε, αλλά μην ξεχνάμε ότι έγινε και μια διαβούλευση. Και είχαμε πάρα πολλά εκατομμύρια που συμμετείχαν, αλλά και πολλά εκατομμύρια τα οποία δεν συμμετείχαν στην έρευνα αυτή. Μην ξεχνάμε λοιπόν λίγο και τα αριθμητικά δεδομένα, κυρία Επίτροπε. Είπα ότι υποστηρίζω σαφώ την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών. Υπήρχαν κάποια ζητήματα όπως η εξοικονόμηση ενέργειας βέβαια που δεν αναφέρονται πλέον στην έκθεση αυτή. Διατρέχουμε όμως πάντα τον κίνδυνο να επηρεαστεί αρνητικά η εσωτερική αγορά. Και νομίζω ότι θα ήταν κρίμα να συμβεί κάτι τέτοιο. Εσείς από ό,τι φαίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ταχθήκατε κατά μιας, ενός μηχανισμού συντονισμού τον οποίο είχαν αναφέρει οι συγητές και οι σκιώδη συγητές και είχαν πει ότι αυτό ο συντονιστικός μηχανισμός θα ήταν πάρα πολύ σημαντικός για την εσωτερική αγορά και ιδίω για το τομέα των μεταφορών. Σας καλώ λοιπόν κύριε Επίτροπε και μία ακόμη φορά να ασχοληθείτε με το ζήτημα αυτό του μηχανισμού συντονισμού. Εξ των σοσιαλιστών τώρα το λόγο έχει η κυρία Γιακονσάρη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ζήτησαν να καταργηθεί η εποχική αλλαγή της ώρας. Εμείς λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε καθήκον να απαντήσουμε στο αίτημα αυτό. Η αλλαγή της ώρας είναι ένα φαινόμενο, μια διαδικασία τεχνητή. Πρέπει να ανήκει στο παρελθόν. Γιατί πολλέ μελέτες και έρευνε, όπω είπε και η κυρία Ούλφσκα, έχουν αποδείξει ότι τα ωφέλη είναι απειροελάχιστα, ενώ αντιθέτω οι αρνητικέ επιπτώσει στην ανθρώπινη υγεία, στην υγεία των ζώων, είναι πολύ σημαντικότερε από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Χρειάζεται όμως ευρωπαϊκός συντενισμό, ώστε οι ρυθμίσει για την ώρα στα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει ένα μοσαϊκό μεταξύ των ζωνών ώρας για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η Κομισιόν μάλιστα είχε υποβάλει και μια πιο ρηξικέλευτη πρόταση για την κατάργηση της εποχικής αλλαγής της ώρας φέτος. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι πρέπει το συντομότερο δυνατό να ε, προχωρήσουμε και να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. μινούτο. κύριος για το ECR έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι περισσότεροι ε, Ευρωπαίοι αντιτέθηκαν, ε, διαφώνησαν με τις εποχικές αλλαγές της ώρας. Είναι μια πρακτική αναχρονιστική θα έλεγα. Αυτό όμως που θέλω να αναδείξω είναι το γεγονός ότι είναι πολύ θετικό το ότι ε, ελήφθη υπόψη η δική μας έκκληση αυτός ο τερματισμός να ισχύσει από το 2021 ε, από το 2021 και μετά. Ξέρετε, έχουμε και συμβάσει και ε, συμφωνίε και με χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να τι σεβαστούμε και να τι στηρίσουμε. Είναι σκάνδαλο ε, το γεγονός ότι δεν συνοδεύτηκε βεβαίως η πρόταση της Κομισιόν από αξιολόγηση επιπτώσεων. Θα έπρεπε να είχαμε λάβει την αξιολόγηση επιπτώσεων ε, πολύ νωρίτερα από ό,τι τη λάβαμε. Και αυτό ε, όχι μόνο, αλλά και για τους, ε, για, για, τους λόγους που θα, για τις επιπτώσεις που θα έχει ο τερματισμός της εποχικής αλλαγής της ώρας στις μεταφορές. Εγώ το μόνο που θέλω να τονίσω είναι ότι το, το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να είναι εκείνο που θα αποφασίσει σε ποια ζώνη θα ανήκει. Κύριε Μπιλμπά Παραντίκα, και το λόγο για δύο λεπτά εξ των φιλελευθέρων. Ε, μια παροιμία λέει ότι επειδή θα ξυπνήσει πιο νωρί δεν σημαίνει ότι θα ξημερώσει πιο νωρί. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Ε, και αυτή είναι και η έννοια τη συμφωνία στην οποία κατέληξε η Συμφωνία Μεταφορών. Χωρί ε, καθυστερήσει αλλά και χωρί βιασύνη θα πρέπει να τερματιστούν οι εποχικέ αλλαγέ τη ώρα. Δίνουμε λοιπόν στον εαυτό μα δύο ακόμα χρόνια για να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν αν θα διαλέξουν την χειμερινή ή τη θερινή ώρα και η μετάβαση να γίνει με εύρυθμο τρόπο. Πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι οι αποφάσει που θα ληφθούν δεν θα δημιουργήσουν περαιτέρω διαστρεβλώσει στην εσωτερική αγορά και στι βασικέ υπηρεσίε. Και δεν θα πρέπει να καθυστερήσουμε από την άλλη μεριά, γιατί όλοι γνωρίζουμε πω οι εποχικέ αλλαγέ πρέπει να τερματιστούν. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ τη άποψη ότι οι βλάβες προκύπτουν ε, είναι πολύ περισσότερες από τι ωφέλειε, ιδιαίτερα για παιδιά και για ηλικιωμένους. Και πολύ δε περισσότερο που ε, οι εποχικέ αλλαγέ ε, δεν συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση ενέργειας όσο παλιότερα. Οπότε χρειάζεται τα κράτη-μέλη και ή τα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλύσουν από κοινού σε μια επιτροπή τι προτάσει κάθε κράτου μέλους και να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να ε, αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Ε, μετά από αυτή την περίοδο, το 2021, θα μπορούσαμε εφτακτά και εύρυθμα να περάσουμε στην κατάργηση των εποχικών αλλαγών. Αυτή η αξιολόγηση θα επιτρέψει να, να βεβαιωθούμε ότι τα προβλήματα που θα λύσουμε θα είναι περισσότερα από αυτά που θα δημιουργήσουμε ε, 4.600.000 πολίτε ε, συμμετέσχουν στην δημόσια διαβούλευση και θα πρέπει να ακούσουμε τη φωνή του Θα πρέπει να δείξουμε ότι τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται δίπλα του και ε, παίζουν το ρόλο που του αντιστοιχεί. Πρέπει να ενημερώνονται τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και με διαφάνεια να προσπαθήσουν να βρουν ισορροπημένε λύσει. Αν με αυτόν τον τρόπο βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας, το, η Ευρώπη θα είναι ε, μια πραγματική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Εξ ονόματο των Πρασίνων, ο κύριος Νταλούντε, το ρευτό λόγο, για ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ορισμένοι από τους συναδέλφους εδώ πέρα ουσιαστικά λένε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να ασχοληθεί με πολλά άλλα ζητήματα και όχι με την εποχική αλλαγή της ώρας. Οι συνάδελφοι αυτοί δεν έχουν καταλάβει τη σημασία του ζητήματος αυτού, καθότι 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις λάβαμε στα πλαίσια της ανοιχτή διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένα 84% των πολιτών αυτών θέλουν την κατάργηση των εποχικών αλλαγών της ώρας. Και υπάρχουν και πάρα πολλές επιστημονικές μελέτες που μας δείχνουν ότι είναι πολύ πιο θετικό να μην έχουμε εποχική αλλαγή τη ώρα. Με την αλλαγή τη ώρα έχουμε περισσότερες κρατικέ προσβολές, περισσότερα τροχαία ατυχήματα κ.ο.κ. Ορισμένοι ανησυχούν για το ότι ενδεχομένως η οδηγία αυτή να δημιουργήσει ένα κατακαιρματισμό των ε, ορών, των ζωνών ορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να δημιουργήσει ένα μηχανισμό συντονισμού, έτσι ώστε να έχουμε ένα εναρμονισμένο σύστημα για την ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποφύγουμε όμως την εποχική αλλαγή της ώρας. η κυρία Κίλωνεν τώρα έχει το λόγο ξενόματος της ΓΚΟΕ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Η αλλαγή της ώρας αναδείχθηκε ως ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στη χώρα μου. Και εγώ καταλαβαίνω γιατί. Είναι ένα πολύ απλό, συγκεκριμένο ερώτημα, στο οποίο μπορεί να δοθεί μια πολύ απλή και συγκεκριμένη απάντηση και που αφορά κάθε πολίτη ξεχωριστά. Γι' αυτό και θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά ε, την υπόθεση αυτή. Ακούσαμε λοιπόν τους πολίτες, αναλάβαμε δράση, αναλάβαμε πρωτοβουλία πάνω σε ένα θέμα που τους απασχολεί. Και παρά το γεγονό ότι δεν μπορούμε ε, να λάβουμε αποφάσεις για φέτος ή για του χρόνου, είναι πολύ σημαντικό το γεγονό ότι έχουμε πλέον μια συγκεκριμένη ημερομηνία, μια συγκεκριμένη χρονολογία, από την οποία και έπειτα θα ισχύσει η σχετική απόφαση για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών τη ώρα. Οι επιπτώσει στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων είναι αδιαμφισβήτητε. Και μιλώ για την υγεία, την ψυχική, την σωματική, την πνευματική των ανθρώπων. Αυτά φαίνονται στις μεταφορές, στην οικονομία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βεβαίω, χρειάζεται χρόνο για να γίνουν οι αναγκαίε προσαρμογέ στη νέα κατάσταση αν θέλουμε πραγματικά να εξασφαλίσουμε ότι θα καταλήξουμε σε μια ευφυή, συντονισμένη απάντηση η οποία θα ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών. Για την ομάδα EFDD, η κυρία Ιαϊούτο έχει το λόγο. Ντανιέλ, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε. Εγώ ουσιαστικά διαφωνώ με την πρόταση αυτή, με την πρωτοβουλία αυτή για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχάς δεν υπάρχει κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να αποδεικνύει πραγματικά ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις από την εποχική αλλαγή της ώρας για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την παραγωγικότητα. Από την άλλη, μια τροποποίηση της οδηγίας ουσιαστικά θα τόνιζε όλο και περισσότερο τις στρεβλώσει ανταγωνισμού ή τι οικονομίε που θα μπορούσαν να προκύψουν στην εσωτερική αγορά ή ακόμα και στην γεωργία. Η έγκριση της θερινής ώρας ως επίσημη ώρα, ουσιαστικά και η εποχική εναλλαγή με τη χειμερινή ώρα οδηγεί σε εξοικονόμηση της ενέργειας και πολύ φοβάμαι ότι αν εγκρίνουμε την οδηγία αυτή θα έχουμε αρνητικές επιπτώσεις και στον τομέα αυτό. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι θα υπάρχει πάντα διακριτική ευχαίρεση στα κράτη-μέλη να επιλέξουν την επίσημη ώρα τους, ενώ ουσιαστικά υποτίθεται ότι θα έπρεπε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να θέλουμε να έχουμε ένα, ευρω... ένα εναρμονισμένο σύστημα ώρας και σε σχέση με τις τρίτες ώρες. Επίσης, δεν υπάρχει καμία καμία τεκμη, επιστημονικά, τεκμηριο, καμία επιστημονικά τεκμηριωμένη απόδειξη όσον αφορά τι αρνητικέ επιπτώσει που έχει η εποχική αλλαγή τη ώρα στη δημόσια υγεία. Α μην ξεχνάμε ότι μολονότι έγινε ανοιχτή διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έγινε ανοιχτό διάλογο και συζητήσει στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Μελάντρο έχει το λόγο ξανόματο του ΙΕΝΕΦ για δύο λεπτά. Η εποχική αλλαγή δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης η εξοικονόμηση ενέργειας ε, πλέον είναι μηδαμινή, ενώ τα αρνητικά αποτελέσματα ε, έχουν πλέον αποδειχθεί. Το, η μετάβαση από την ώρα του χειμώνα στην ώρα του καλοκαιριού δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Αν ε, μάλιστα συνεχιστεί αυτή η αλλαγή, ή αν επιλεγεί η καλοκαιρινή ώρα μόνιμα, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα και στους ε, ανθρώπους και στα ζώα. Το τέλος εποχικής αλλαγής λοιπόν είναι μια ανάγκη. Χρειάζεται όμως ε, συντονισμός. Το κάθε κράτος όμως θα πρέπει να έχει την επιλογή της, του καθορισμού της επίσημης ώρας, της, ώρας του θα πρέπει να αποφύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναμειχθεί. Είναι όταν αναμίχθηκε με, και επέβαλε την τακτική αλλαγή της ε, ώρας, δημιούργησε προβλήματα τα οποία τώρα δεν μπορεί να λύσει και να αποσύρει αυτή την απόφαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ακούσαμε την άποψη των πολιτικών ομάδων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τώρα πλέον και τις μπλε κάρτες. Και ο κύριος Κόκ έχει πρώτος τώρα το λόγο για ένα μισή λεπτό. Κυρία Επίτροπε, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας σημαίνει ότι πρέπει να απαλλαγούμε από όλα όσα δεν μας ωφελούν. Οι συνθήκες λοιπόν είναι όριμες πια για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών. Α θέσουμε επιτέλου ένα τέρμα στις αρνητικέ επιπτώσεις στην υγεία το 20% του πληθυσμού και στι αρνητικέ επιπτώσεις που έχουν στην οικονομία οι αλλαγέ αυτές, στις μεταφορές, στην ασφάλεια των μεταφορών αλλά και στην ε, διαταραχή του βιορυθμού των ζώων. Ακόμη και οι συνάδελφοι που διαφωνούσαν ε, παλαιότερα με τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών συμφωνούν πλέον εδώ και 10 χρόνια καλό να τερματιστεί. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι θα τερματιστεί ή θα καταργηθεί η θερινή ώρα. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν αν θέλουν να διατηρήσουν την κανονική ή τη θερινή ώρα. Για να ε, αποφευθούν λοιπόν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός, ένας μηχανισμός συντονισμού. Τρεις ζώνες ώρας νομίζω ότι αρκούν για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κύριος Νέκοφ, τώρα για ένα λεπτό παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα των ε, αλλαγών της ώρας βεβαίως δεν είναι πρώτη φορά που συζητείται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα ε, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ε, ανέφεραν σε μια τεράστια διαβούλευση που έγινε ότι θέλουν να καταργηθεί η πρακτική αυτή. Επιστημονικά, οικονομικά, η πρακτική αυτή είναι αναχρονιστική, περιορίζει την παραγωγικότητα των εργαζομένων, περιορίζει τα ωφέλη που κάποτε επιδιώχθηκαν να επιτευχθούν. Εγώ λοιπόν προτείνω την, ε, ε, Είμαι υπέρ τη πρόταση αυτή, εφόσον βεβαίω υπάρξει ένα μηχανισμό συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν στρεβλώσει στη λειτουργία τη ενία αγορά. Καλό λοιπόν και το Συμβούλιο να αναλάβει και να αρθεί στο ύψο των, περιστάσεων να καταλήξει σε θέση. Κύριε τώρα ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ε, ήμουν υπέρ της κατάργησης των εποχικών αλλαγών της ώρας. Γιατί κάτι τέτοιο θα απλουστεύσει και την καθημερινότητα των ε, πολιτών. Διότι αυτές οι αλλαγές της ώρας, όπως υπόθηκε και νωρίτερα, τελικά δεν οδηγούν στις ε, επιθυμητές εξοικονομήσεις ενέργειας. Αυτό ήταν ο αρχικός σκοπός, αλλά ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν αυτές οι εξοικονομήσεις. Αν όμως ε, ακούσουμε ε, τις προτάσεις της ε, Κομισιόν θα χάσουμε την, ε, την εναρμόνιση. Εμείς θέλουμε να υπάρξει ένας συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ε, ενιαίας αγοράς. Η έκκληση λοιπόν του Κοινοβουλίου για την θέσπιση μηχανισμού συντονισμού θεωρώ ότι είναι θετική, διότι δεν θα πρέπει η κατάργηση των εποχικών αλλαγών ε, τελικά να οδηγήσει σε υποχώρηση της λειτουργίας ε, της ε, εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει το κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει αν θέλει να διατηρήσει την κανονική του ώρα ή την θερινή ώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν θεσπίστηκαν οι εποχικές αλλαγές της ώρας, σκοπός ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας. Ε, και επίσης ε, σκοπός ήταν να αποφευχθούν ε, τα ατυχήματα. Ε, γιατί το πρωί κυκλοφορούν στους δρόμους και περισσότερα παιδιά βεβαίως από το βράδυ. Χρονοβιολόγοι λοιπόν έλαβαν το βραβείο Νόμπελ γιατί διαπίστωσαν ότι για ανθρώπους, ιδίως για ασθενείς και ηλικιωμένους, ε, δημιουργεί προβλήματα η αλλαγή τη ώρα. Όταν λοιπόν έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία πια στα χέρια μα, γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Η Ρωσία και η Κίνα έχουν ήδη καταργήσει τι εποχικέ αλλαγέ τη ώρα. Νομίζω μπορούμε να το κάνουμε και εμεί. Και όσον αφορά την εσωτερική αγορά, όταν θεσπίστηκε η αλλαγή, συμφωνήθηκε μια συγκεκριμένη ώρα. Μάλιστα συμμετείχε και η Ελβετία, παρά το γεγονό ότι ο πληθυσμό τη χώρα είχε αντιτεθεί, είχε διαφωνήσει. Ξέρω, η Ελβετία δεν είναι μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλα αυτά συμμετείχε σε εκείνη τη διαδικασία. Ε, το ίδιο σίγουρα μπορούμε να το κάνουμε και σήμερα Γι' αυτό και καλό κάθε συνάδελφο να υπερψηφίσει την πρόταση αυτή. Πέντε χρόνια που είμαι μέλος άλλαξαν πολλά. Ένα πράγμα δεν άλλαξε. Ότι η εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει καλύτερα. Το δικό μας ε, κοινοβούλιο ξέφρασε την άποψή του για αυτό το θέμα. Ε, εντόπισε το ότι δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για να διακοπεί η εποχική αλλαγή. Αυτή η απαγόρευση, πρωτοβουλία ε, είναι μία ακόμα προσβολή στην αρχή της επικορικότητας. Η φιλοσοφία σας ε, για μια όλο και πιο στενά ενωμένη Ευρώπη είναι εγωιστική. Θα έπρεπε τα κράτη-μέλη να παίρνουν τις αποφάσεις αυτές, ανάλογα με το τι του επιβάλλει η οικονομία και η γεωγραφία τους όχι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αν η κυβέρνησή μας μας εκπλήξει και βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαι σίγουρος ότι θα αγνοήσουμε αυτή την πρόταση. Κύριε Μέιντελ, τώρα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Επίτροπε, Η σημερινή συζήτηση καταδεικνύει ότι όντως αφουγκραζόμαστε την άποψη των Ευρωπαίων πολιτών. Όπως υπόθηκε και από τους συναδέλφους, το 84% των Ευρωπαίων πολιτών που συμμετείχαν στην ανοιχτή διαβούλευση Ευρωπαϊκής Επιτροπής τάχθηκαν υπέρ της κατάργησης των εποχικών αλλαγών της ώρας. Έτσι λοιπόν, ως εισηγήτρια της γνωμοδότησης του ΕΛΚ για την Επιτροπή ΙΜΚΟ, ασχολήθηκα ιδιαίτερα με το ζήτημα αυτό. Φαίνεται ότι οι εποχικές αλλαγές οδηγούν σε περισσότερη αϊπνία, σε αδυναμία συγκέντρωσης, σε περισσότερα ατυχήματα τροχαία αλλά και στον χώρο εργασίας και στο παρελθόν, η εξοικονόμηση ενέργεια ήταν το βασικό επιχείρημα που χρησιμοποιείται για να δικαιολογηθεί η εποχική αλλαγή τη ώρα. Δεν υφίσταται όμω ένα τέτοιο επιχείρημα πλέον. Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι ακόμα και αν υπήρχε ένα οικονομικό επιχείρημα υπέρ τη εποχική αλλαγή τη ώρα, μπορεί αυτό να παρίνει περισσότερο από τη δημόσια υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει να δείξουμε στου πολίτε ότι λαμβάνουμε πολύ σοφαρά υπόψη την άποψή του. Έτσι λοιπόν, το αργότερο το 2021 θα πρέπει να σταματήσουν οι εποχικέ αλλαγέ τη να Συναπόκειται πια στο Συμβούλιο να αναλάβει δράση. Σας ευχαριστώ. Νίκολσον τώρα. Κύριος Νίκολσον, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα τους συναδέλφους που είπαν ότι δεν είναι το πιο σημαντικό ζήτημα το οποίο καλεί να αντιμετωπίσει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Γιατί αν δείτε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την εποχική αλλαγή της ώρας ε, μπορεί να μην είναι ίσως το πρώτο θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παραδεχτεί ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι απαραίτητες ε, έρευνες ή τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να δικαιολογηθεί η κατάργηση της εποχικής αλλαγής της ώρας. Έχουμε από τη Βόρεια Ιρλανδία, έχουμε ήδη αρκετά προβλήματα με το backstop και με το Brexit και νομίζω ότι είναι τρελός αυτή τη στιγμή να ε, έχουμε ενδεχομένω όμορες περιοχές στην παραμεθόριο, οι οποίες θα βρίσκονται στην τελώς διαφορετική ε, ζώνη ώρα. Θα είναι παράλογο να προκύψει κάτι τέτοιο. Έχουμε ήδη πάρα πολλά προβλήματα. Α μην προσθέσουμε και αυτό το πρόβλημα. Το σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή λειτουργεί καλά. Α μην το αλλάξουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να απορρίψουμε την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Λίζε έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γιατί να τα κάνουμε απλά τα πράγματα όταν μπορούμε να τα περιπλέξουμε κιόλα. Αυτή είναι η... αυτός είναι ο χαρακτηρισμό που μπορώ να δώσω στη στάση του Συμβουλίου αλλά και του Κοινοβουλίου. Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, όχι μόνο στην ε, ηλεκτρονική διαβούλευση που διεξήγαγε η Κομισιόν, και γιατί να κάνουμε διαβούλευση άλλωστε αν δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι λένε οι πολίτες αλλά ακόμα και σε αντιπροσωπευτικές έρευνες δήλωσε ότι δεν θέλει τις αλλαγές. Ως γιατρός λοιπόν σας βεβαιώνω ότι υπάρχουν σημαντικότατα προβλήματα για την υγεία του ανθρώπου. Πόσο σοβαρά είναι, πόσο μεγάλα είναι μπορεί να χρειαστεί να το διαρευνήσουμε περαιτέρω. Αλλά πάντως είναι γεγονός ότι η αλλαγή της ώρας δεν επιφέρει κανένα όφελος σε κανέναν και γι' αυτό και πρέπει να καταργηθεί. Τα στοιχεία λοιπόν και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν ε, νομίζω ότι δεν είναι αρκετά πιστικά κατά της πρότασης της Επιτροπής Μεταφορών. Διότι το γεγονός ότι ε, υπάρχει πιθανότητα στην Ευρώπη να δημιουργηθεί ένας κατακαιρματισμός των ε, ζωνών ώρας, αυτό είναι μια πιθανότητα ακόμη και σημερινή. Ισχύει σήμερα. Ακόμα και σήμερα κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι αλλάζει ζώνη ώρας. Γι' αυτό και καλώ όλους τους συναδέλφου να υπερψηφίσουν την πρόταση της Επιτροπής Μεταφορών και από εκεί και πέρα επιτέλους να πιάσει δουλειά και το Συμβούλιο. κυρία Λουκατσικέσκα τώρα έχει το λόγο για να λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η κατάργηση των εποχικών αλλαγών της ώρας δεν θα, δεν θα έπρεπε να δημιουργεί τόσο μεγάλες εντάσεις εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο. Αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτά τα πολύ απλά θέματα, τι θα κάνουμε και στα πιο σοβαρά θέματα δηλαδή. Παρά όλα αυτά, εγώ είμαι μεταξύ εκείνων που και με τα δύο χέρια υπερψηφίζουμε ε, αυτήν την πρόταση που άλλωστε βασίζεται και στα όσα μας ζήτησαν οι πολίτες μέσα από την διαβούλευση που συμμετείχαν κατά εκατομμύρια στη διαβούλευση αυτή οι ιατρικέ πτυχές του θέματος, οι γεωργικές πτυχές, οι οικονομικές πτυχές του θέματος, όλες βοούν ότι πραγματικά πρέπει επιτέλους να απαλλαγούμε από αυτήν την αναχρονιστική πρακτική της αλλαγή της ώρας. Φυσικά, είναι πολλές φορές δύσκολο κανείς να ξεπεράσει συνήθειες δεκαετιών. Αλλά Δυστυχώ σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει πραγματικά ούτε μισό επιχείρημα το οποίο θα μπορούσε να στηρίξει τη διατήρηση του σημερινού καθεστώτο. Βεβαίω χρειάζεται χρόνο ώστε να γίνουν οι αναγκαίε προσαρμογέ από τα κράτη-μέλη για να μην χρειαστεί η Κομισιόν να παρατείνει ή να αναβάλει την θέση σε ισχύ αυτού του τερματισμού τη ώρα. Κέλλη, Ο κ. Κέλλη, ένα λεπτό. ποτέ δεν ε, βρήκα τη λογική αυτής της εποχής αλλαγής. Ε, και μάλιστα όταν ε, δημιουργήσαμε μια ομάδα για αυτό το θέμα, ε, κατά τη διάρκεια των ασιών μας αντιληφθήκαμε ότι ε, τα ωφέλη λιγότερα από τις βλάβες που προκαλούνται από την εποχή αλλαγή. Η Κομισιόν είχε προτείνει μάλιστα η εποχική αλλαγή να τερματιστεί φέτος. 84% των συμμετεχόντων στη διαβούλευση το επιθυμούσαν. Από τα 4,6 εκατομμύρια άτομα που συμμετείχαν. Θα πρέπει όμως να υπάρξει ένας μηχανισμός συντονισμού έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και να αποφασίσουν με ποιο τρόπο θα γίνει αυτή η μετάβαση. Ε, το πότε θα γίνει η, ο τερματισμό και το αν θα επιλεγεί η θερινή χειμερινή ώρα. Ευχαριστώ. Κυρία Σράιερ Πιέρκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όντω ε, έγινε μια έρευνα και πάρα πολλοί ε, συμμετείχαν στην έρευνα αυτή. Και αναφέρομαι στην διαβούλευση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι περισσότεροι τάχθηκαν υπέρ τη κατάργηση των εποχικών αλλαγών τη ώρα. Δεν μιλάμε πλέον για εξοικονόμηση ενέργεια. Αυτό είναι εντελώ αναχρονιστικό. Το δείξανε και οι ίδιε οι έρευνε. Υπάρχει πρόβλημα με του βιορυθμού των ανθρώπων. Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, υψηλά ποσοστά καρδιαγκιακών προσβολών. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μα. Χρειαζόμαστε σαφώς μια καλή συνεργασία μεταξύ των κρατών και αν δεν το πετύχουμε αυτό, τότε δεν νομίζω ότι είμαστε αντάξει των Ευρωπαίων πολιτών. Θεωρώ ότι θα πρέπει πραγματικά να καταργηθεί το ιστορικό αυτό πρόβλημα. Κάθε χρόνο 5 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν λόγω της εποχικής αλλαγής της ώρας. Α σταματήσει πλέον το σύστημα αυτό. Η διαβούλευση ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, θεωρώ, γιατί κατέδειξε τελικά ότι ε, υφίστανται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σημαντικέ δυσκολίε, τι οποίε πρέπει να υπερκεράσουμε. Εφτά επιτροπέ συμμετείχαν και ιδίω η Επιτροπή Μεταφορών, η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, κατέθεσε μια συγκεκριμένη έκθεση και στην έκθεση αυτή δεν αφαιρθήκαμε μόνο στι μεταφορέ, αλλά και σε άλλα ζητήματα. Πρόεδρο. κύριε Σράερ Πιέρικ, σε εσά αναφέρομαι. Κυρία Σράερ Πιέρικ, με συγχωρείτε. Υπάρχει μια μπλε κάρτα για εσά, τη δέχεστε. Πολύ ωραία. Την ερώτηση θέλει να κάνει ο κύριος Βάντεν Μίντεμπουρκ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ, ακούμε την ερώτησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στραεπίκ, εσείς ε, κατάγεστε από μεθοριακή περιοχή ανάμεσα στην Ολλανδία και την ε, Γερμανία. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος οι δύο ε, αυτές χώρες να βρεθούν σε διαφορετικές ζώνες ώρας. Πώς θα εξηγήσετε σε ανθρώπους που ζουν κοντά στα σύνορα ότι θα πρέπει να ζουν σε δύο διαφορετικές ζώνες ώρας. Εσεί δέχεστε τον κατακαιρματισμό τη ενιαία αγορά. Και αν όχι, πώ θα τον εμποδίσετε. Τι θα πείτε στου επιχειρηματίε και σε όλου του άλλου που δραστηριοποιούνται και ζουν σε αυτή τη μεθοριακή περιοχή όταν θα σα θέτουν τέτοια ερωτήματα. Ευχαριστώ ε, τον Ολλανδό συνάδελφό μου για αυτή την ερώτηση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί μια χαρά μπορούν να συζητήσουν και να συμφωνήσουν. Έχουμε ήδη στην Ευρώπη τρεις διαφορετικές ζώνες ώρας και πρέπει κανείς να ακούσει τους πολίτες τους. Το πρόβλημά σας είναι ότι ακούτε μόνο τους επιχειρηματίες. Εγώ δεν έκανα αυτό. Εγώ παρακολουθώ την υπόθεση και τη συζήτηση αυτή εδώ και 12 χρόνια και από το Εθνικό μου Κοινοβούλιο, πρωτού εκλεγώ Ευρωβουλευτής και νομίζω ότι πλέον είναι υπερόριμες οι συνθήκες. Κύριος Γκρίσπς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση αυτή αποτελεί την κορύφωση προσπαθειών πολλών ανθρώπων και στην προηγούμενη θητεία είχε θεσπιστεί και μια σχετική ομάδα εργασίας υπό τον κύριο Γκρόελ και σε αυτή τη θητεία είχαμε την ομάδα εργασίας υπό τον κύριο Σβόμποντα. Από τις προσπάθειες αυτές λοιπόν καταλήξαμε σε αυτή την πρόταση που συζητούμε και σε αυτή την έκθεση που συζητούμε σήμερα σε πάρα πολλά κοινοβούλια κρατών μελών της Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Φιλανδία, στην Πολωνία και σε άλλες χώρες έχει συζητηθεί το θέμα επί και σε βάθος. Δεν πρόκειται λοιπόν για κάποιο θέμα καινοφανέ. Η δε δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε κατέδειξε ότι υπάρχουν εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτε που θέλουν την κατάργηση τη αλλαγή τη ώρα. Όμω θα πρέπει να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση. Κάλιο αργά Κάλιο αργά παραποτέ αφενός, αλλά πιο καλά είναι να γίνουν τα πράγματα γρήγορα. Γιατί θεωρώ ότι ε, θα αποτελέσει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά αφουγκράζεται τις ανησυχίες και τα προβλήματα των πολιτών. Υπάρχουν προβλήματα υγείας, πνευματικής και σωματικής, ε, ακόμα και οικονομικά προβλήματα που προκαλούνται από αυτήν την αλλαγή της ώρας. Πρέπει επιτέλους λοιπόν να προχωρήσουμε. Κύριος Λάγκη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κανείς δεν θα αμφισβητήσει ότι μια ε, μειοψηφία ε, ε, έχει, αντιμετωπίζει κάποια παροδικά προβλήματα υγείας. Όμως εγώ επαναφέρω το εξής επιχείρημα. Ο άνθρωπος χρειάζεται ηλιοφόνια. Αλλά εδώ υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Όσο και να συζητάμε αυτό το θέμα, πάνω από 2% ευρωβουλευτές δεν συμμετέχουν ποτέ σε αυτές τις συζητήσεις. Νομίζω ότι η όλη διαδικασία, η όλη πρόταση είναι δυσανάλογη, δεν υπάρχει αξιολόγηση επιπτώσεων, πρέπει να την πετάξουμε στα σκουπίδια αυτή την πρόταση. Γι' αυτό και λέω απερίφραστα ότι εγώ θα την καταψηφίσω την πρόταση αυτή και εγώ πραγματικά ανυπομονώ να έρθει επιτέλους η ε, επόμενη φορά σε μια εβδομάδα που θα ξαναλλάξουμε και θα πάμε στη θερινή ώρα. Ευχαριστώ κύριος Πέτρελε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω την αλλαγή αυτή. και μάλιστα ελπίζω το συντομότερο δυνατό να καταργηθεί η εποχική αλλαγή. Όχι μόνο για οικονομικούς λόγους. Είναι σημαντικός ο άνθρωπος. Η σημασία που έχουν, αυτοί, έχουν αυτές οι εποχικές αλλαγές για τους ανθρώπους και για την υγεία τους. Αυξάνουν τους κινδύνους εγκεφαλικών επεισοδίων και εμφραγμάτων. Μειώνουν την ικανότητα συγκέντρωσης, αυξάνουν τον αριθμό των ατυχημάτων κλπ. κλπ. Σε μέρες που ακολουθούν την αλλαγή της, ε, την εποχική αλλαγή της ώρας αυξάνει το αριθμό των τροχιών ατυχημάτων για παράδειγμα. Οπότε υπάρχουν λόγοι να καταργηθεί αυτή η εποχική αλλαγή. Χωρίς όμως να δημιουργήσουμε πρόσθετα προβλήματα. Ο στόχος είναι να διευκολύνουμε τους ανθρώπους τη ζωή τους. Κανένας δεν θα ήθελε 10 γειτονικέ χώρε να έχουν 10 διαφορετικέ επίσημε ώρε. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Κύριε Πέτερλε, επειδή έχουμε και χρόνο, ε, υπάρχει μια ερώτηση για σας μέσω μπλε κάρτα. στη δέχεστε από τον κύριο Λάγκεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εσείς πού βασίζεστε όταν λέτε ότι ε, δεν δημιουργούνται βλάβες. Το αντίθετο λένε οι ε, Αμερικανοί ε, επιστήμονες. Εγώ βασίζομαι σε έρευνες που έχουν γίνει και τις οποίες συνέλεξε το προσωπικό μου. Νομίζω ότι έχω τα σωστά στοιχεία και έχω υποβάλει τα σωστά επιχειρήματα υπέρ της πρότασης αυτής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φαντάλη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα εγκαταστήσουν ως επίσημη ώρα τους μόνιμα τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα, αλλά δεν υπάρχουν αρκετά επιχειρήματα. Ήδη στην Επιτροπή Μεταφορών υπήρχαν πολλοί εμπειρογνώμονες που μας είπαν ότι όλα αυτά τα οποία λέμε για την δημόσια υγεία ουσιαστικά δεν ισχύουν στην πράξη, δεν είναι αρκετά βάσιμα επιχειρήματα. Θα έλεγα ότι και πάλι το ότι θα βελτιωθούν οι μεταφορές, ή άλλες οικονομικές πτυχές εσωτερικής αγοράς δεν είναι κάτι το οποίο στέκει στην πράξη. Θα έλεγα ότι είναι συναισθηματικά φορτισμένη περισσότερο η συζήτηση, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Θα αυξηθεί η σύγχυση, θα καταρκματιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ζημιωθεί η εσωτερική αγορά. Πραγματικά θα έχουμε πολλέ διαφορετικέ ζώνε ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να απορρίψουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δείξει στεναρή στάση. Πολύ ωραία. Μπλε κάρτα υπάρχει για την προηγούμενη παρέμβαση. Τη δέχεστε καταρχάς, δέχεστε μπλε κάρτα. Πολύ ωραία. Σας ακούμε. Η κυρία Ζράιρε Πιέρικ έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λίγο συζήτηση μεταξύ Ολλανδών έχει καταλήξει αυτό. Πάντως, αυτή τη στιγμή λέγεται ότι δεν έχουμε βαθύνει πάρα πολύ. Εγώ θα έλεγα ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχω έρθει σε επαφή με καρδιολόγου και άλλου εμπειρογνώμονε, εμπειρογνώμονε στον τομέα τη ασφάλεια, των μεταφορών και υπάρχουν πλέον πάρα πολλά έγγραφα, μια πολύ σημαντική τεκμηρίωση. Νομίζω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχουν βάσιμα επιχειρήματα. Πραγματικά έχουμε εμβαθύνει στο ζήτημα πάρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σα καλώ να δείτε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει. Α ακούσουμε και την απάντηση από τον κύριο Βαντάλεν. Μα κοιτάξτε, έγινε μια ακρόαση, σημαντικότατη ακρόαση από το δικό μας το κοινοβούλιο και ήρθανε πάρα πολλοί εμπειρογνώμονε και όλοι μίλησαν κατά της πρότασης αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν υπάρχει Τίποτα που να αποδεικνύει τελικά ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να καταργήσουμε την εποχική αλλαγή τη ώρα. Είναι συναισθηματικά φορτισμένη η συζήτηση αυτή. Ουσιαστικά θέλουμε αυτή τη στιγμή να ικανοποιήσουμε τι ευχέ ενό μικρού ποσοστού των Ευρωπαίων πολιτών. Ολοκληρώνω τη διαδικασία Catch the Eye αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την μπλε κάρτα για βουλευτές της ίδιας πολιτικής ομάδας, καθότι όμως ε, η όλη αυτή η συζήτηση κέντρηση των ενδιαφέρων των περισσότερων, κάναμε μια εξαίρεση. Ο κύριος Στάραν τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπαν οι κύριοι Λάγκε και Βαντάλεν. Ο, ο Β' Δεύτερος και ο Κάιζερ ε, είδαν το έργο τους να συνεχίζεται από τον Χίτλερ και από τον Χίτλερ το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ένα από αυτά, τα, μία από αυτές πράξεις ε, ε, ήταν η αλλαγή της ώρας. Αυτή η αλλαγή της ώρας είναι ένα από τα τελευταία υπολείμματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ας την ακυρώσουμε λοιπόν. Δεν θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο χρόνο στο Συμβούλιο και σε εσά, κύριοι για να τα βρείτε μεταξύ σας. Ε, ε, δεν μπορούμε από την άλλη μεριά να, να, πείσουμε, επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν ένα patchwork από διαφορετικές ε, ώρες. Το Τόκιο και η Νέα Υόρκη μπορούν να λειτουργήσουν ο πρόεδρος διακόπτη τον ομιλητή. Σας ευχαριστούμε. Ζρέλεκ τώρα παρακαλώ. Όχι, όχι, δεν προβλέπετε μπλε κάρτα. Κύριε Ζρέλεκ, παρακαλώ για ένα λεπτό. Είστε στην αίθουσα. Ντάβος, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε Μπούλτς. Αυτό που συζητάμε εδώ είναι ένα από τα λιγότερα σημαντικά θέματα μεταξύ πολύ σημαντικών θεμάτων ιδίω αν λάβει κανεί υπόψη του τι αντιδράσει που έχουν υπάρξει αλλά και τι απαντήσει των πολιτών. Θέλω όμω να σταθώ σε ορισμένα θέματα που αναδείχθηκαν από τη συζήτηση. Ω μέλο τη άτυπη ομάδα εργασία, εγώ πάντοτε ε, υποστήριζα την κατάργηση των αλλαγών τη ώρα και φυσικά και θα υπερψηφίσω την έκθεση αύριο. Ωστόσο, θα ήθελα να ζητήσω από του αξιότιμου συναδέλφου που έχουν φέρει τα αντίθετα επιχειρήματα να μα πούν ποια ήταν τα επιχειρήματα πάνω στα οποία βασίστηκε η θέσπιση της αλλαγής της ώρας όταν αυτή έγινε. Πώς είναι δυνατόν να λέτε ότι η Κομισιόν δεν έκανε σοβαρή έρευνα. Ρωτήθηκαν οι πολίτες και με σαφήνεια τάχθηκαν υπέρ της κατάργησης του ισχύοντος συστήματος. Στην Κροατία, για παράδειγμα, 20.000 πολίτες συμμετείχαν στην πρωτοβουλία αυτή. 10 φορές περισσότεροι από εκείνους που συνήθως συμμετέχουν σε αντίστοιχε διαδικασίες για την υλοποίηση ευρωπαϊκών οδηγιών. Ο κ. Λόπες. Η συζήτηση και η απόφαση αυτή δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις ε, ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, γεωγραφικές, κοινωνικές, οικονομικές κλπ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο όνομα της της ενιαίας αγοράς προτείνει το τέλος της εποχικής αλλαγή, της εποχικής αλλαγής. Ε, δεν, η επιστημονική κοινότητα είναι διχασμένη όμως. Ούτε και για το ε, αν θα πρέπει να γίνεται η εποχική αλλαγή και για το αν αυτή η αλλαγή έχει ωφέλη, βλάβες και ποια είναι περισσότερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να έχει ξεχάσει ότι ο καθορισμός της επίσημης ώρας είναι εθνική αρμοδιότητα. Οπότε οι εποχικές αλλαγές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την άποψη του, των πολιτών, ε, της επιστημονικής κοινότητας και της κυβέρνησης κάθε χώρας. Ευχαριστώ. Non c'è. Onorevole Blanco Lopez, un minuto. Ultimo intervento. Blanco Lopez, για ένα λεπτό παρακαλώ. Είναι το σου μιλητή στη διαδικασία Catch Το μικρόφωνο παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εποχική αλλαγή της ώρας έχει συνέπειες στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Έχει οικονομικές, ενεργειακές, επιπτώσεις, επιπτώσεις στην ασφάλεια που επηρεάζουν την, το βιωτικό παιδό και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να πάρουμε ελαφρά την καρδία την πρόταση της Κομισιόν. Η πρόταση αυτή δεν συνοδεύεται από μια εξαντλητική αξιολόγηση. Το είπαμε αυτό. Και η Οδηγία 2084 ε, όσο και η πρόταση που μας υποβάλλεται δεν βασίζονται σε ε, στέρεα στοιχεία. Και δεν είναι δυνατόν να πάρουμε βεβαιασμένες αποφάσεις ε, που θα, κατα... δημιουργήσουν σύνορα και διαφορές ώρες εκεί που δεν υπάρχουν. Είναι σημαντικό να αναλύσουμε σε μεγαλύτερο βάθος ε, τις ε, συνέπειες αυτής της απόφασης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ας ακούσουμε τώρα την απάντηση της Επιτρόπου, κυρία Μπούλτσα. Βιολέτα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αξιότιμα μέλη. Άκουσα με πολύ προσοχή την παθιασμένη αυτή συζήτηση που έλαβε χώρα. Και προτού σχολιάσω περαιτέρω, θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι το πολύ σημαντικό. Είναι εθνική εξουσία και αρμοδιότητα η απόφαση για την ώρα. Ήδη σήμερα ισχύει αυτό το πράγμα. Και όπως υπόθηκε, έχουμε τρεις ζώνε ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή και αυτό δεν στρεβλώνει ούτε αναστατώνει σε καμία περίπτωση την εσωτερική αγορά. Θα το εκτιμούσα λοιπόν πολύ αν μπορούσατε πραγματικά να το λάβετε αυτό υπόψη σα κάθε φορά που σχολιάζετε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και παρότι βλέπω ότι υπάρχει ένας, κάπως, ένας κάποιος σκεπτικισμός στις παρατηρήσεις σας, βλέπω τελικά ότι οι περισσότεροι είστε έτοιμοι να εγκρίνετε την πρόταση της Επιτροπής σας βάσει της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έλαβε χώρα πέρυσι. Θεωρώ ότι στέλνουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό διότι ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο αυτό και ουσιαστικά η συμμετοχή ήταν 10 ε, φορές μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή Ευρωπαίων πολιτών σε οποιαδήποτε άλλη διαβούλευση, σε οποιαδήποτε άλλη φορά του ζητήσαμε να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένε ερωτήσει. Άρα ενδιαφέρονται για το ζήτημα αυτό οι Ευρωπαίοι πολίτε και εμεί είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε. Το ζήτημα λοιπόν αυτό θα μπορούσε να φανεί πιο πολύπλοκο τελικά από ό,τι θα περίμενε κανείς εκ πρώτης όψεως. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη διάκριση εξουσιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Αυτό όμω ισχύει ήδη σήμερα. Δεν είναι κάτι το οποίο επινόησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σώνει και καλά για την πρόταση αυτή. Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε και να σεβαστούμε, να τηρήσουμε αυτή τη διάκριση εξουσιών κάθε φορά που θα πάρουμε στο μέλλον αποφάσεις. Όπως σας είπα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ότι θα υπάρχει μια στενή παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της οδηγίας και θα συνεργαστούμε προκειμένου να αποφύγουμε οποιοδήποτε αναστάτωση για τους Ευρωπαίους πολίτες ή για τους οικονομικούς φορείς. Και Προσωπικά πραγματικά είμαι πεπισμένη ότι κάθε κράτος μέλος γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώ έχει το ζήτημα και γι' αυτό ακριβώ το λόγο οι αποφάσει που θα λάβουν τα κράτη-μέλη του επόμενου μήνε θα είναι πιστεύω συντονισμένε. Πάντω παραμένει εθνική επιλογή. Πρόκειται να είναι μια επιλογή των κρατών μελών. Το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να διασφαλίσει ότι όλοι θα αποφασίσουμε ταυτόχρονα, την ίδια χρονική στιγμή δηλαδή. Και προφανώ θα προβλέψουμε ώστε να κινηθούν έτσι τα πράγματα. Και μάλιστα θα ενθάρρυνα και τα κράτη-μέλη προκειμένου να γνωρίζουν τελικά ποια επίσημη ώρα να επιλέξουν, να διεξάγουν και αυτά εθνικές διαβουλεύσεις και θα δοθεί στα κράτη-μέλη ο παρέτο χρόνο προκειμένου να κάνουν τη διαβούλευση αυτή με τρόπο δημοκρατικό και ανοιχτό και διαφανή. Εν κατακλείδη, για μία ακόμη φορά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω να σας ευχαριστήσω όλους σας και την εισηγήτρια και τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές διότι αφιερώσετε τόσο πολύ χρόνο στο ζήτημα αυτό και εγκρίνοντας την έκθεσή σας θα, μπορέσετε να ξεκινήσετε τις διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές και πιστεύω ότι θα οδηγηθούμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα στα πλαίσια της Φιλανδικής Προεδρίας. Καλή τύχη λοιπόν για αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε την Επίτροπο. Και τώρα θα ακούσουμε την απάντηση της συγγήτριας. Μαρίτα Ουλουτσκόκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που αξιοποίησαν την ευκαιρία και ξέφρασαν τις απόψεις τους για αυτό το θέμα. Η συζήτηση ήταν πολύ ζωηρή, πολύ ενδιαφέρουσα. Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα και πιο ζωηρή ε, που έχω παρακολουθήσει εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό αποδεικνύει δε ότι το θέμα αυτό άπτεται και αφορά άμεσα τις ζωές των ανθρώπων. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που η Επιτροπή Μεταφορών, που έχει πάντοτε στραμμένο το, την προσοχή, στραμμένη την προσοχή της στις καθημερινές προτάσεις, ποτέ δεν θα υπέβαλε πρόταση η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρέβλωση ε, ή σε διατάραξη της λειτουργίας της ενιαίας ε, αγοράς. Δεν ξέρω αν είχε ζητηθεί η έκθεση αυτή να συνταχθεί από την Επιτροπή Πολιτισμού, μπορεί τα πράγματα να ήταν και λίγο διαφορετικά. Όμως ζητήθηκε από την Επιτροπή Μεταφορών. Και αυτό ε, μας οδήγησε σε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία και συνεκτιμήσαμε, όπως είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τελικά τα επιθυμητά αποτελέσματα, ωφέλη όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας. Και έτσι καταλήξαμε στην πρότασή μας ε, ώστε να καταλήξουμε σε κατάργηση των αλλαγών της ώρας που θεωρώ ότι είναι μια προσγειωμένη πρόταση η οποία θα είναι αυτή που θα μας οδηγήσει σε, σε εξοικονόμηση χρημάτων, θα ωφελήσει την υγεία ανθρώπων και ζώων και γενικά θα έχει συνολικά πολύ θετικέ επιπτώσει στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για τη συζήτηση αυτή που έγινε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, ανέδειξε διάφορε διαστάσει και νομίζω ότι αποδεικνύει η συζήτηση αυτή ότι ω Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να έχουμε πολύ θετικέ ιδέε και για άλλου τομεί. Ευχαριστήσουμε και την εισηγήτρια. Ολοκληρώνεται η συζήτηση στο σημείο αυτό και Θα γίνει σύντομα και η ψηφοφορία. Να ευχαριστήσουμε την Επίτροπο Μπούλτσα που ήταν σήμερα μαζί μας. Και περνάμε τώρα στην κοινή συζήτηση όσον αφορά την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε εδώ πέρα δύο εκθέσεις από τον κύριο Μπούσεκ, μία έκθεση από τον κύριο Πέτερσεν και μία έκθεση από τον κύριο Τζανονάτο. Θα ήθελα να δώσω καταρχάς τον λόγο στον κύριο Βέρνερ για τέσσερα λεπτά. Στην κυρία Βέρνερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κανιέτε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την τιμή σήμερα να ε, αντικαταστήσω τον συνάδελφο Μπούζεκ που είναι ο εισηγητής του Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά. Ο κύριος Κάρινς που ήταν αρχικός εισηγητής ε, της πρότασης αυτής ε, είναι πλέον Πρωθυπουργό τη Λετωνία. Εκείνο είχε ξεκινήσει τη διαδικασία και τη διαπραγμάτευση με τα άλλα δύο θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι εδώ βεβαίω, αλλά παρόλα αυτά θέλω να τον ευχαριστήσω για το έργο του και για τη συνεργασία που είχαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει ε, υπέβαλε τον Νοέμβριο του 2016 τι προτάσει τη για την καθαρή πράσινη ενέργεια και οι δύο προτάσει τη για την οργάνωση τη αγορά ηλεκτρική ενέργεια είναι οι πιο ολοκληρωμένε του πακέτου. Ποιο είναι το θέμα. Ο κανονισμός θεσπίζει νέους κανόνες για την ε, ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει υποστεί πολλές μεταβολές ε, τα τελευταία χρόνια. Ο ρόλος ε, των οικονομικών φορέων, ε, των ε, παραγωγών, των καταναλωτών επίσης έχει αλλάξει και αυτό είναι αναγκαίο να υπάρξει μια νέα διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ηλεκτρικής, αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για να είναι εφικτή η μετάβαση, η ενεργειακή. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις, πρέπει να γίνει νέο σχεδιασμός, πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία περιφερειακή μεταξύ των εθνικών αγορών. Ο καταναλωτής επίσης στο νέο σύστημα αποκτά κεντρικό ρόλο. Οι καταναλωτές, οι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας πλέον θα μπορούν ενεργά να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της, ηλεκτρικής, της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Για να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, οι πελάτες θα έχουν στο μέλλον τη δυνατότητα να λαμβάνουν λογαριασμούς Ηλεκτρική ενέργεια που θα είναι πέρα για πέρα κατανοητή σε όλους. Γιατί ξέρετε, δεν θα εκπλήξει κανέναν αν σας πω ότι μέχρι σήμερα πρέπει κανείς να διατρέχει και να φιλομετρεί σελίδε επί σελίδων λογαριασμών μέχρι να καταλάβει τι ακριβώς πληρώνει και γιατί το πληρώνει. Επίσης, θεσπίζονται πιστοποιήσεις σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε κάθε πολίτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να κατανοεί και να μπορεί να συγκρίνει τις, ε, τα διάφορα ε, τιμολογιακά συστήματα και να κάνει ενημερωμένες επιλογές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι θα πρέπει να προστατευτούν ιδίως οι ευάλωτοι, η ενεργειακή ένδια είναι μια πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το λόγο θεσπίζεται υποχρέωση των κρατών μελών στο εξή να παρακολουθούν αν επαρκούν ή εθνικοί κανόνες που έχουν θεσπίσει προκειμένου να προστατεύονται τα δικαιώματα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Ιδίω θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που με την εμπειρογνωμοσύνη τους συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτού, αυτής της διαδικασίας για αυτό το θέμα και θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά κύριε Κανιέτε για την πολύ επικοδομητική στάση που τηρήσατε πάντοτε στις διαπραγματεύσεις. Η Αυστριακή Προεδρία επίσης συνέβαλε σοβαρά ώστε αύριο επιτέλους να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να ψηφίσουμε επί αυτής της έκθεσης. Χρειαστήκαμε μόλις έξι τριμερείς διαλόγους, την πρώτη τελευταία φορά 17 ώρες και την τελευταία φορά 16 ώρες βεβαίως. Παρόλα αυτά είναι τεράστιο το έργο ε, ήταν πραγματικά ε, τιτάνιο το έργο, το, το τιτάνια επιτυχία το γεγονός ότι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε επί Αυστριακής Προεδρίας την συζήτηση και την διαπραγμάτευση αυτή. Θέλω επίση να ευχαριστήσω του συναδέλφου για την εμπιστοσύνη του για την επικοδομητική του συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω του εργαζόμενους τη γραμματέία τη Επιτροπή Ήτρε, όλου του Κοινοβουλίου, του πολιτικού συμβούλου των πολιτικών ομάδων και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα τους βοηθούς για όλα όσα έκαναν. Θεωρώ ότι από κοινού βάλαμε ένα πολύ, κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα που θα μας οδηγήσει στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος Πέτρεσεν, εισηγητής και αυτός για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όλους όσοι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις στην Κομισιόν, το Συμβούλιο των Υπουργών και προφανώς ε, τους εξαίρετους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περάσαμε πολλές ώρες διαπραγματευόμενοι και πολύ συχνά με στη νύχτα. Τα αποτελέσματα όμως μας κάνουν περήφανους. Τουλάχιστον θα έπρεπε να μας κάνουν περήφανους. Γιατί είμαστε ένα βήμα πριν τον γκρεμό, πριν την ήττα πριν το να χάσουμε αυτή τη μάχη για την κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Οι πολίτες κατεβαίνουν στον δρόμο και απαιτούν δράση. Έχουμε δει του εφήβου μας να διαδηλώνουν σε όλη την Ευρώπη ζητώντας ένα καλύτερο κλίμα και λύσεις για τα προβλήματα, τα περιβαλλοντικά προβλήματα που οδηγούν, σε, οδηγούν χιλιάδες ανθρώπους στο, στην απόδραση από ξηρασίες ή από πλημμύρες. Στενά εθνικά συμφέροντα παρεμποδίζουν την ε, αναγκαία μετάβαση. Το ενεργειακό πακέτο δεν λύνει όλα τα προβλήματα βέβαια. Ε, η, παρόλο που η ηλιακή ενέργεια, η, η αιωλική ενέργεια είναι ευθυνότερες από τον άνθρακα, η μετάβαση δεν γίνεται γρήγορα. Έχουμε δει ότι η αιωλική ενέργεια μπορεί να φέρει φθηνό ρεύμα στις μπρίζες μας. Παρ' όλα αυτά, πολλές κυβερνήσεις εξακολουθούν να χρησιμοποιούν άνθρακα για την παραγωγή ενέργεια σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να ενισχύσει αυτή την πρόταση, αλλά πολλέ εθνικέ κυβερνήσει προσπαθούν να την ε, μετριάσουν. Προσπαθούμε λοιπόν λοιπόν να δώσουμε περισσότερους, ε, περισσότερες αρμοδιότητες και πόρους στον Acer, τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Και λέμε ότι ο Acer θα πρέπει να μπορεί να έχει και ίδια έσοδα μέσω τελών για ορισμένες δραστηριότητές του. Γιατί όταν αφήσουμε τα κράτη-μέλη να τιμολογούν ε, όλες τις δραστηριότητες σχετικές με την ενέργεια, οδηγούμαστε σε αδιέξοδο. Έχουμε εντάξει την ε, βιώσιμη ενέργεια στην, στις διασυνορικές μας σχέσεις, αλλά ε, πολλές κυβερνήσεις ακόμα υστερούν. Οι υπουργοί στο Παρίσι, όταν υπέγραψαν τις ωραίες ε, δηλώσεις έκαναν πολύ καλά, αλλά όταν κάθονται γύρω-γύρω από ένα τραπέζι Βρυξέλλε, δεν κάνουν το ίδιο. Την περσμένη εβδομάδα ε, οι αρχοί κρατών κυβερνήσεων ε, δεν κατάφεραν να υποστηρίξουν το σχέδιο για την ε, ενεργειακά ουδέτερη Ευρώπη του 2050. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, να επενδύσουμε περισσότερα χρήματα στην έρευνα Και θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε αυτούς τους πόρους αν ε, φορολογήσουμε τα πλαστικά ε, και τον άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ όλους για τις διαπραγματεύσεις και για την προσπάθειά τους. Σε δύο μήνες θα ζητήσουμε από τους πολίτες μας να ψηφίσουν. Μην το ξεχνάμε αυτό και μην αγνοούμε την απέτηση των πολιτών μα να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Αυτό μα ζητάνε τα παιδιά μα και τα εγγόνια μας. Ευχαριστούμε κύριε Πέτερσεν. Τώρα θα ακούσουμε τον άλλο εισηγητή, τον κύριο Τζανονάτο. Φλάβιο, έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όταν κάναμε τα πρώτα βήματα για αυτή τη δέσμη μέτρων που είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ενεργειακή Ένωση, πριν από πολλούς μήνες δηλαδή, γνωρίζει ήδη από τότε ότι όλος ήταν ιδιαίτερα δύσκολο πολλά τα διαφορετικά συμφέροντα και πολλέ δυσκολίε και τα εμπόδια στον αφορά την ολοκλήρωση των ενεργειακών αγορών. Μολονότι λοιπόν ο, δύσκολο, ο δρόμος ήταν πιο δύσκολος από ό,τι περιμέναμε και μολονότι υπήρχε έντονη αντιπαράθεση απόψεων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους τριμερείς διαλόγους, καταφέραμε τελικά να καταλήξουμε σε κάποιες βελτιωμένες νομοθετικές συμβαστικές λύσεις. Στα πλαίσια της ετοιμότητας αντιμετώπισης του κινδύνου στον τομέα της ηλεκτρονικής ενέργειας θα πρέπει πραγματικά να λάβουμε υπόψη την πολύ σημαντική εργασία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα κάθε φορά που προκύπτει μία διακοπή της ηλεκτρικής ενέργειας ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα στο δίκτυο και ξέρετε ότι αυτό μπορεί να συμβεί λόγω των κλιματικών αλλαγών, λόγω μιας τρομοκρατικής επίθεσης, λόγω ιδιαίτερης υψηλής σύνδεσης και χρησιμοποίησης του δικτύου, τα κράτη-μέλη βρίσκονται εντελώς απομονωμένα και εναπόκεινται τελικά στην καλή θέληση που ενδεχομένω να δείξουν οι όμορε χώρε προκειμένου να ξεπεράσουν τα σημαντικά αυτά ενεργειακά προβλήματα. Αυτά είδαμε και τον Ιανουάριο του 2017 στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου επλήγησαν πολλέ ευρωπαϊκέ Καταλαβαίνετε όμως τα προβλήματα αυτά πραγματικά ζημιώνουν τελικά τον τελικό καταναλωτή, αυξάνουν τι τιμέ, αλλά ζημιώνουν και την οικονομία και τι βιομηχανίε. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε πλέον τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να μπορεί να παρέχεται ομαλά η ενέργεια προς όλους αυτούς που την έχουν ανάγκη και να μπορούμε ουσιαστικά να ξεφεύγουμε από ε, τα προβλήματα, τα εμπόδια τα οποία προκύπτουν σε εθνικό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προωθήσουμε την αμοιβαία συνεργασία και δυστυχώ μέχρι στιγμή η συνεργασία αυτή δεν ήταν επαρκή, επειδή δεν ακολουθεί το ίδια μεθοδολογία μεταξύ των κρατών μελών, είτε επειδή πολλέ φορέ υπήρχε πλεονάζουσα παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια ή επειδή δεν υπήρχαν οι απαραίτητε συμφωνίε αμοιβαία συνδρομή. Νομίζω ότι μέσω της νέα αυτής πρόταση κανονισμού μπορούμε τελικά να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση που θα λειτουργήσει υπέρ των κρατών μελών και να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ε, συνέβαλε με τρόπο καθοριστικό και αν δεν είχε αναλάβει το ρόλο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα είχαμε καταλήξει τελικά σε μία συμβαστική λύση. Περιμένω ότι θα καταφέρουμε να εγκρίνουμε την απόφαση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να έχουμε μια κοινή πλέον μεθοδολογία αντιμετώπιση των κινδύνων στον τομέα τη ηλεκτρική ενέργεια προκειμένου να βοηθηθούν όλε οι χώρε και προκειμένου τελικά να υπάρχει ένα ομοιογενέ ενιαίο μοντέλο αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των κρατών μελών και να μπορούν να βοηθούνται όχι μόνο οι επίσημες εθνικές αρχές, αλλά όλοι οι παρεμβαίνοντες, όλοι οι εμπλεκόμενοι στον ε, τομέα της ενέργειας παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα τα κράτη-μέλη μέσω του κανονισμού αυτού να τηρούν τους κανόνες αμοιβαία συνδρομής και να καταφέρουμε να βοηθήσουμε και τις χώρες εκείνες που δεν έχουν την απαραίτητη υποδομή ή που δεν υπάρχουν απαραίτητες διασυνδέσεις. Έχουμε το καθήκον να βοηθούμε οι μεν τους δε. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι υπάρχουν πιο συγκεκριμένα κριτήρια πλέον όσον αφορά τον, το ζήτημα της αποζημίωσης. Και πάλι εδώ πέρα προβλέπεται η διακριτική ευχαίρεια για τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Δεν θα πρέπει οι διαπραγματεύσεις αυτές να αποτελέσουν ένα μέσο προκειμένου να ταραχθούν, αν θέλετε, οι επιτευχθήσεις ισορροπίες σε σε άλλε πτυχέ αυτέ τη δέσμη μέτρων. Καταφέραμε να το ξεπεράσουμε και τον κίνδυνο αυτό χάρη στην πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με όλου του εισηγητές για όλα τα υπόλοιπα νομοθετήματα από τι αρμόδιε επιτροπέ. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μπούζεκ, ο οποίο συντόνισε τις εργασίες μα πολύ καλά. Να ευχαριστήσω τους σκιώδει εισηγητές για την εξαιρετική εργασία του, για τη συμβολή του σε όλα τα στάδια τη εργασία αυτή και να ευχαριστήσω βέβαια και τον Επίτροπο Κανιέτε. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Άριας ο Επίτροπος. Παρακαλώ. Κυρίε και κύριοι, με χαρά είμαι εδώ σήμερα για να συζητήσουμε τα τελευταία κομμάτια του πακέτου για την ενέργεια. Αυτές οι τέσσερις πράξεις, δύο κανονισμοί, μια οδηγία και οι κανόνες για τον Acer, είναι τα τελευταία κομμάτια του παζλ. Είναι το μεγαλύτερο νομοθετικό πακέτο που είχε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα ενέργειας. Ολοκληρώνουμε μια σύγχρονη, μια μεταρρύθμιση εξυγχρονισμού που μας προετοιμάζει για το μέλλον. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο που μας στήριξε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Μας επέτρεψε αυτό να εξασφαλίσουμε πολιτική συμφωνία το Δεκέμβρη. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους συζητητές. Ο Κάριντς, τον οποίο συγχαίρω που έγινε και πρωθυπουργός της Λετωνίας, τον και τον κύριο Πέτερσεν. Προφανώ και τον πρόεδρο Μπούσεκ και όλου του πολιτικού συντονιστέ και του κοιόδη ηγητέ που αυτή η συμφωνία χωρί αυτού δεν θα ήταν δυνατή. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τη συμπληρωματικότητα και τη συνέπεια αυτή τη πρόταση. Ε, συμφωνήσαμε σε ένα πολύ φιλόδοξο πακέτο που θα μα προχωρήσει ένα ακόμα βήμα στην συμπλήρωση τη Ενεργειακή Ένωση. Ήταν μία ακόμα από τις προτεραιότητες της ε, Κομισιόν Juncker, τις οποίες ε, εγκρίνατε πριν από πέντε χρόνια. Αυτή η συμφωνία θα εξασφαλίσει ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πιο βιώσιμη, πιο ανταγωνιστική και πιο ασφαλής. Αυτοί οι κανόνες είναι καλοί για τους καταναλωτές, για τον πλανήτη και για την οικονομία. Από την πλευρά του καταναλωτή, για πρώτη φορά ε, ενεργειακή νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει τόσο πολλά μέτρα προστασία των καταναλωτών. Οι καταναλωτέ μπορούν πλέον να γίνουν δραστήριοι παίκτες που θα συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση. Αυτό είναι απόλυτο απαραίτητο. Η ενεργειακή μετάβαση δεν θα πετύχει εκτό και αν συμμετάσχουν οι πολίτε και η κοινωνία. Μέσω αυτή τη νομοθεσία οι καταναλωτέ θα έχουν καλύτερη ενημέρωση. Ε, οι λογαριασμοί θα γίνουν πιο σαφείς πιο ξεκάθαρη. Θα είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο να αλλάξουν οι κατανοητέ πάροχο. Ενδεχομένως και σε 24 ώρες από το 2026 και μετά. Ε, θα έχουμε εργαλεία εύκολης σύγκριση έτσι ώστε οι πολίτε να κάνουν πιο ενημερωμένοι, να πάρουν πιο ενημερωμένοι τι αποφάσεις τους. Σε ό,τι αφορά την εναλλακτική επίλυση διαφορών, γίνεται μια δήλωση για το πώ θα αξιολογήσουμε τέτοιου μηχανισμού. θα επιτρέψουμε στους πολίτες μας να ε, κάνουν τις πιο ανταγωνιστικές επιλογές έτσι ώστε να εξοικονομούν χρήματα. Επίσης οι καταναλωτές θα μπορούν να παράγουν, να αποθηκεύουν και να πολλούν ενέργεια στην αγορά μόνοι τους ή συλλογικά. Για πρώτη φορά αναγνωρίζουμε τις ενεργειακές κοινότητες χρηστών. Με αυτόν τον ε, τρόπο ε, εφαρμόζουμε τη δέσμευσή μας ο πολίτης να είναι στο κέντρο των πολιτικών μας. Αυτές αυτοί οι καινούργιοι κανόνες θα καταστήσουν τις αγορές πιο ευέλικτες και πιο ε, ενωμένες. Ε, αυτό θα έχει πολύ θετικές επιπτώσεις στην οικονομία. Θα μπορούν να υιοθετηθούν πιο, γρήγορες, πιο γρήγορα καθαρές ε, ευέλικτες λύσεις. Και αυτό θα δημιουργήσει και θέσεις εργασία. Έχουμε ενισχύσει την περιφερειακή συνεργασία για τους κανόνες ε, που επιτρέπουν η υπερβάλλουσα ε, ενέργεια να μπορεί να τεθεί ε, σε διαπραγμάτευση και τη εμπορίας. Ο καινούριο, το καινούριο πλαίσιο για το μηχανισμό μηχανισμούς δυναμικού θα οδηγήσει σε πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας η Κομισιόν ε, θα κάνει μια δήλωση στα πρακτικά σε ό,τι αφορά ε, την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών σχεδίων. Επίσης, μια άλλη δήλωση σε ό,τι αφορά τον ορισμό των διασυνδετών. Θα υπογραμμίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στο φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια. Τέλος, δεδομένου ότι η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική, πρέπει να εξασφαλίσουμε και την ασφάλεια εφοδιασμού για την οικονομία και του πολίτε μα. Ο κανονισμό προετοιμασία εναντίον των κινδύνων θα καταστήσει το σύστημά μα πιο σταθερό και θα εισάγει την έννοια τη ε, ε Τώρα, τι φέρνει στο περιβάλλον και στη βιωσιμότητα αυτό το καινούριο σύστημα. Έχουμε πετύχει, συμφωνήσει φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους και το καινούριο σύστημα θα συνεισφέρει στην επιτυχία αυτών των στόχων. Προκειμένου να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις του Παρισιού, οι αγορές μας θα είναι πιο ευέλικτες και θα μπορούν να προσαρμοστούν πιο εύκολα. Ο μηχανισμός μας θα διασφαλίζει ότι οι λύσεις μας για την, ενέργεια και ασφάλεια του, του ενεργειακού αφοδιασμού συνάδουν με τους περιβαλλοντικούς μας στόχους. Όλα αυτά θα βοηθήσουν τη βιομηχανία και την οικονομία της Ευρώπης να πάρει το σωστό δρόμο, τη σωστή κατεύθυνση. Θα μειώσουμε όμως και την τοπική μόλυνση. Οι νέοι μα κανόνες θα ε, ε, κοιτάνε και προς άλλα σημεία του κόσμου. Όλο αυτό το πακέτο μέτρων μας καθιστά το πρώτο μέλος τη Συμφωνία του Παρισιού που έχει υιοθετήσει πλέον όλη την απαραίτητη εσωτερική νομοθεσία ε, προκειμένου να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις τη. Ταυτόχρονα μα θέτει σε πολύ καλή θέση στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις. Άρα λοιπόν εμείς ανοίγουμε το δρόμο για να ακολουθήσει ο υπόλοιπο κόσμος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη Επιτροπή Περιβάλλοντο Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια Τροφίμων, ο κύριο Ζωρίνιο έχει το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπολείπεται των υποχρεώσεών της και των δεσμεύσεων της ε, ε, κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Η Ενεργειακή Ένωση όμως κινείται προς την άλλη κατεύθυνση. Συγγνώμη κύριε Σορίγιο. Κύριε Ζωρένιο, συγγνώμη. Ε, οι δύο κύριοι εκεί πάνω ψηλά, μπορείτε να σταματήσετε σας παρακαλώ ή να βγείτε εκτός εθούσης. Μας ενοχλείτε. Ενοχλείτε τη συζήτηση. Σας παρακαλώ είτε να καθίσετε και να σταματήσετε τη συζήτηση, είτε να βγείτε εκτό αιθούση και να συνεχίσετε τη συζήτηση εκεί. Σα ευχαριστώ. Κύριε Ζωρίνιο, με συγχωρείτε. Να ξεκινήσω από την αρχή. Ναι, ναι, ωραία. Κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υστερεί σε σχέση με τι υποχρεώσει τη ε, σε ό,τι αφορά την σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα. Όμω, υπάρχουν και εξαιρέσει η ενέργεια και η ψηφιακή ένωση είναι αντίθετα παραδείγματα και γι' αυτό το λόγο συζητάμε τα συγκεκριμένα νομιστικά κείμενα. Όμως δεν αρκεί να σιωνιώνουμε πρόοδο. Πρέπει να ηγηθούμε στον κόσμο ε, στην ενεργειακή μετάβαση υπέρ των πολιτών μας και υπέρ μιας ε, καθαρής και ευθύνης ενέργειας. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη μετάβαση με διαφάνεια στην αγορά και να δώσουμε προτεραιότητα στην παραγωγή ενέργειας με ανανεώσιμε πηγέ. Η ενιαία εσωτερική αγορά δεν μπορεί να είναι συνώνυμο της αγορά χωρί κανόνες. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αδικίες με τρόπο διαφανή, με ασφάλεια και με καινοτομία. Θα πρέπει να δώσουμε ένα καινούριο φως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στου πολίτες τη. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στους ε, εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Λάγεν. Έχετε 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι χρειαστήκαμε σχεδόν τρία χρόνια για να εγκρίνουμε το πακέτο αυτό. Και αυτό δεν οφειλόταν βεβαίως ε, ούτε στο Κοινοβούλιο ούτε στην Επιτροπή, αλλά κατά κύριο λόγο στο Συμβούλιο που μπλόκαρε τη διαδικασία. Μπορούμε να είμαστε όμως ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα που επιτύχαμε για στις διαπραγματεύσεις ε, για τον ε, Acer θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο Πέτερσεν που ηγήθηκε της δικής μας αποστολής όμως ήδη από τις 20 Φεβρουαρίου του 2018 είχαμε εγκρίνει στην Επιτροπή την έκθεση χρειαστήκαμε σχεδόν ένα χρόνο για να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο. Γιατί η Επιτροπή ήθελε να δώσει περισσότερες αρμοδιότητες στον Acer, το Συμβούλιο καθόλου. Καταφέραμε λοιπόν να επιτύχουμε ο ρόλος του Acer να συμβαδίζει με τις εξελίξεις της εποχής μας. Βρισκόμαστε πλέον σε αυτό το σημείο όπου σήμερα ο Acer έχει περιορισμένες μεν μεγαλύτερες δε σε σχέση με το παρελθόν αρμοδιότητες και αυτό θα, το, θα τις επιτυχάνει μέσω της παρακολούθησης των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων. Γι' αυτό και θέλω να τονίσω ότι η διαπραγμάτευση για τον Acer στέφτηκε με επιτυχία. Πρόεδρο, ευχαριστώ εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών ο η κυρία Βέρνερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο χρόνια εργαστήκαμε επί της μεταρρύθμισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη νέα διαμόρφωση θέτουμε τα θεμέλια για μια αποκεντρωμένη ασφαλή, βιώσιμη αγορά ενέργειας ώστε να επιτύχουμε την ενεργειακή μετάβαση. Βεβαίως η επιλογή των ενεργειακών πηγών αποτελεί ύψιστης και κεντρικής σημασίας. Οι ανανεώσιμες θα πρέπει να είναι το μέλλον και γι' αυτό ως επικεφαλής των διαπραγματευτών της δικής μου πολιτικής ομάδας εγώ τόνισα ότι θα πρέπει πρώτα να ε, συνδέονται στη, στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη συνέχεια όλες οι άλλες. Βεβαίως θα πρέπει να καταργηθούν οι επιδοτήσεις στον άνθρακα. Εμείς ως σοσιαλδημοκράτες επίσης πετύχαμε οι ε, ευρωπαϊκές κοινο, ε, κοινοπραξίες πολιτών στον τομέα της ενέργειας να ε, την χάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης και να μην αποτυχάνουν ε, σε, λόγω εμποδίων τεχνητών που τους θέτουν οι μεγάλες εταιρείες. Σημαντικό είναι επίσης να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, κάτι που διασφαλίζεται και μέσα από τις ε, συγκριτικές ιστοσελίδες και τη δυνατότητα των πολιτών να αλλάζουν παρόχους μέσα σε 24 ώρες. Εγώ θα ήθελα βεβαίως ε, να είχαν αναλάβει σημαντικότερο ρόλο οι δημοτικές επιχειρήσεις ενέργειας. Δυστυχώς όμως αυτή η ιδέα δεν προκρίθηκε, δεν έτυχε της πλειοψηφίας και δυστυχώς είναι μια χαμένη ευκαιρία για μένα γιατί ιδίω στην ηλεκτρική κινητικότητα θεωρώ ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι κρατικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν, θα μπορούσαν να είναι εκείνες οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικότατα στην προώθηση αυτών των μορφών. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη που μου έδεξαν για την ιδιαίτερα επικοδημοτική συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστώ εκ μέρους των ε, φιλελευθέρων η κυρία Μιλινάρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να, να συγχαρώ όλους τους συζητητές για το γεγονός ότι κατακτήσαμε αυτό το ορόσημο για την ολοκλήρωση του πακέτου για την καθαρή ενέργεια που θα δώσει στους πολίτες μας ένα νέο σύστημα το οποίο θα δίνει καλύτερα απαντήσεις όσον αφορά τη διασυνδεδεμένη ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ως ε, σκιώδης για την ετοιμότητα εναντί των κινδύνων χαιρετή χαιρετίζω την πρόταση της Κομισιόν η οποία είναι αναγκαία όπως αποδείχθηκε και από την μη συντονισμένη απάντηση που δόθηκε στην, στο κύμα ψύχους που έπληξε την Ευρώπη το 2017. Εργαστήκαμε λοιπόν σε διάφορα επίπεδα για να καταλήξουμε στην ε, υποχρέωση των κρατών μελών να συντονίζονται εκ των προτέρων η ο έγκυρος σχεδιασμός ε, θα εξασφαλιστεί μέσα από έγκυρους και προβλέψιμους κανόνες μέσω της θέσπισης ε, συστημάτων και καθεστώτων εκ των προτέρων. Θεωρώ ότι εξασφαλίστηκαν τρία βασικά στοιχεία. Αφενό, εξασφαλίζεται ενωσιακή προσέγγιση χάρη στην αξιολόγηση κινδύνου που θα εγκρίνεται από τον Acer και μέσω τη συμμετοχή των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων σε όλε τι φάσει σχεδιασμού. Επίση, εξασφαλίζεται διαφάνεια και παροχή κινήτρων για την κοινή χρήση δεδομένων, ταυτόχρονα εξασφαλίζοντα την εμπιστευτικότητα και ε, λόγω ε, της ε, δυνατότητας να επιλέγονται μη αγορές επιλογές μόνο ως έσχατη λύση. Αυτά μειώνουν τον κίνδυνο blackout, διακοπών ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύουν την ασφάλεια ε, των ενεργειακών πολιτών και εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία των κρατών μελών μας στον ενεργειακό τομέα. Θα ήθελα να ολοκληρώσω ευχαριστώντας όλους τους συζητητές, τους συνεισηγητές και τις διαπραγματευτικές ομάδες για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστώ εκ μέρους των ε, Πρασίνων ο κύριος Μαρτσελέση. Έχετε ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η μείωση του χρήση του άνθρακα είναι απόλυτη προσεραιότητα προτεραιότητα. Και αυτοί, αυτά τα νομοθετικά κείμενα κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. Ε, χαίρομαι που θα στηριχθούν οι ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ε, οι κοινότητες των καταναλωτών ε, με κατάργηση των επιδοτήσεων στον, στον άνθρακα. Ε, κανένας δεν θα πρέπει να, πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στο τέλος του μήνα και στο τέλος του κόσμου. Κάτι όμως παραπάνω πρέπει να κάνουμε για να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις του Παρισιού δεν θα πρέπει να δίνουμε άδεια για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και στην ε, Πολωνία για την ε, χρήση πηγών ενέργειας που μολύνουν το περιβάλλον. Οι πράσινοι θα, προσέξουν, θα παρακολουθήσουν πάρα πολύ την Κομισιόν, γιατί το χρωστάμε στην νεό, στους νέους. Κάθε εβδομάδα βγαίνουν στους δρόμους για να μας δώσουν μάθημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη Ευρωμάδα τη Αριστερά, η κυρία Κορνέλια Έρνστ. Έχει ένα λεπτό. Ναι. Νομίζω ότι στον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει κανείς να αναρωτηθεί. Το αποτέλεσμα αυτό επαρκεί για τις επόμενες δεκαετίες. Θα, συμφ... συνεισφέρει στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Προωθεί επαρκώς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια, έχει, χαρακτηρίζεται από κοινωνική δικαιοσύνη. Για μας πρέπει να σας πω ότι το ποτήρι είναι μισογεμάτο. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι υπάρχουν θετικές ε, προβλέψεις, αλλά ασκούμε κριτική στο γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς η ενεργειακή ένδια. Με πολύ ήπιε διατυπώσεις μόνο αντιμετωπίζεται. Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την ε, πανευρωπαϊκή ρύθμιση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως όσον αφορά την, αποδοχή, την αύξηση της αποδοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όμως βλέπουμε ταυτόχρονα ότι τα, κατα... τα δικόματα των καταναλωτών δεν εξασφαλίζονται επαρκώς. Θέλουμε να σταματήσει η επιδότηση του άνθρακα. Ωστόσο, με τις χωρητικότητες που υπάρχουν αυτές στη στιγμή, δυστυχώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί χρειαζόμαστε κάτι άλλο, μια προτεραιότητα σύνδεσης, όχι μόνο για τις μικρές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά για όλους. Αυτό δυστυχώς δεν, δεν έγινε κατορθωτό, παρόλο που εμείς ως αριστερά προσπαθήσαμε. Γι' αυτό θα έλεγα ότι το ποτήρι είναι ταυτόχρονα και μισογεμάτο και μισοάδιο. E Εκ μέρους του EFDD, ο κύριος Μπάλοκ. Έχετε ένα λεπτό. Yes, please. Thank you, Madam. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κρίση της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη είναι αποτέλεσμα ε, ανεύθυνων επιλογών της ε, Κομισιόν. Στη σημερινή έκθεση ε, αναφερόμαστε σε σημαντικά θέματα όπως ε, τα παράπλευρα αποτελέσματα των επιδοτήσεων. Ο κ. Ναλότο από την άλλη μεριά πιστεύει ότι η περαιτέρω εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας βοηθήσει να, βοηθήσουμε, θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε μελλοντικές κρίσεις ενέργειας στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικέντρωσε την ενεργειακή της πολιτική σε ακριβές και μη αξιόπιστες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, αυτό υποσκάπτει την ανταγωνιστικότητα και στέλνει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε άλλες χώρες εκτός Ευρώπης ε, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι θέσεις εργασίας και οι επενδύσεις. Ελπίζω ότι το Ηνωμένο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακυρώνοντας όλες, όλα τα κομμάτια της ε, πολιτικής ε, περιβάλλοντος και ενέργειας. Έχουμε την ευκαιρία να βγούμε ξανά στον πραγματικό κόσμο και να επενδύσουμε σε αξιόπιστες πηγές ενέργειας όπως το άνθρακας και η πυρηνική ενέργεια εκμεταλλευόμενοι και εθνικές πηγές ενέργειας ε, όπως το σχιστολιθικό αέριο. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους του ENF η κυρία Λεσβαλιέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σημαντική ενέργεια για τους πολίτες, για τις βιομηχανίες, για τις μεταφορές και αποτελεί μία από τις στρατηγικές πολιτικές ενός κράτους μέλους. Αν εμεί θεωρούμε ότι η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών είναι απαραίτητη και ευκταία, από την άλλη εθνική κυριαρχία είναι πάρα πολύ μεγάλης σημασίας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε τι κλιματικέ αλλαγέ και να βοηθήσουμε του καταναλωτέ. Στην πραγματικότητα όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δημιουργήσει μια τεράστια εσωτερική αγορά ηλεκτρική ενέργεια, όπου υπονομεύεται η εθνική πτυχή και οι εθνικέ αγορέ το να μπορούμε να διαχειριστούμε μόνοι μας την πλεονάζουσα παραγωγή ή την ιστερούσα παραγωγή σε συνεργασία με τους γείτονές μας ή και να καταφέρουμε να προσαρμόσουμε την παραγωγή μας στις νέες τεχνολογίες αποτελεί ουσιαστικά μία στάση καθαρά εθνική ένα κράτο μέλο από μόνο του, και αυτό συνέβαινε όλε τι τελευταίε δεκαετίε, αποφασίζει για τα ζητήματα αυτά. Δογματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει τώρα να επιβάλλει νέε αποφάσει, οι οποίε ουσιαστικά εκμηδενίζουν εντελώ οποιαδήποτε εθνική κυριαρχία στον τομέα τη διαχείριση ηλεκτρική ενέργεια. Και αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή σε όλε τι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη μόνα του και ελεύθερα θα πρέπει να αποφασίζουν πότε θα συνεργάζονται και με ποια κράτη-μέλη και δεν θα πρέπει να αναγκάζονται να, δεν θα πρέπει να, αναγκάζονται να ακολουθούν τι επιθυμίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει μια πλήρη απελευθέρωση τη αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Α μην ξεχνάμε τα πολύ αρνητικά παραδείγματα που έχουμε από χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Στι περισσότερε περιπτώσει, τρίτε αυτέ χώρε οδηγήθηκαν, οδηγήθηκαν σε απόλυτη αποτυχία. Καθένα από τα τέσσερα αυτά κείμενα της δέσμης μέτρων αποτελεί ουσιαστικά έναν ακρογωνιαίο λίθο για τη δημιουργία της περίφημης αυτής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελεί ένα πετραδάκι προκειμένου να καταρακωθεί ακόμα περισσότερο οποιαδήποτε να απομείνουν σε εθνική κυριαρχία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Α μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διεθνοποιήσει την ηλεκτρική ενέργεια, να την ανοίξει στον αχαλήνοτο εξωτερικό ανταγωνισμό. Α μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η εθνική κυριαρχία. Τα κράτη-μέλη θα μπορούν σε εθνικό επίπεδο να αποφασίζουν για την ενεργειακά ζητήματα και να αποφασίζουν πότε και με ποια κράτη-μέλη θα συνεργαστούν. Περνάμε στου επόμενου ομιλητέ. Ο κύριο Μπλάνκο Λόπε έχει στη διάθεσή του ένα λεπτό. Ε, με την συζήτηση για τρίμηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ε, ολοκληρώνουμε την, ε, το πακέτο ε, της Ενεργειακής Ένωσης. Θέλω να σας συγχαρώ κύριε Επιτροπέ για την εργασία της Κομισιόν αλλά να αναγνωρίσω επίσης και το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Στο ύψος της πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε για το μέλλον. Χρειαζόμαστε ενεργειακή νομοθεσία σύμφωνη με τις ε, συμφωνίες του Παρισιού και με την τεράστια πρόκληση της ανθρωπότητας που είναι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η μεγαλύτερη ένταξη των ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ε, ο πιο ισχυρός ρόλος των καταναλωτών, ο ρόλος Τη Ευρωπαϊκή Ένωσης για την καταπολέμηση της ενεργική φτώχειας. Όλα αυτά μας κάνουν παγκόσμιο παίκτη, ισχυρό παίκτη ε, και μας δίνουν μια νομοθεσία ισχυρή που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των καιρών. Θα πρέπει να, είμαστε, να νιώθουμε περήφανοι ως Ευρωπαίοι για τη δουλειά που έχουμε κάνει και να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερα γιατί η πρόκληση είναι τεράστια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σκλέρ, για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ως ασκιώδης εισηγητής για τον ε, κανονισμό για τον Οργανισμό Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργεια, τον ACER, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πέτρεσεν για όλε τι προσπάθειε που κατέβαλε για τι πολύ ε, θετικέ διαπραγματεύσει. Μπορεί να μην έχουμε πετύχει ακόμα του στόχου μα πλήρω, αλλά έχουμε καταβάλει σημαντικέ προσπάθειε προκειμένου να έχουμε αποτελεσματικέ ενεργειακέ πολιτικέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη συνολική δέσμη μέτρων που προωθούμε. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω και δεν νομίζω ότι το κάλυψαν οι συνάδελφοι έχει να κάνει με τι αγορέ ηλεκτρική ενέργεια και πιο συγκεκριμένα με το ζήτημα τη εφαρμογή. Ο επίτροπο Κανιέται πριν από λίγο αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό πολλές φορές και το έχει θίξει πάρα πολλές φορές όταν ήρθε στην Επιτροπή μας. Η Ενεργειακή Ένωση είναι κάτι το οποίο πρέπει να εφαρμόσουν, να ελοποιήσουν τα κράτη-μέλη, διότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ήδη σήμερα υφίσταται το εξή ζήτημα πώς μπορεί ένα κράτος μέλος από μόνο του να εφαρμόσει αυτή την ευρωπαϊκή δέσμη μέτρων. Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι, αν θέλετε, τα εμπλεκόμενα ταμεία, τα μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να εφαρμόσουμε στην πράξη τα νομοθετήματα αυτά. Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή τον κύριο Πέτρεσον και τους κοιόδης ηγητές για την πολύ καλή δουλειά τους. Ε, θέλω επίσης να εκφράσω ότι τα συγχαρητήριά μου για το ρόλο της Κομισιόν και της Αυστριακής Προεδρίας. Ο Acer είναι πολύ καλός, ε, θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ισχυρό, πιο διαφανή και τα, ε, κέντρα τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού επίσης θα παίξουν σημαντικό ρόλο ε, όταν ε, οι ρυθμιστικές αρχές μεταφοράς ενέργειας θα λαμβάνουν τις αποφάσεις τους. Χαίρομαι που αποφασίσαμε πως ο οργανισμός χρειάζεται καλύτερη χρηματοδότηση και πιο πολύ προσωπικό. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρασνοντεύσκη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια άλλη διάσταση του θέματος, χωρίς να επανέλθω σε όσα έχουν ήδη συζητηθεί και ήδη ακουστεί. Εγώ θέλω να στρέψω το βλέμμα μου στο μέλλον και στο επικείμενο νομοθετικό έργο που μας περιμένει στο πλαίσιο αυτού του ανεργειακού πακέτου. Νομίζω ότι είναι πλέον καιρός να θεσπίσουμε πραγματικές προϋποθέσεις για μια πραγματικά δίκαιη ενεργειακή μετάβαση προτού προχωρήσουμε σε περαιτέρω υλοποίηση φιλόδοξων στόχων για το κλίμα. Προτού πούμε ότι θα επιδιώξουμε μια πραγματικά ε, ουδέτερη από άποψη άνθρακα Ευρώπη έως το 2050 θα πρέπει να αξιολογήσουμε πραγματικά τους κινδύνους που προέρχονται από τα ορυκτά καύσιμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο κτλ. Πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν σε περιοχές που θα εγκαταλείψουν την ηλεκτροπαραγωγή με βάση τον ε, ε, άνθρακα όπως η Νότια Βουλγαρία για παράδειγμα όπου είδαμε ήδη πολύ σημαντικές αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Αυτό πρέπει να αποφευθεί στο μέλλον στις επόμενες περιπτώσεις που θα έχουμε αντίστοιχες διαδικασίες θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια, η δικαιοσύνη της και στο επίκεντρο της προσοχής μας θα πρέπει να τεθούν τα νοικοκυριά εκείνα που απειλούνται ήδη από ενεργειακή ένδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Catch the Δύο μιλητέ έχουμε. Ο κύριο Κέλλη. Having been involved Είμαι πάρα πολύ ευτυχής γιατί στη διάρκεια της θητείας αυτής δουλέψαμε πάρα πολύ για το θέμα αυτό ε, πρώτα απ' όλα έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούμε με τη Συμφωνία ε, των Παρισίων και βεβαίως έτσι ώστε να περάσει η απαραίτητη νομοθεσία για την δέσμη για την ενέργεια. Δεύτερον, όταν και αν θέλει κανείς να χρησιμοποιήσει τις ανανεώσιμες ε, πηγές ε, ενέργειας είναι σημαντικό να λάβει υπόψη του όσο γίνεται περισσότερο όλες τις δυνατότητες ε, της ε, τεχνολογίας. Ε, πρέπει να σας πω ότι έχουμε στην χώρα μου οραματιστεί πολλούς τρόπους έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριο Σκαπούτο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε η νέα δέσμη θα δώσει την δυνατότητα ε, να ε, διευρυνθεί η διασυνοριακή αγορά ε, και η ηλεκτρική ενέργεια να είναι πιο σεβόμενη το κλίμα. Ενδυνάμωση επίσης των δικαιωμάτων των καταναλωτών μέσω πλέον σαφών αρχών, δυνατότητα και ύπαρξη εργαλείων που δίνουν τη δυνατότητα σύγκρισης, καθώς επίσης επίσης και τη διευκόλυνση αλλαγής εντός 24 ωρών προμηθευτού. Ωστόσο, το σχέδιο δεν φαίνεται αρκετά φιλόδοξο όσον αφορά την αυτοπαραγωγή με ταυτόχρονο ε, αυτοέλεγχο επίσης. Η δέσμη θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα από ένα κεντρικό ε, μοντέλο ε, καυσίμων σε ένα αποκεντρωμένο ευρύ μοντέλο. Ο στόχος λοιπόν θα έπρεπε να είναι ε, να διευκολυνθεί οποιοδήποτε θέλει να κάνει αυτοπαραγωγή ενέργειας με ταυτόχρονη παροχή συμβουλών και περιορισμών όπου αυτό είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Επίτροπος παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Madam President, eh, honorable members, ladies and gentlemen. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία και γιατί στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τα θέματα αυτά, για τους φακέλους αυτούς υπήρξατε ιδιαίτερα αξιόπιστος ε, εταίρος. Η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση μπορεί να είναι πλήρως ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα και την έκβαση των διαπραγματεύσεων. Ευελπιστώ ότι αυτό θα καταδειχθεί και στην αυριανή ε, ψηφοφορία έτσι ώστε να έχουμε μια δέσμη για την ενέργεια που θα είναι ικανή να μας περάσει ικανοποιητικά στον 21ο αιώνα. Οι υποσχέσεις οι οποίες δόθησαν στους πολίτες πριν από πέντε χρόνια πλέον ε, ολοκληρώνονται και ε, επομένως ε, δείχνουμε στους πολίτες ότι περνούμε από τα λόγια στα έργα. Βεβαίως η συμβολή σας θα είναι αποφασιστική και θα χρησιμοποιήσουμε και τον κανονισμό διακυβέρνησης έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες και όσον αφορά και την κλιματική αλλαγή. Αυτή τη στιγμή ζητούμε και από τις κυβερνήσεις πλέον πλέον να αναλάβουν δράση. Και τώρα που ξεκινούν οι προεκλογικές εκστρατείες ε, ε, θα ήθελα να ζητήσω από όλους και από τους κύριους υποψηφίους, τους πέτσιν καντιντάτε να εξηγήσουν πολύ καλά τα θέματα αυτά αποζητώντας δέσμευση και υποστήριξη και από πλευρά των πολιτών. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπο και τώρα ο κύριος Βέρνερ ε, θα έπρεπε να πάρει το λόγο κανονικά, αλλά μου ζήτησε συγγνώμη εκ των προτέρων γιατί έπρεπε να παρευρεθεί σε μια παράλληλη συναντρίαση. Γι' αυτό δεν θα μπορέσει να πάρει το λόγο και το λόγο έχει ο κ. Πέτρεσεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσίασε το μεγάλο ενεργειακό πακέτο. Πλέον έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή και μπορούμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο κεφάλαιο μετά από πολλά χρόνια εργασίας και χαιρόμαστε που τα επόμενα πέντε χρόνια θα... Μάλλον τα τελευταία πέντε χρόνια καταφέραμε να καθορίσουμε την νομοθεσία αυτή με τον Επίτροπο η οποία θα έχει μεγάλο αντικτύπωση στην ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχει μεγάλο ε, ρόλο λοιπόν για τον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα επόμενα χρόνια σε ό,τι αφορά την νομοθεσία και την εφαρμογή, την υλοποίηση τη νομοθεσία. Ε, είναι πολύ σημαντικά λοιπόν όλα αυτά και στην ε, Ολομέλεια. Αυτά που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Τι μα δείχνουν ότι το Κοινοβούλιο επέμεινε για το επίπεδο φιλοδοξία και μάλιστα ύψωσε τον ε, πύχη. Αυτό θα πρέπει να το προωθήσουμε λοιπόν και στην προεκλογική εκστρατεία. Θα πρέπει λοιπόν ο κανονισμός ε, και η ΕΑΣΑ να εφαρμοστούν πλέον. Αυτά αποτελούν προϋπόθεση αυστηρή για να υπάρξει αυτή η πράσινη μεταμόρφωση. Είμαι βέβαιος ότι η Ευρώπη σε όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να είναι η ηγετική δύναμη. Θα πρέπει το 2050 να κοιτάξουμε το αργότερο τα θέματα για το διοξείδιο του άνθρακα και σε μια σχετική εκδήλωση στην Κοπενχάγη ήταν σαφές ότι και ο κόσμος επιθυμεί να αναλάβουμε δράση προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα να, ευχαριστώ, να ευχαριστήσω και την Επιτροπή και τους συναδέλφους για την καλή συνεργασία. Είναι πολύ καλό σημάδι. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος Εισηγητρής, ο κύριος Σανονάτο, Έχετε λόγο για δύο λεπτά κι αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω για να είμαι ειλικρινή σε αυτά που είπα πριν, ε, γιατί συμμερίζομαι τα όσα είπε μόλις ε, και ο Επίτροπος ε, Κανιέτε, αλλά συμμερίζομαι και τα περισσότερα από αυτά που ανέφεραν οι συνάδελφοί μου βουλευτές που μίλησαν για τα διάφορα σημεία. Όσον αφορά κάποιες λίγες επικριτικές παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα εδώ, και εδώ άκουσα με μεγάλη προσοχή, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι δεν αφορούν οι επικρίσεις αυτές αυτή τη συζήτηση, αλλά αφορούν περισσότερο το κατά πόσον είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί ενιαία αγορά ε, ενέργειας εδώ. Τώρα εμείς λέμε πώς και συζητούμε πώς θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί εμείς είμαστε ήδη πεπισμένοι και επομένως μετατίθεται, μετατοπίζεται η συζήτηση ε, προς ένα θέμα το οποίο δεν αφορά στην ουσία ε, την υποκατασκευή ε, αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ε, είδα ότι έφτασε και ο, Ντομινί, ο Γενικός Διευθυντής Ντομινί Κριστορή στην αίθουσα. Τον ευχαριστώ ε, ιδιαιτέρως, όπως ευχαριστώ και τον Επίτροπο Ρίας Κανιέτε και τους υπολείπους. Τον ευχαριστώ γιατί μου έδωσε να κατανοήσω και κατανόησε άμεσα και ο ίδιος κάποιους απαραίτητους μηχανισμούς. Ευχαριστώ και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά και μέχρι την επόμενη. Ευχαριστούμε τον εισηγητή και έτσι η κοινή συζήτηση ολοκληρώθηκε. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Έκθεση του κυρίου Τιδιέ σε ό,τι αφορά τι αντιπροσωπευτικέ δράσει για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων και των καταναλωτών. Ο κύριος Τιδιέ έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε Γιουροβάκα, τη συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και ένα χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαι ένα χρόνο μόλις μέλος και είμαι πάρα πολύ περήφανος που είμαι ε, συγγραφέας ενός ε, κειμένου που είναι τόσο σημαντικό για όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Αύριο θα μιλήσουμε για τις αντιπροσφυγές ε, κατά καταχρηστικών ε, πρακτικών από μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν ήταν εύκολο το καθήκον μου. Πολύ φοβόταν πως αυτή η αναθεώρηση θα δώσει ε, χώρο σε, αντιπροσ... σε ε, άδικες αγωγές, καταχρηστικές αγωγές και θα μας οδηγήσει στο να ακολουθήσουμε τα κακά κείμενα του Αμερικανικού συστήματος ε, πιο συγκεκριμένα. Να σας πω πως άλλοι φοβόντουσαν πως το κείμενο αυτό θα τελειώσει τελικά ως ένα τεράστιο, μια τεράστια δεξαμενή που θα χαθεί το άτομο γιατί κανείς δεν θα ήξερε ποιος θα χρησιμοποιήσει αυτές τις προσφυγές για να ζητήσει αποζημίωση από μια εταιρεία, γιατί για παράδειγμα η εταιρεία αυτή έχει μολύνει τον αέρα που εισπνεί και δεν θα χρησιμοποιούνται δεν κανείς να τις χρησιμοποιήσει γιατί θα είχαμε αλλοιώσει τη φύση του κειμένου που έχει σκοπό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο να προστατεύσει τα δικαιώματα του καταναλωτή. Στην πραγματικότητα μπορώ να πω πως εμείς φτιάξαμε ένα κείμενο πολύ στενά συνεργαζόμενοι με όλους τους σκιώδεις και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω πολύ θερμά για το εξαιρετικό πνεύμα συνεργασίας με μια πολύ λεπτή ισορροπία που αφενός συνδυάζει την αυξημένη ανάγκη προστασίας του καταναλωτή και αφετέρου δίνει την απαραίτητη ε, νομική ασφάλεια και βεβαιότητα σε εταιρείε. γιατί αποδεικνύει για πρώτη φορά πως και τα δύο μπορούν να επιτευχθούν, δηλαδή και ασφάλεια και προστασία. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα εγκρίνουμε το κείμενο αυτό μερικές εβδομάδες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές και αυτό είναι μια εξαίρετη απόδειξη του τι μπορούμε να κάνουμε όταν συνεργαζόμαστε, όπου γίνεται πολύ χρήσιμη ε, στην καθημερινότητα καθενός ε, από τους συμπολίτε μας η Ευρώπη. Θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα συλλογικών προσφυγών, όπου ένας επιβάτης, ένας που αγοράζει αυτοκίνητο, ένας που αγοράζει πλυντήριο θα έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον μιας ε, ε, καταχρηστικής πρακτικής είτε αυτού που του έχει πωλήσει τη λευκή συσκευή είτε ε, του, της εταιρεία που έχει κατασκευάσει το αυτοκίνητό του είτε εναντίον της αεροπορικής εταιρεία. και θα μπορούν με τον τρόπο αυτό να λάβουν και κάποια αποζημίωση για τη βλάβη την οποία έχουν υποστεί. Έτσι, για να νομιμοποιηθεί αυτή η συλλογική προσφυγή, έχει βασιστεί σε συγκεκριμένες αρχές και παραμέτρους. Αυτή η προσφυγή δεν θα υποκαταστήσει αυτές οι οποίες υπάρχουν ήδη σήμερα σε κάποια κράτη-μέλη και θα σεβαστεί τις, ε, τις εθνικές παραδόσεις στις προσφυγές ε, με όμως τη δημιουργία νέων τέτοιων ε, δυνατοτήτων στα εννέα κράτη-μέλη που δεν είχαν Επίσης, η αποζημίωση επιστρέφει στον καταναλωτή. Δηλαδή, είναι ένα όχημα που θα επιτρέπει στον καταναλωτή να βρει το δίκαιο του, χωρίς κανείς άλλος να κερδίζει οτιδήποτε. Και για να αποφύγουμε τις καταχρήσεις, είπαμε πως η ο ιτηθής διάδικος θα πληρώνει τα έξοδα, αλλά δεν μπορεί κανείς να λάβει διπλή αποζημίωση για την ίδια βλάβη. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλώ να υπερψηφίσουμε αύριο τη μεταρρύθμιση αυτή. Γιατί το κείμενο αυτό δεν ε, ε, εξυπηρετεί κανένα λόμπι, καμία ιδεολογία, κανένα συμφέρον. Απλώς προστατεί, προσπαθεί να προστατεύσει τα δικαιώματα καθενός από όλους τους καταναλωτές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντίτιε. Δεν βλέπω τον κύριο Ντέιγιον στην αίθουσα, οπότε θα δώσω το λόγο στην κυρία Γιούροβα, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Πρόεδρε, ε, αξιότιμα μέλη, θα ξεκινήσω ευχαριστώντα τον κύριο Τζιτζιέ που ω εισηγητή έκανε τόσο καλή δουλειά στην πρόταση αυτή, όπω επίση και όλου του υπόλοιπου συναδέλφου σα από την ΙΜΚΟ και από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, γιατί τη δουλειά που έκαναν. Χαιρετίζουμε αυτή την γρήγορη κατάληξη τούτου του θέματος και ελπίζουμε πως αύριο θα εγκριθεί. Εμείς συμφωνούμε, οι καταναλωτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορούν να επιβάλλουν τα δικαιώματά τους σε τέτοιου είδους υποθέσεις και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αυτή την οδηγία. Μέσω λοιπόν αυτών των αντιπροσωπευτικών αγωγών υπέρ των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών θα έχουμε νομιμοποιημένες νομιμοποιημένες φορείς, για παράδειγμα ενός καταναλωτών, ανεξάρτητες αρχές, ανεξάρτητους φορούς, να μπορούν να αναλάβουν δράση, να παρέμβουν όταν έχουμε καταπάτηση του καταναλωτικού δικαίου και να βοηθούν έτσι ώστε να ε, λάβουν αποζημίωση όσοι ε, υπέσαν βλάβη. Θα βοηθήσει αυτό του ευαίσθητου καταναλωτέ σε περιπτώσει όπου δεν έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τα δικαιώματά του μεμονωμένα. Η πρόταση ανταποκρίνεται στην ανάγκη για την υποχρεωτική ε, εκτέλεση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, λαμβάνοντα υπόψη την αναλογικότητα και την επικουρικότητα. Δίνει λοιπόν στα κράτη-μέλη περιθώριο ελιγμών για ε, βασικά ε, διαδικαστικά θέματα. Θέλουμε να βρεθούν λύσεις οι οποίες εξασφαλίζουν τα δικαιώματα του καταναλωτή και εξασφαλίζουν πως οι εμπορευόμενοι επίσης την χάνουν δίκαιες αντιμετώπισης και από την αρχή ξεκαθαρίσαμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να δημιουργήσει εδώ μία ε, κουλτούρα αγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον τρόπο αυτό δεν ανοίγουμε ε, αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει έτσι. Όχι, η συλλογική αποζημίωση στην Ευρώπη είναι δίκαιη για τον καταναλωτή και για τις επιχειρήσεις και δεν έχει τιμωρητικές ε, κυρώσεις ούτε ε, φέρνει αυτές τις αγωγές καθομοδικίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο που διεξάγονται στις Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό προκρίνει τις συλλογικότητες που θέλουν να στηρίξουν τα δικαιώματα του καταναλωτή στην Ευρώπη. Χαίρομαι που στηρίζετε κι εσείς αυτές τις αρχές και ξέρω πως ε, οι νομιμοποιούμενοι φορείς είναι μια έννοια που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, όπως επίσης και το γεγονός πως τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν τους διαδικαστικούς κανόνες, έτσι ώστε να υπάρχουν ξεκάθαροι και ισχυροί κανόνες για ένα αναλογικό και αντιπροσωπευτικό σύστημα αποζημιώσεων που ταιριάζει στο ευρωπαϊκό μοντέλο. Και με αυτό και με αυτή την καινοτομία πιστεύω πως αυτή η πρωτοβουλία στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον Ευρωπαίο καταναλωτή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση του νοιάζεται. Και πιστεύω πως ο τρόπος με τον οποίο θα ε, ψηφίσετε αύριο, που είμαστε και σε προεκλογική περίοδος, είναι πολύ σημαντικός. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ούτε τον κύριο Μάγερ βλέπω. Και επομένως ε, θα περάσουμε ε, στις, ε, στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ο κύριο Σβόποντα για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κυρία Επιτροπέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον κύριο Διτιέ, για τη δουλειά που έχει κάνει για το κείμενο αυτό. Και να ευχαριστήσω και εσά κυρία Επιτροπέ, γιατί οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένουν ένα κάποιο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και θεωρώ ότι αυτό το κείμενο αποτελεί μια καλή σύμβολη στην, στο επίπεδο αυτό προστασίας. Ε, περιλαμβάνει μια σειρά σημείων. σε ό,τι αφορά τι συλλογικέ ε, προσφυγέ ε, σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις για αυτές. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε όλα αυτά να γίνονται όταν πρόκειται για προστασία των καταναλωτών πραγματικά και όχι για κατάχρηση για να βγάζει κανείς χρήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Τελβό για 1,5 λεπτό από τους σοσιαλδημοκρατές. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Παρά το έντονο λόμπινγκ που αντιμετωπίσαμε και την ε, χάρη στην αντίσταση της αριστεράς και χάρη και στον κύριο Διδιέ καταφέραμε να πετύχουμε μια, ένα καλό συμβιβασμό. 29, 19 κρατημέλη σήμερα έχουν τέτοιους μηχανισμούς συλλογικών ε, προσφυγών. Αυτή η νέα πρόταση οδηγίας θα εξασφαλίσει ελάχιστα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των ε, καταναλωτών που θα μπορούν πλέον να ασκήσουν αλληλέγγυες δράσεις για να προασπίσουν τα συμφέροντά τους. Και θα θέλαμε λοιπόν να διευκολύνουμε, να διευκολύνουμε τη δημιουργία ενώσεων ε, εκπροσώπησης ε, των ε, καταναλωτών για να υπάρχει διαφάνεια να αποφύγουμε σύγκρουση συμφερόντων και να επιταχύνουμε την όλη διαδικασία τελικά για την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή. Δύο πράγματα με λοιπόν. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, γιατί οι καταναλωτές, οι πολίτες μάλλον δεν είναι μόνο καταναλωτές. Έχουμε θέματα γενομικά, έχουμε ε, παράγοντε περιβαλλοντικού σε ό,τι αφορά και τις ε, επιχειρήσει. Σε περιπτώσεις λοιπόν αυτές θα πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες για τις λογικές ε, πρόσφυγες. Κατά δεύτερον, δεν καταφέραμε να βρούμε μια κοινή θέση και έτσι λοιπόν αυτή τη δεν θα υπάρχει ένας μηχανισμός τέτοιος που θα είναι πολύ σημαντικός για τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτόν τον εύθυμο χαρακτήρα, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Πακέ ούτε αυτός στην αίθουσα, άρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Φαμίλτενμπουρχ. Από τους φιλελεύθερους, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η σταθερή άμα εσωτερική αγορά αποτελεί προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη των πολιτών. Έχουμε τα θέματα του Dieselgate, τα θέματα της Facebook που μειώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα σε ό,τι αφορά λοιπόν τις συλλογικέ συμβάσεις. Είναι σημαντικό στοιχείο αυτό και με την νομοθεσία που ψηφίζουμε αύριο θα δημιουργήσουμε σημαντικές προϋποθέσεις για τους πολίτες προκειμένου να αναλαμβάνουν δράση από κοινού και να ζητούν αποσημειώσει για να προστατεύσουμε λοιπόν τον καταναλωτή και να υπάρχει καλύτερη ισορροπία μεταξύ καταναλωτή και παραγωγού. Αύριο λοιπόν ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνουμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα είναι πλέον το μπαλάκι στην πλευρά στο γήπεδο του Συμβουλίου και να ξεκινήσει τι διαπραγματεύσει μετά τι εκλογέ με το νέο Κοινοβούλιο προκειμένου να βρίσκουν το δίκαιο, το δίκαιο τους σε όλη την Ευρώπη οι καταναλωτέ. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ κύριε Λεμπρετών. Εξ ονόματος του ΕΝΕΦ, ένα λεπτό κύριε Λεμπρετών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια Ευρώπη τη business μονάχα ε, στην ε, ε, υπηρεσία των, του μεγάλου κεφαλαίου και των τραπεζών. Το σχέδιο εδώ, το οποίο μας έχει υποβληθεί, δίνει την δυνατότητα για αντιπροσωπευτικές αγωγές, αυτό που οι Αμερικάνοι ονομάζουν clash actions. Ε, σημαίνει ότι ορισμένοι καταναλωτές οι οποίοι έχουν υποστεί παρόμοια ζημία να έχουν τη δυνατότητα κοινή αντιπροσωπευτική αγωγή ενώπιον των δικαστηρίων. Έπρεπε οπωσδήποτε να δημιουργηθεί αυτή η δυνατότητα γιατί λίγες είναι οι χώρες μεταξύ των οποίων έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ε, με τον τρόπο αυτό και μέχρι την υπάρχουσα κατάσταση ε, μονάχα οι Αμερικανοί πολίτες είναι προστατευμένοι ε, σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Όπως ας πούμε στα πλαίσια του Dieselgate 22 ευρώ έχουν ε, δοθεί στους ε, ζημιωμένους Αμερικανούς ενώ τίποτα στους Ευρωπαίους. Εδώ αναφέρεται ότι οι αντιπροσωπευτικές αγωγές μπορούν να γίνουν από νομιμοποιημένους φορείς οι οποίοι δεν θα έχουν σκοπό το κέρδος και ότι θα υπάρχει η δυνατότητα πλήρους αποζημιώσεως της οποιασδήποτε βλάβης. Επίσης ε, θα πρέπει και αναφέρεται αυτό να γίνονται ε, σεβαστές ε, οι αρχές αντιπροσωπευτικών αγωγών που υφίστανται και ισχύουν ήδη σε ορισμένες χώρες όπως στην Γαλλία. Ευελπιστούμε πάντως ότι η κατάσταση όσον αφορά τις αντιπροσωπευτικές αγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πιο εύκολες από ότι οι πολύ γραφειοκρατικές γαλλικές. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρουζιάρ δεν είναι εδώ. Η κυρία ναι, ναι. Σαλντεμόζε, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή ε, η πρόταση οδηγίας ε, γιατί ξέρουμε ότι ακόμα και σε χώρες οι οποίες έχουν την, τους μηχανισμούς αυτούς είναι πάρα πολύ δύσκολο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και επομένως επίγει η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Βεβαίως εδώ μιλάμε για πολύ θετικά στοιχεία, για αντιπροσωπευτικές κοινέ αγωγές, μιλάμε για την δυνατότητα να ε, αντιμετωπίσουν μια συγκεκριμένη επιχείρηση από κοινού ε, κάποιοι ζημιωμένοι ε, πολίτες. Είδατε τι έγινε με το Dieselgate είδαμε ότι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ε, πολύ χειρότερη από ό,τι στις Ηνωμένε Πολιτείε. και επομένως πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει τους ε, πολίτες. Αυτό το χρειαζόμαστε έτσι ώστε να βελτιώσουμε την εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Πάκετ, ε, σας βλέπω μεταξύ μας. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Κατ' εξαίρεση σας τον δίνω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. το Dieselgate μας έτριψε τα περιστατικά αυτά στη Μούρη, γιατί ε, είδαμε τι προβλήματα υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τελικά αυτός που έπεσε θύμα ε, της όλης υπόθεσης ήταν ο καταναλωτής, ε, τον οποίο καταλήψαμε στη μοίρα του. Γιατί στην τελική ανάλυση ποιος καταναλωτής ε, θα αντισταθεί με, στις μεγάλες επιχειρήσεις μέσω ε, δύσκολων και δυσνόητων νομικών διαδικασιών. Δαβίδ δηλαδή εναντίον Γολιάθ. Αυτό που είναι σαφέ είναι ότι θα πρέπει οι καταναλωτέ να αποζημιώνονται για την ζημία την οποία υπέστησαν. Για να κάνουν τον αγώνα αυτό και για να αντιτηρήσουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών θα πρέπει οι καταναλωτές θα να έχουν την, τις ε, αρμοδιότητες που χρειάζονται για να μπορούν να αντισταθούν σε όλα αυτά. Και στη Φλάνδρα έχουμε τέτοιους μηχανισμούς. Ελπίζω σύντομα να έχουν τέτοιους μηχανισμούς και όλοι οι καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γκέμπαρτ, Για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπό Γιούροβα γιατί επιτέλους δρομολόγησε ένα στοιχείο το οποίο το Κοινοβούλιο το ζητάει πάρα πολύ καιρό και το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αγνοούσε επί σειρά ετών. Ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα την Επιτροπή Γιουροβά. Θα ήθελα λοιπόν να μπορούσα να βγω να πω στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι επιτέλους έχουν πλέον μία λύση για να βρουν το δίκαιο τους με συλλογικές συμβάσεις. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς καλές είναι οι εργασίες μας, καλές είναι οι προτάσεις μας, καλή είναι και αυτή η έκθεση στην τελική ανάλυση αν και θα μπορούσε να βελτιωθεί, μάλλον βελτιώθηκε πάρα πολύ από, τους, ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώ όμω δεν το κάνουμε που δεν παίζει και το Συμβούλιο. Αποφάσισε ποια ήταν η βάση λοιπόν για τις συμπραγματεύσει με το Κοινοβούλιο και αυτό είναι λυπηρό γιατί αυτό θεωρώ ότι αφαιρεί πολλά δικαιώματα από τους Ευρωπαίους πολίτες και διαιωνίζει μια κατάσταση. Μα εμποδίζει να κάνουμε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε τελικά στου πολιτέ. Αυτό πραγματικά θέλουμε να το πετύχουμε. Θέλουμε να βρουν το δίκαιο του. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε και στη νέα θητεία να το απαιτούμε αυτό, να εργαζόμαστε προ την κατεύθυνση αυτή, προκειμένου αυτά τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών να τα εγγυόμαστε πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο. Δεν βλέπω να ζητά κανεί. το λόγο στο Catch the Eye. Το λόγο έχει η κυρία Γιούροβα. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα είπατε. Και πραγματικά ε, το Dieselgate είναι ναι, μία από τις ε, αιτίες για τις οποίες δώσαμε αυτή την όθηση σε αυτή την πρόταση, γιατί μπορέσαμε να εξηγήσουμε πως χρειαζόμαστε τη δυνατότητα οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να ε, μπορούν ε, συλλογικά να περασπίσουν τα δικαιώματά τους. Και μπορώ να σας πω πως σε κάθε κράτος μέλος υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις με ε, τέτοιου είδους παραβιάσεις. Έχουμε στην Ισπανία το πρόβλημα με τα ενυπόθηκα δάνεια που καλύπτει 6.000 άτομα. Δεν είναι μόνο το Dieselgate λοιπόν, ίσως είναι η πιο γνωστή υπόθεση, αλλά υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος αρκετές. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και, την... και τους εισηγητές. Πιστεύω πως η έκθεση αυτή της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων θα στηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο να σας πω πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πείσουμε τα κράτη-μέλη μετά τις εκλογές πως αυτό είναι το απαραίτητο βήμα προς τα εμπρός για να προστατεύσουμε καλύτερα τους ε, Ευρωπαίους καταναλωτές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντιντιέ, θέλετε να κλείσετε εσείς αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Επίτροπος Γιούροβα είπε δύο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πρώτον, ότι ο στόχος δεν είναι να τιμωρήσουμε οποιονδήποτε, αλλά ε, αποκλειστικό στόχος είναι η αποζημίωση ε, των ε, θυμάτων και η διόρθωση οποιοδήποτε σφάλματος. Και δεύτερον, να μην, δεύτερο σημείο, να μην είμαστε ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος με τα class action της Αμερικής. Ακούσαμε και τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ το ΕΛΚ ε, για την πλήρη υποστήριξη, το Ζιλ Μπρετόν για το θετικό πνεύμα, καθώς επίσης και τη Ζαν Φοντερβό, η οποία με εντυπωσίασε με την ε, ε, ικανότητα διαλόγου και την προσπάθειά της εξέβρεσης συμβιβαστικής ε, ε, λύσης καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να σας πω ότι αν επανεκλεγούμε, οπωσδήποτε θα συνεχίσουμε ε, και θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την εργασία αυτή στα πλαίσια του ημερούς διαλόγου. Εν πάση περιπτώσει πάντως να μην λησμονείτε ότι εγώ δεν θα υποχωρήσω ούτε μία σπιθαμή. Βασιστείτε πάνω μου, βασιστείτε πάνω μας για την προστασία των ε, καταναλωτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Διδιά. Αύριο θα λάβει χώρα η ψηφοφορία. Ε, περιμένουμε να καθίσει και ο Επίτροπος Αρίας Κανιέτη, τον οποίο αναμένουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να ξεκινήσουμε και το επόμενο θέμα. Euh, Πολύ ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε. Έχουμε εδώ τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα του Dieselgate και έχουμε τον κύριο Αρία Σκανιέτη. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, 3,5 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ξέσπασε το Dieselgate και έκτοτε μάθαμε πως οι κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραβίασαν τους κανόνες για τη ρήπανση. Αυτό ήταν εξαιρετικά βλαβερό και για την υγεία των Ευρωπαίων πολιτιών και γιατί χάθηκε η εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τον κλάδο και γιατί επηρέασε ε, την εμπιστοσύνη στο ε, ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οχήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να ξεπεραστεί το σκάνδαλο αυτό, να ε, αποδοθούν ευθύνε και να μην επαναληφθεί. Πολλά πετύχαμε. Το Μάιο του 2018 στήσαμε ένα πιο αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο που εξασφαλίζει μεγαλύτερη ανεξαρτησία και διαφάνεια στην έγκριση τύπου. Οπότε αυτό θα βελτιώσει πολύ την κατάσταση θα έχουμε πολύ πιο συγκεκριμένες δοκιμές για τις εκπομπές ερπογόνων ουσιών με διαδικασίες οι οποίες θα είναι πιο αντιπροσωπευτικές για τις εκπομπές ε, κατά τη διάρκεια της κίνησης στο δρόμο. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή τα ντίζελ εκπέμουν 40 μιλιγράμμ νόξ το χιλιόμετρο και ήταν στο παρελθόν 700 με 800 ε, μιλιγκράμμ ε, όταν ε, οδηγούσαν σε πραγματικές συνθήκες. Άρα το ρυθμιστικό μας πλαίσιο είναι από τα πιο αυστηρά στο στον κόσμο και έχουμε βρει ένα πιο σύγχρονο και ρεαλιστικό τρόπο να μετράμε αυτές τις εκπομπές με το πλαίσιο δοκιμασιών που δοκιμών που έχουμε για τα ελαφρά οχήματα. Και ξέρετε πως αυτό είναι καλύτερο και για τον καταναλωτή που ε, ενημερώνεται καλύτερα με τις νέες αυτές δυνατότητες δοκιμών που έχουμε εγκρίνει. Επίσης, έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβάση εναντίον κράτων μελών για ε, θέματα έγκρισης τύπου. Και από αυτές τις ε, υποθέσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία και έχουν οδηγήσει σε αλλαγές σε κάποιες περιπτώσεις στην νομοθεσία των κρατών μελών από το Νοέμβριο του 2017 ε, και μετά για την ανάκληση των οχημάτων φτιάξαμε μια πλατφόρμα ε, και αυτό με την ευκαιρία των ιδεών που μας έδωσε το σκάνδαλο Dieselgate. Και να σας πω πως μέχρι σήμερα ε, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη νομική αρμοδιότητα να επιβάλλουμε ανακλήσεις. Εξακολουθεί να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών που είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν τους ε, κατασκευαστές και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την ε, διαδικασία. Αλλά από το Σεπτέμβριο του 2020 η νέα οδηγία θα επιτρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις και πρόστιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ευρωπαϊκές δοκιμές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ε, εξαντλητικές πληροφορίες για το τι γίνεται με τις ανακλήσεις και πώς έχουν επηρεάσει τα οχήματα αυτά το ευρωπαϊκό περιβάλλον και τον αέρα που εισπνέουμε. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να επιβάλλουμε τους νέους κανόνες που έχει δημιουργήσει η Κομισιόν και τις οποίες έχουν, εναντίον των οποίων έχουν προσφύγει ε, στο Γενικό Δικαστήριο. Βέβαια, Έχουμε αυτή τη στιγμή τους κανόνες συμμόρφωσης που χρησιμοποιούμε και αυτοί οι παράγοντες συμμόρφωσης ε, είναι υποχρεωτική για να δούμε ε, στατιστικά τι γίνεται με αυτές τις νέες δοκιμές και επίσης ο κινητός εξοπλισμός μέτρησης ε, τι περιθώρια σφαλμάτων επιτρέπει και πόσο αποτελεσματικός είναι. Ήθελα να σας ενημερώσω πως εμείς έχουμε προσφύγει κατά της απόφασης δεν έχουμε ξεπεράσει τι αρμοδιότητέ μα. Έχουν προσφύγει και η Γερμανία και η Ουγγαρία και δεν έχουμε ε, ξεπεράσει ε, τα όρια ε, της εντολής μας. Βεβαίως δεν γνωρίζω αυτή η προσφυγή τι τροπή θα λάβει. Ξέρω πως ετοιμάζουμε μία πρόταση η οποία πρόκειται να εγκριθεί τον Απρίλιο. Θα προτείνουμε στους συνομοθέτες να εγκρίνουν τους ε, παράγοντες συμμόρφωσης και το δεύτερο παράγοντα να τον μειώσουμε εφόσον το εξασφαλίζει η τεχνολογική πρόοδος. Το κάναμε άλλωστε ήδη μία φορά και θα πρέπει μαζί με τις δοκιμές να επιβάλλουμε και τους ε, ε, παράγοντες αυτούς, ε, κάτι το οποίο είναι θετικό για όλους. Σύμφωνα με τα όσα είπε και η έκθεση του ελεγκτικού Συνεδρίου για την απόκριση στο σκάνδαλο Dieselgate, πρέπει να σας πω πως έδωσε αφετηρία και όθηση σε πολλές νομοθετικές προτάσεις και το ελεγκτικό συνέδριο υπογραμμίζει πως μπορούν να γίνουν περισσότερα αλλά θα χρειαστεί χρόνος μέχρι αυτές οι νομοθετικές αλλαγές να επηρεάσουν ε, τον αέρα που εισπνέουμε. Εμείς έχουμε ε, ετοιμάσει έναν οδικό χάρτη προς τα πιο καθαρά οχήματα έτσι ώστε να μην ξαναπεράσουμε αντίστοιχη κατάσταση στο μέλλον. Και παρουσιάσαμε τον οδικό χάρτη στις 18 Μαρτίου ε, στο φόρουμ στο Κράιοβα με συγχωρείτε, στην έκθεση αυτοκινήτων στο στην Κράιοβα. Και στόχος μας είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε και το ίδιο να μένουμε και από τα κράτη-μέλη και από την αυτοκινητοβιομηχανία μας. Και ας δούμε το μέλλον μας πιο θετικά. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια. Έχουμε στόχο για τη μείωση για το ε, διοξείδιο του άνθρακα. Το ίδιο θα κάνουμε και για τις ε, απόλυτες ανθρώπινες ζωής και θα πρέπει επίσης να δούμε ε, τι θα γίνει και με τα οχήματα στο μέλλον. Θα ξεκινήσει η συζήτηση με τους σοσιαλιστές. Ε, η συνάδελφος έχει το λόγο για δύο λεπτά. Κυρία Νταλόν. Λυπάμαι που δεν είναι εδώ η κυρία Μπλικοφκά. Ε, για να μας μιλήσει εδώ για, τον ε, περίφημο, ε, για την περίφημο παράμετρο συμμόρφωσης. Βέβαια, είμαστε ικανοποιημένοι στις γενικές γραμμές που έχει και τα μέτρα που έχει λάβει η Κομισιόν. Βέβαια, αυτός, ο, αυτή η παράμετρο συμμόρφωσης είναι πολύ ελαστικός και δυστυχώς ακυρώθηκε από το δικαστήριο δικαστήριο. Εάν ε, ε, είχε ανακύρωσε λοιπόν ε, αυτή την εκτελεστική πράξη ε, το δικαστήριο είναι γιατί αντιτίθεται εις τον τύπο Euro 6 που αναφέρεται στα NOx και πρέπει να πω ότι η ίδια η Επιτροπή μπροστά από τις, τους βουλευτές ενώπιον των βουλευτών της ειδική Επιτροπής ΕΜΙΣΕ είχε λάβει συγκεκριμένες Προ ε, προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι ε, ε, πραγματικά εκπληκτικό πώς μπορούν να δίνονται τέτοιες διασφαλίσεις και μάλιστα για μέσα οι οποίες πόρο απέχουν από αυτές τις οποίες εμείς θα μπορούσαμε να προτείνουμε και οι οποίες θα κάλυπταν τις ανάγκες της υγείας των πολιτών πάντα σύμφωνα και με την τάξη Euro 6 η Κομισιόν έχει κερδίσει χρόνο σε αυτήν τη διαδικασία αντιπαράθεσης με το, με το δικαστήριο, αλλά δυστυχώς εμείς σαν πολίτες δεν έχουμε πια χρόνο. Κάθε εβδομάδα Χιλιάδες πολιτών κατεβαίνουν στους δρόμους έτσι ώστε να καταδείξουν το επίγον της καταστάσεως. Ε, στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις πνίγονται από τα διοξίδια του αζότου ε, και από τις εκπομπές αυτές ε, οι κάτοικοι. Επίσης, στο Παρίσι να σας πω ότι ήδη έχουμε ξεπεράσει 19 μέρες έναντι των τριών που υποτίθεται ότι ήταν το όριο, έχουμε ξεπεράσει λέω το όριο των ε, ε, μικρών σωματιδίων ε, θα πρέπει και τα κράτη και η Κομισιόν να πάρουν σύντομα τα μέτρα τους. Ευχαριστώ, ο κύριος Ντεμεσμέκερ. Ένα δεύτερο σκάνδαλο Dieselgate. Αυτό θέλαμε να αποτρέψουμε με την σχετική επιτροπή, με τη σχετική ερευνητική επιτροπή Παρακολουθούμε λοιπόν το ζήτημα αυτό και πρέπει να ομολογήσω ότι μπήκε και η άναξη, Παρόλο που μπήκε η άνοιξη όμως δεν έχουμε ακόμα δει τα, τη νέα σοδιά. Ε, με επίτροπος, η, η Επίτροπος Μιαγνώσκα είπε ότι το Dieselgate ουσιαστικά δεν έχει ολοκληρωθεί και η έκθεση του Ερεκτικού συνεδρίου δεν είναι καθησυχαστική. Θα μπορούσε να προκύψει ένα δεύτερο Dieselgate. Θα πρέπει όμως να διδαχθούμε από τα παθήματα ε, του παρελθόντος. Τι γίνεται λοιπόν με την ε, μείωση των προτύπων σε ό,τι αφορά το άζωτο. Έγιναν διάφορα τεστ στον δρόμο και συνδέθηκε αυτό με μείωση των προτύπων. Εμείς ψηφίσαμε κατά τότε γιατί έχουμε τη τεχνολογία που χρειάζεται για να πετύχουμε τα επίπεδα αζότου τα οποία χρειάζεται χωρίς να υπάρχει αρνητικός αντικτύπος σε ό,τι αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Το ρετικό συνέδριο το μάλλον το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι αυτή η μείωση του, των προτύπων για το άζωτο είναι παράνομη. Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγγέλει αυτό το προσφεύγει κατά τις απόφασεις του, του δικαστηρίου. Ο κ. Γερμπράντη έχει τώρα το λόγο, λέει η Πρόεδρο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και έχουμε δύο σημεία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω σήμερα το βράδυ. Καταρχά, ότι το Κοινοβούλιο ποτέ δεν έλαβε πραγματική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, Επιτροπή, την Ερευνητική Επιτροπή. Λάβουμε μία απάντηση της ε, Επιτρόπου Πιανκόφισκα, όχι όμως για τις συμπεράσματα, αλλά για τις συστάσεις. Κάποια στοιχεία μόνο. Αυτό μας είπε ότι ήταν... Ε, κάποια στοιχεία μάλλον στην αποκλειστική αρμοδιότητα γνώση ε, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν μπορούσε να τα απαντήσει. Να δώσει απαντήσει στην Επιτροπή μας. Αυτό θεωρώ ότι είναι θέμα Ευρω... νομιμότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλω πριν το τέλο τη θητεία να δοθούν σωστέ και κατάλληλε απαντήσει και στα συμπεράσματα και στι συστάσει μα Δεύτερο σημείο που θα ήθελα να δείξω. Ποτέ ουσιαστικά δεν διορθώσαμε τα σπασμένα του Dieselgate. Προέκυψε νέα νομοθεσία, αυτό ναι. Αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν όλα αυτά τα κίνητα τα κυκλοφορούν στι ευρωπαϊκέ πόλει. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν. Μία ισχυρή δυναμική, συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση. Πλέον το έχουμε αφήσει στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη λοιπόν λαμβάνουν μέτρα, αλλά με τέτοιο τρόπο που ενδεχομένως να γλιτώσουμε τα αυτοκίνητα αυτά στην κάθε χώρα, αλλά ουσιαστικά τι γίνεται, εξαγάγονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν υπάρχει λοιπόν σοβαρή αντιμετώπιση και δεν λαμβάνει σοβαρά ο αντίκτυπο στην υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Ο μοναδικό λοιπόν φορέας που μπορεί να κάνει μια τέτοια ευρωπαϊκή δράση συντονισμού είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα παρακαλώ λοιπόν Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα πάρετε στα σοβαρά όλα αυτά και να διοργανώσετε μια τεράστια δράση και άσκηση με τα κρατημέλη για να βγουν από τους δρόμους μας τα αυτοκίνητα αυτά. Να φροντίσουμε να συμβαδίζουν με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και σε ό,τι αφορά το λογισμικό και το υλικό τους να υπάρχει σχετική αναβάθμιση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Eichhout από τους Πράσινους για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Και όντως θα εκφράσω και εγώ τη δυσαρέσκειά μου όπως και οι υπόλοιποι βουλευτές. Φυσικά έγιναν βελτιώσεις και έχουμε εργαστεί σκληρά για αυτές. Ωστόσο, πολλά θέματα ακόμα δεν έχουν λυθεί. Αυτό που είπε ο συνάδελφος Γερμπραντή. Εξακολουθούν να υπάρχουν τέτοια αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν και μολύνουν την ατμόσφαιρα. Είναι αυτοκίνητα Dieselgate. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν, δεν παίρνει καν δράσει, δεν παίρνει καν πρωτοβουλία για να διορθώσουν την κατάσταση. Δεν Είναι σχετικό αυτό. Μία ερώτηση λοιπόν να κάνω. Ξέρουμε ότι έχουμε διάφορε περιπτώσει παραβίαση και η Επίτροπο Μπιακόφσκα έλεγε και διαρκώς υποσχόταν ότι θα ξεκινήσουν και άλλες διαδικασίες επί παραβάσεις. Ήταν αυτό για να μας καθησυχάσει. Δεν μας έλεγε την αλήθεια ή πραγματικά δρομολογούνται και άλλες διαδικασίες επί παραβάση. Πού βρισκόμαστε με τις υπόλοιπες περιπτώσεις λοιπόν. Τελευταίο θέμα. Έχουμε διάφορες περιπτώσεις ε, στον διαμεσολαβητή. Και θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και στις τεχνικές ομάδες εργασίας. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δίνει τα πρακτικά των τεχνικών συναντήσεων. Χρειαζόμαστε τα στοιχεία αυτά. Ιδάλλως έχουμε την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προστατεύει τα κρατημέλη που προστατεύουν τα βρώμικα και τα απλητά τους, αν θέλετε. Η κυρία Κιλώνα έχει τώρα το λόγο, λέει η Πρόεδρος. Arvoisa rouva Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι πως το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε τον καθρέφτη και να δούμε τι κάναμε για τα καταναλωτη... δικαιώματα του καταναλωτή. Αυτό είναι το βασικότερο βήμα. Να σας πω ότι έχω συζητήσει με πάρα πολύ κόσμο και όλοι κάνουν την ίδια πολύ καλή ερώτηση. Τι μπορούν να κάνουν για να δώσουν τη μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος για να μειώσουν τι εκπομπέ κτλ. Και κυρίως αυτοί που έχουν οχήματα diesel. με ρωτάνε ποια είναι τα νομικά εχέγγυα που τους εξασφαλίζουν όταν καλή την πίστη αγόρασαν τα οχήματα αυτά και όταν μιλάμε κυρίως για τι πραγματικές εκπομπές. Άρα λοιπόν αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την νομοθεσία μα και με το ποιε είναι οι δράσει μα και το αν είναι υπαρκή, αλλά και το γεγονό πω ο καταναλωτή πώς μπορεί να εμπιστεύεται τα προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται και τα οποία εμείς εγκρίνουμε μέσω της νομοθεσίας που εγκρίνουμε. Πιστεύω λοιπόν πως θα πρέπει να το συζητήσουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να συζητήσουμε το μέλλον των οχημάτων με κινητήρα diesel. Πώς μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε, πώς μπορούμε να τα ε, βελτιώσουμε και τι θα γίνει με το βιο-δίζελ. Γιατί όλα αυτά τα ερωτήματα χρειάζονται να απαντηθούν. Όχι μόνο το τι θα γίνει μετά το gate. Δεν νομίζω λοιπόν ότι δίνουμε απαντήσεις και πιστεύω πως πολλά θα πρέπει να βελτιώσουμε έτσι ώστε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. Η κυρία Εύη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ και δύο χρόνια προσπάθησε η Διερευνητική Επιτροπή, να, επιτροπή μας να ξεκαθαρίσει τα όσα συνέβησαν με το Dieselgate, αλλά δυστυχώς ε, η κατάσταση δεν ήταν καθόλου ξεκαθαρισμένη, ε, όπως άλλωστε δεν ήταν ξεκάθαρη και η θέση της Κομισιόν και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Τώρα έχουμε ε, το σύστημα της συμμόρφωσης των οχημάτων με ένα σύστημα επαγρύπνησης και επιτήρησης ε, πιο ε, αυστηρό, ε, το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να αποφύγουμε στο μέλλον τέτοιου είδους εγχειρηματοποίησης των δοκιμών. Αλλά όλα αυτά πραγματικά είναι μια τεράστια κατραπακιά σε όλα αυτά τα οποία έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έπρεπε να έχουν υπάρξει ανακλήσει σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα έπρεπε να έχουν τιμωρηθεί οι αυτοκινητοβιομηχανίες οι οποίες έχουν μολύνει ε, το περιβάλλον, τον αέρα που αναπνέουν οι πολίτες και οι καταναλωτές. Άρα δεν είναι δυνατόν να πέσουν οι τίτλοι τέλους για αυτήν την κατάσταση. Έχουμε ευθύνη απέναντι στους πολίτες που όπως και εμείς και εκείνοι περιμένουν ε, την τελική, το τελικό συμπέρασμα, ε, την τελική σελίδα των εργασιών που έγιναν και στα πλαίσια της ΕΜΗΣ αλλά και παντού. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά η κυρία Σαλντεμόζε. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, εγώ Αισθάνομαι και εγώ λίγο όπως οι προηγούμενοι συνάδελφοι που είπαν ότι δεν καταλαβαίνουν όλους αυτούς τους επένους της ε, Κομισιόν σε σχέση με τα όσα έκανε η ίδια. Πώς είναι δυνατόν κανείς να είναι τόσο ευχαριστημένος βεβαίως. Υπάρχουν κάποιοι νέοι κανόνες που θα αρχίσουν να ισχύουν από το 2020. Ωστόσο υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι πάρα πολλά τα εκατομμύρια των ε, αυτοκινήτων που μολύνουν ε, ε, το περιβάλλον και που κινούνται στους δρόμους μας δεν είναι δυνατόν να ε, μην έχουμε ε, μία πλήρη ανάκληση των αυτοκινήτων που ε, παρουσιάζουν πρόβλημα με σκοπό τον εξυγχρονισμό τους. Έχει γίνει σε ορισμένες χώρες αυτό. Θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα αυτοκίνητα τα οποία μολύνουν, ποια είναι τα αυτοκίνητα τα οποία σκοτώνουν τον κόσμο. Αυτό θα πρέπει να το πει και η Κομισιόν και να καταλάβει ποιος είναι ο προβληματισμός μας. Πρέπει να βρεθεί κάποια λύση στο μέλλον θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ανάκληση όλων των αυτοκινήτων τα οποία έχουν παρουσιάσει προβλήματα. Και ε, οπωσδήποτε θα πρέπει ανεξάρτητοι οργανισμοί ε, να ε, ε, κάνουν δοκιμές, τεχνικές δοκιμές με απολύτως διάφανο τρόπο έτσι ώστε να ξέρουμε, να μπορούμε να ελέγξουμε κατά πόσον οι κανόνες γίνονται σεβαστοί θα πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι ούτε για το κλίμα, ούτε για το περιβάλλον, ούτε για την υγεία ε, τα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προκαλούν πρόβλημα ή ζημία. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για τα οχήματα τα οποία εξάγονται στην Ανατολική Ευρώπη γιατί διαφορετικά απλώς πεδαριοδός προσπαθούμε να μετακινήσουμε και να μετακυλήσουμε το πρόβλημα. Η Κομισιόν θα πρέπει όλα αυτά να τα λάβει υπόψη της. Ο κύριος Λοτόφσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το Dieselgate ήταν ένα πραγματικό ε, σκάνδαλο ε, και η συνεργασία με τις αυτοκινητοβιομηχανίες ε, δεν έλαβαν υπόψη όλους τους προβληματισμούς. Στην ουσία είναι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που προσπαθούν να βρουν το δίκαιο τους ακόμα και ενώπιον των δικαστηρίων. Αυτό το Dieselgate είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σοβαρό ε, αλλά βεβαίως δεν μπορεί να συρρυκνωθεί μονάχα ε, στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στριμωγμένοι με την πλάτη στον τοίχο ε, και που προσπαθούν να βρουν λύση στο πρόβλημά τους. Ο αγώνας, ας πούμε, για καθαρό περιβάλλον και καθαρό αέρα δεν είναι δυνατόν να περιορίζεται σε ένα τέτοιου είδους αγώνα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντελή. Αγαπητοί περίπου τέσσερα χρόνια μετράμε από την στιγμή ε, του Dieselgate. 30 εκατομμύρια ήταν τα οχήματα τα οποία μόλυναν πολύ περισσότερο από όσοι έπρεπε. Δημιουργήθηκε μάλιστα και μία ε, ειδική επιτροπή. Έκανε συστάσεις. Όλα αυτά χωρίς ε, καμία συνέχιση αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, αφήνουμε τους, ε, τα οχήματα αυτά να μολύνουν, αφήνουμε ε, αυτούς τους αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στους δρόμους. Εντάξει, μωρέ, δεν έγινε και τίποτα, ε, αλλά πραγματικά κάτι πρέπει να αλλάξει. Αυτό που ζητούμε είναι να καταλάβουμε τα διδάγματα του Dieselgate, να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να προστατέψουμε τους καταναλωτές και όχι αποκλειστικά τους αυτοκινητοβιομηχάνους. Εσείς με ποια πλευρά ε, ε, τίθεστε, με ποιους συστοιχίζεστε, επιτέλους να σταματήσουν τα λόγια και να αρχίσουν οι πράξεις. Πρόεδρος, δεν έχω έτοιμα αγόρευση στα πλαίσια του Catch the Eye και επομένως κύριε Επίτροπε σας δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την ε, συζήτηση. Είναι πολύ σχετικά όλα τα σχόλια και οι ερωτήσεις. Αρκετοί μιλήσατε για τη διαδικασία επί παραβάση για follow-up για το Dieselgate. Το 2016 ξεκινήσαμε με έξι ε, τέτοιες. Γερμανία, Ισπανία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ελλάδα, ε, Τσεχία και Ιταλία. Γιατί δεν εφάρμοσαν στην νομοθεσία τους είτε ε, το σύστημα κυρώσεων ε, ε, για την αυτοκινητοβιομηχανία είτε δεν παρακολούθησαν σωστά. Επίσης, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο, Ισπανία και Γερμανία ειδοποιήθηκαν πως συνεχίζει η διαδικασία και το ίδιο συνέβη και με την Ιταλία για κάποιο συγκεκριμένο κινητήρα δίζελ. δεν ήταν πλήρες οι απαντήσεις τους και έχουν ξεκινήσει και νέες διαδικασίες τις οποίες θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε. Κάποιοι από εσάς αναφερθήκατε και στις ανακλήσεις. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι στην κοινή πλατφόρμα που έχουμε με την απόφαση του 2018 και τα περισσότερα κράτη-μέλη ενημερώνουν αυτή τη στιγμή για τις υποχρεωτικές ανακλήσεις και είναι δημόσια τα δεδομένα αυτά. Μόνο 8 κράτη-μέλη έχουν ε, υποχρεώσει σε ανάκληση οχήματα Volkswagen με τους ε, ε, λανθασμένους μετρητές στο Ηνωμένο Βασίλειο έγιναν κάποιες ε, ανακλήσεις ε, που 18 ε, Μαρτίου έχουν φτάσει στο 80% των οχημάτων. Υπάρχουν όμως και κάποια κράτη-μέλη το οποίο στις ανακλήσεις είναι κάτω από το 50%. Εμείς θέλουμε να έχουμε 100% ανακλήσεων για αυτούς τους κινητήρες έτσι όπως είπαμε και στον οδικό χάρτη όπου θέλουμε μέχρι το τέλος του 2019 να έχουμε αντιμετωπίσει το ζήτημα. Εμείς θέλουμε να σας εξασφαλίσουμε πως θα φτάσουμε ε, στο τέλος την υπόθεση της Ελκέτ και τα κράτη-μέλη θα λάβουν όλα τα ε, μέτρα που είναι απαραίτητα για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Θα συνεχίσουμε να κοιτάμε τους ε, εφαρμοστικούς κανόνες για την έγκριση τύπου έτσι ώστε να είναι κατάλληλοι και θα είμαστε πολύ προσεκτικοί με την εφαρμογή των νέων κανόνων και θα προσφέρουμε κάθε στήριξη στα κράτη-μέλη όποτε χρειάζονται για να στήσουν ένα πλαίσιο παρακολούθησης αγοράς. Αλλά θα πρέπει να τονίσουμε πως η παρακολούθηση και η επιβολή είναι θέμα κρατών μελών και θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις ε, οχημάτων που δεν συμμορφώνονται. Καλούμε λοιπόν όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, τα κράτη-μέλη και την αυτοκινητοβιομηχανία να συνεργαστούν και επίση στηριζόμαστε συνεχιζόμενη ε, ε, στήριξη που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνει και αυτή η συζήτηση και θα γίνει η ψηφοφορία την Πέμπτη. Και μπορούμε τώρα ε, να δώσουμε το κύριο, στο λόγο στον κύριο Περβάντη που έχει Γερμανή που θέλει να κάνει μία ε, παρατήρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε την ερώτησή μου γιατί δεν αποκρίθηκε σε όλες τις συστάσεις και τα συμπεράσματα της Επιτροπής, της Ειδικής Επιτροπής. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε τώρα, αλλά θα ήθελε να ζητήσετε εσείς, κυρία Πρόεδρε, γραπτή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν και ή δυνατόν τούτη την εβδομάδα για να λάβουμε δράση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκεμπράντη. Πραγματικά αυτό θα ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη συζήτηση που είναι η έκθεση Μπόνι σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίνου και άλλου ουσιαίους παραμέτρους και την κατάρριση του κανονισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αριθμού 1222 του 2009. Ο κύριο Μπόνι. <clears throat> Κυρίε και κύριοι, κύριε Επιτροπά, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεισηγητές γιατί καταφέραμε από κοινού να καταλήξουμε σε κάποιο γενικό συμβιβασμό παρά το γεγονό ότι η απόψη ήταν αποκλίνουσε σε πρώτη φάση και έτσι λοιπόν αύριο στην ψηφοφορία θα αποφασίσουμε προ τα που θα κινηθούμε. Είναι σημαντικό λοιπόν να ζητήσουμε κοινέ λύσει ρεαλιστικέ. Υλοποιήσε μα. Δυστυχώ δεν μπορέσουμε να τα περάσουμε όλα αυτά εδώ σήμερα, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχουν πραγματικά τεχνικοί έλεγχοι. Γι' αυτό θα θέλαμε να υποχρεώσουμε την Επιτροπή να προβεί σε κάποιες ενέργειες πριν από την επόμενη αναθεώρηση του κανονισμού. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι μιλάμε για το ένα... Το, οι οδικές μεταφορές οφείλονται για το 22% των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τα επίσωτρα λόγω της τριβής. Μιλάμε για μέχρι 10% κατανάλωση καυσίμων των αυτοκινήτων, άρα τα σωστά επίσωτρα θα φροντίσουν προκειμένου τα οχήματα να είναι και πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνα και πιο α, λιγότερο, να, να παράγουν λιγότερο ήχο και να είναι πιο ασφαλή. Και στη τελική ανάλυση οι καταναλωτές λοιπόν θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι καταναλωτές ε, δεν γνωρίζουν αρκετά τα θέματα και της ε, ηχητικής μόλυνσης ε, και της πρόσφυσης σε πάγο και υγρές ε, επιφάνειες. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν καινοτόμα στοιχεία. Επίσης, στο σύστημα λοιπόν επισήμανσης θα περιληφθούν και νέα επίσητρα τα οποία δεν ε, περιλαμβάνουν στον παρελθόν. Και έτσι λοιπόν όλα αυτά θα αποτελέσουν ένα κίνητρο το οποίο θα προωθήσει και την κυκλική οικονομία. Έχουμε συμπεριλάβει λοιπόν και μια υποχρέωση στην αναθεώρηση της οδηγίας προκειμένου να υπάρχει υποχρέωση διεξαγωγής τέτοιων ελέγχων σε ό,τι αφορά και τα μικροπλαστικά Πλέον όλα αυτά περιλαμβάνονται στη σήμανση. Για να είναι σαφή όλα αυτά προς τον καταναλωτή και ο νέος κανονισμός επίσης ε, θα δώσει μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλες αυτές τις ε, προδιαγραφές προκειμένου να υπάρχει τήρηση των σχετικών κανονισμών και κανόνων γιατί υπάρχει υποχρέωση καταχώρηση των επισώτρων σε ειδικέ ε, βάσεις δεδομένων και θα πρέπει να υπάρχουν και σχετικά τιμολόγια τα οποία θα θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα αυτά τα στοιχεία, όλε αυτέ τι προδιαγραφέ, προκειμένου τελικά να υπάρχει δυνατότητα να γίνεται σωστή σύγκριση των προϊόντων βάσει των κριτηρίων. Να υπάρχει λοιπόν διαφάνεια για του καταναλωτέ μεγαλύτερη α, υπευθυνότητα προ το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Κύριε Αρία ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μικαήλ Μπόνη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τον κανονισμό από το 2009 και επομένως Λαμβάνοντας υπόψη και τις ε, τεχνολογικές ε, ε, πρόοδους, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει επικυρωποίηση. αναφερόμαστε λοιπόν και σε αυτήν την τροποποίηση των ετικετών και της επισήμανσης στα πλαίσια της επικυρωποίησης της δέσμης την προηγούμενη χρονιά. Ε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα ελαστικά μπορούν να επηρεάσουν από 5 έως και 10% την κατανάλωση των καυσίμων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να έχει κανείς, να έχει ο καταναλωτής τεκμηριωμένες επιλογές έτσι ώστε να ε, επιλέγει τα ελαστικά σύμφωνα και με την κατανάλωση ενέργειας που συνδέεται με αυτά. Γνωρίζουμε ότι πέραν της εξοικονόμησης εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να έχουμε ε, και ε, σημαντικότατη εξοικονόμηση των ε, επιμολυντικών παραγόντων. Πρέπει να συγχαρώ λοιπόν τον εισηγητή καθώς επίσης και την αρμόδια επιτροπή για την πρόοδο που έχουν κάνει. Πιστεύω ότι μέσω της εκθέσεως αυτής ενδυναμώνεται η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρίως όσον αφορά την ε, πλήρη ε, ε, σήμανση και τις σωστές ετικέτες κυρίως όσον αφορά τις πωλήσει εξ και τις επιγραμμικές. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει και βάση δεδομένων όπου θα ε, αναφέρονται όλα ε, τα ε, στοιχεία αυτά. Η Κομισιόν θεωρεί ότι θα πρέπει επιπλέον να ενδυναμωθεί, ενδυναμωθούν οι κανόνες Απ' την άλλη πλευρά δεν είναι δυνατόν ε, τα επίσωτρα τάξεως F και G, ε, χαμηλότερων δηλαδή τάξεων, ε, δεν μπορούν πλέον να προωθούνται στην εσωτερική αγορά. Θα πρέπει επομένως και οι ίδιες οι βιομηχανίες να κατανοήσουν καλύτερα την κατάσταση και να προσαρμόσουν την παραγωγή τους. Ε, το θέμα της πρόσφυσης επίσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ε, και επομένως η Κομισιόν ε, αναφέρει ότι όταν θα έχει δημιουργηθεί αξιόπιστο τεστ, αξιόπιστο στο τρόπος δοκιμής θα πρέπει να αλλάξουν και τα σημεία συμμόρφωσης. Τρίτον, δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε οποιαδήποτε αποδυνάμωση των, των υποχρεώσεων κυρώσεων στις ε, χώρες μέλη, ούτε οποιαδήποτε αφαίρεση της ετικέτας η οποία θα πρέπει να είναι απολύτως ορατή. Αυτά και τα υπόλοιπα θα μπουν στη διαδικασία συναπόφαση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μαρτάν για ένα λεπτό εξ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Κύριε Μαρτάν παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Μπόνι ε, γιατί είχε πάντοτε ευήκονους. Όμως ε, δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ε, το περιεχόμενο. Πολύ συχνά μιλάμε μόνο για καταναλωτές άνδρες και γυναίκες και όχι για πολίτες άνδρες και γυναίκες. Εγώ θέλω να μιλήσω για πολίτες. Αυτό το θέμα της ετικέτας μπορεί να μην σώσει τον κόσμο, αλλά είναι ένα καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά είπατε και εσείς κύριε, κύριε Επίτροπε, τα μικροπλαστικά ε, αποτελούν ένα τεράστιο ε, ποσοστό ε, ουσιών που στην ουσία βρίσκονται στο περιβάλλον που ζούμε όλοι και που παίζουν τα παιδιά μας. Η έκθεση δεν δείχνει το δρόμο για αυτό το θέμα. Επίσης δεν γίνεται λόγος και για την ποιότητα του πλαστικού που χρησιμοποιείται χρησιμοποιείται. Επίσης, εμείς θέλουμε η χνηλασιμότητα του καουτσούκ που χρησιμοποιείται για τα ελαστικά αυτά και το οποίο δεν θα πρέπει οπωσδήποτε να μολύνει, α πούμε, τον υδροφόρο ορίζοντα. Επόμενο ομιλητή ο κύριος Ράντο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πέτροπα, συνάδελφοι, οι οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν ε, το 25% της ενεργειακής κατανάλωσης και γι' αυτό λοιπόν μιλάμε για πολύ σημαντικό μερίδιο όχι μόνο της ενεργειακής κατανάλωσης, αλλά και της υγείας, της προστασίας από την χορύπανση. Γι' αυτό λοιπόν και είναι τόσο σημαντικό να υπάρξει μια θεώρηση του κανονισμού αυτού και να συμπεριληφθούν και κάποια νέα κίνητρα για ελαστικά υψηλότερης ποιότητας. Επενδύοντας λοιπόν σε καλύτερα ελαστικά, πετυχαίνουμε υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Υποστηρίζω την ιδέα. Να απαγορευτούν τα επίσωτρα χαμηλής ποιότητα και υποστηρίζουμε και την ιδέα να επιτεθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ζουρίνιο, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για τα ελαστικά. Να σας πω πως πάρα πολύ σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια, γιατί είναι ένα προϊόν ευρείας κατανάλωσης και μπορεί να φέρει